cosa che devo chiedere Tutte interrompe la parola. Eh, vediamo, deve essere questo. Sì. Ma il microfono. Pronto, pronto, pronto, pronto. Sì, sì, ci sente. Bene. Okay. Ah, ecco, abbiamo la relatrice presente tra noi. Έχουμε την εισηγήτρια παρούσα, την κυρία Άμαν Ράιτεν, και επειδή η μέρα είναι ιδιαίτερα φορτωμένη, θα πρέπει να τηρήσουμε το χρονοδιάγραμμα με ακρίβεια, παρόλο που έχουμε καθυστερήσει λίγα λεπτά και αμέσως ας ξεκινήσουμε τις ε, εργασίες μας, τις παρεμβάσεις. Όπως βλέπετε από την ημερήσια διάταξη, το πρώτο σημείο αφορά την πρόταση ψηφίσματος για, για την πρόοδο που έχει επιτευχθεί ε, με την Τουρκία. Θα δώσω το λόγο στην εισηγήτρια, την κυρία Ομεν Ρόιτεν, η οποία θα μας παρουσιάσει εν συντομία την έκθεσή της που είναι διαθέσιμη μόνο στα αγγλικά για την ώρα. Υπενθυμίζω επίσης για να δώσω τις πληροφορίες ότι το απόγευμα θα έχουμε τη δυνατότητα να ξανασυζητήσουμε το στάδιο των διαπραγματεύσεων με την Τουρκία με τον Υπουργό Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης της Τουρκίας, τον κύριο Μπάγκης. Έχετε το λόγο εσείς κυρία Όμεν Ρέιτεν. Ναι κύριε Πρόεδρε αξιότιμοι συνάδελφοι, δεν ε, βλέπω να είναι πολύ πρωινοί όλοι οι συνάδελφοι, αλλά εν πάση περιπτώσει εσείς ε, κύριε Πρόεδρε ήρθατε τουλάχιστον και χαίρομαι. Κύριε Πρόεδρε, είναι η πρώτη αυτή η έκθεση προόδου αυτής της ε, νέας θητείας. Γι' αυτό θα ήθελα να σας πω πως το βρίσκω μεγάλης σημασίας για την ε, αξιοπιστία μας το να αναφερθούμε αντικειμενικά και ισορροπημένα στην πρόοδο και προσπάθησα με το γραφείο μου και με την Εύα να κάνω αυτό το πράγμα. Επίσης, συμφωνώ με τις επικοδομητικές παρεμβάσεις ε, των ε, συναδέλφων, αλλά ελπίζω βεβαίως να μην έχουμε πάρα πολλές ε, τροπολογίες, γιατί κατέθεσα νομίζω αυτή την έκθεση ακριβώς γιατί είναι η ισορροπημένη. Το σχέδιο αυτό δεν βασίζεται μόνο στην έκθεση της ε, Κομισιόν, την οποία και ευχαριστώ, αλλά και στις ε, πολλές συνομιλίες που είχα την περασμένη Δευτέρα. Συγχωρείτε τον τελευταίο μήνα και στις Βρυξέλλες και στην ε, Τουρκία και θεωρώ πως ε, ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να επικρίνουμε αλλά και να ενθαρρύνουμε την ε, Τουρκία και φέτος έχουμε τρεις μεγάλες προτεραιότητες στην έκθεση πρώτη. Η ευρεία δημόσια συζήτηση που ξεκίνησε από το καλοκαίρι η τουρκική συζήτηση για τους Κούρδους και τους Αλεβίτες. Θεωρώ πως πρέπει να τους ενθαρρύνουμε και ταυτόχρονα ελπίζω όλοι οι συμμετέχοντες μετά τα πρώτα βήματα που έγιναν τώρα να συνεργαστούν επικοδομητικά για συγκεκριμένη νομοθεσία γιατί βεβαίως καλή στατική αλλά πρέπει να μεταφραστεί και σε νομοθεσία και λέω νομοθεσία αλλά βεβαίως πρέπει να λάβουμε υπόψη όλες τις ευαισθησίες της τουρκικής κοινωνίας Είναι λοιπόν τώρα η ευκαιρία για όλα τα α, μέρη και θα πρέπει να τους υποστηρίξουμε. Δεύτερον, κατόπιν που αποτελεί και την καρδιά της ε, διαδικασίας ε, ένταξης είναι τα πολιτικά κριτήρια. Σε κάποια είχαμε πάρα πολύ λίγη πρόοδο, σε κάποια άλλα βεβαίως είχαμε ε, πρόοδο στην ομοθεσία, αλλά όχι στην εφαρμογή. Να δώσω ένα παράδειγμα όσον αφορά τα δικαιώματα των γυναικών. Έχουμε ένα νομικό πλαίσιο που είναι καλό, αλλά η γάμοι με καταναγκασμό ή τυχόν κακοποίηση των γυναικών δεν τιμωρούνται αρκετά. Αντιλαμβάνομαι ότι πρέπει να αλλάξει η νοοτροπία, αλλά βεβαίως και οι διαδικασίες. Αυτό σημαίνει πως πρέπει να υπάρξει τιμωρία της διαφθοράς των βασανιστήριων όλων αυτών των πραγμάτων. Και βεβαίως όταν μιλάμε για την εφαρμογή αυτό έχει απόλυτη σχέση με την πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη για ριζική μεταρρύθμιση της δικαιοσύνης. Οι πολίτες πρέπει να μπορούν να εμπιστεύονται την αποτελεσματικότητα, την ανεξαρτησία και της δικαιοσύνης και το ότι δεν θα είναι αυτή κομματική και νομίζω πως ε, αυτή είναι μια σωστή στρατηγική που έχει χαραχθεί συνεργασία με τους εταίρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και ελπίζω πραγματικά κυβέρνηση και αντιπολίτευση να συνεργαστούν για να έχουμε συγκεκριμένα αποτελέσματα. Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τώρα να περάσω και σε κάποια πιο συγκεκριμένα σημεία. Κάποια αρνητικά. Τα δικαιώματα των θρησκευτικών μειονοτήτων ε, στα οποία και εγώ και η ομάδα μου δίνουμε μεγάλο βάρος. Είναι ένα εξαιρετικό σημείο για να δώσει ένα καλό μήνυμα η τουρκική πλευρά. Π.χ. για τη θεολογική σχολή της Χάγης, της ε, Χάλκης, Έχουν υποθεί πολλά, αλλά δεν έχει γίνει ακόμα τίποτα. Επίσης, ελευθερία του τύπου. Δεν έχουν γίνει πολλά πράγματα και δεν μιλάμε μόνο για το φορολογικό πρόστιμο που έπεσε σε μια εταιρεία, αλλά και για site τα οποία έκλεισαν. Κατά την άποψή μου, πρέπει να αλλάξουν τα πράγματα βαθιά στην δομή των ΜΜΕ στην Τουρκία. Καθώς μιλάμε για συγκροτήματα επιχειρήσεων που έχουν και ΜΜΕ για να εκπροσωπούν τα συμφέροντά τους έναντι του δημοσίου τομέα. Μετά, δικαιώματα των ε, συνδικάτων. Δεν είναι λεπτομέρειες αυτές. Όταν μιλάμε για το δικαίωμα απεργίας, όταν μιλάμε για τις συλλογικέ διαπραγματεύσεις, πρέπει να έχει σαν όπλο και την απεργία ο εργαζόμενος. Επίσης, διεθνείς συνθήκες του Διεθνούς ε, Οργανισμού Εργασίας δεν έχουν μεταφερθεί στην τουρκική νομοθεσία. Επίσης, για το πρωτόκολλο της ε, Συμφωνίας της Άγκυρας. Πρέπει να εφαρμοστεί και αυτό διαφορετικά θα παραμείνει πάνω από τις διαπραγματεύσεις του Κυπριακού να επικρέμεται. Επίσης, οι παραχωρήσεις προς την ε, Αρμενία και το άνοιγμα των σχέσεων είναι μια ιστορική ευκαιρία που πρέπει πράγματι να την εκμεταλλευτούν. Η υπογραφή της Συμφωνίας Ναμπούκο. Ένα θετικό μήνυμα. Η υπογραφή συμφωνίες, ε, συμφωνιών επανεισδοχής με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σημαντικές. Τελευταία παρατήρηση κύριε Πρόεδρε. Η πόλωση της κοινωνίας και της ε, πολιτικής νομίζω ότι εμποδίζει συχνά τις μεταρρυθμίσεις και είναι κρίμα γιατί μπλοκάρει την χώρα αλλά και την διαδικασία εξυγχρονισμού. Και η διαδικασία εξυγχρονισμού, ή μεταρρυθμίσεις, είναι απολύτως απαραίτητες. Όχι για να το κάνει η Τουρκία για την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά για τους ίδιους Τούρκους πολίτες, γιατί μόνο τότε μπορεί η Τουρκία να γίνει μια σύγχρονη χώρα. Κύριε Πρόεδρε, ε, σας ευχαριστώ για την προσοχή σας και αναμένω τη συνεισφορά των συναδέλφων και ελπίζω να μπορέσουμε να συμφωνήσουμε χωρίς πάρα πολλές ε, τροπολογίες οι οποίες τελικά δεν ξεκαθαρίζουν και τα πράγματα. Τόσο πολύ ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Όμεν Ρόιτεν. Η παρουσίασή σας υπήρξε πλήρης, περιεκτική, εντός των ορίων που είχα στη διάθεσή σας ήταν πολύ ευρία εκάλυψη. Ευχαριστώ. Περνάμε στη συζήτηση. Είμαστε από την αρχή περιορισμένοι χρονικά. Ο πρώτος να μιλήσει είναι ο κύριος Χάουιτ που έχει το λόγο για δύο λεπτά. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να συγχαρώ τη Ρία. Νομίζω την ισορροπημένη έκθεσή της, πολύ καλή βάση και μαζί με το φίλο μου τον Ραϊμόν θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να συνεργαστούμε μαζί της. Στη ψηφοφορία για τη στατική διεύρυνση είδαμε ότι μπορεί να επιτευχθεί συνένεση στο νέο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την Τουρκία. Κάτι πρέπει να προσπαθήσουμε να πετύχουμε στον αφορά τον κύριο Μπροκ και αυτού που ανησυχούν όπω και εκείνο τα κριτήρια τη Κοπενχάγη ε, συμπεριλαμβάνονται στην έκθεση, υπογραμμίζονται και υποστηρίζουμε αυτή την προσέγγιση. Συμφορώ ένθερμα με αυτά που είπε η κυρία Μενράιτεν. Πράγματι χρειάζεται ενότητα, όχι από πλευρά ε, τη κυβερνήση τη Τουρκία, αλλά και όλα τα πολιτικά κόμματα πρέπει να ενωθούν και η κοινωνία τη Τουρκία και θα αναφέρθηκε στι πρόοδου που έχουν επιτευχθεί ε, για το κράτο δικαίου και τα πρόστιμα που επευλήθησαν κατά των ε, μέσων ενημέρωση είναι κάτι που επικρίνει και ζητούμε να ανοίξει το ενεργειακό κεφάλαιο. Για τη δικαστική μεταρρύθμιση θα πρέπει να σημειώσουμε ότι στην έκθεση πρώτη Ευρωπαϊκή Επιτροπή επενούν τα όσα συμβαίνουν στην Τουρκία τον τελευταίο χρόνο στον τομέα αυτό, αλλά επίση υπάρχουν τομεί όπου θα μπορούσαμε να έχουμε περισσότερε λεπτομέρειε. Θα ήθελα να συνεργαστούμε με τη ΡΙΑ όσον αφορά αυτό το θέμα, όσον αφορά επίση το πώ ποια θα είναι η μορφή τη εκθέσεώ μα, να πω ότι η έκθεση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή κοιτάει το παρελθόν, προσμετρά την πρόοδο, ελπίζω αυτό το ψήφισμα να κοιτάει προ το μέλλον και να δώσει προκλήσει στου φίλου μα, του Τούρκου και συμμάχου, ε, για να δουν τι προόδοι μπορούν να επιτευχθούν. Διότι υπάρχει άνευ προηγουμένο παράθυρο ευκαιριών στην εσωτερική πολιτική τη Τουρκία, όπου μπορούν να κάνουν ε, περισσότερε μεταρρυθμίσει οι Τούρκοι. Δεύτερον, α μην κοιτάμε κατά πρόσωπο τα πραγματικά επιτεύγματα. Αυτό που έγινε με την Αρμενία όσον αφορά το κουρδικό, εκεί υπάρχουν ακόμα πολλά προβλήματα σχετικά με τα ζητήματα, αλλά έγιναν κάποια άλματα τα οποία ήταν απροσδόκητα, δεν τα αναμέναμε και πρέπει να τους δώσουμε ε, βαθμούς αν θέλετε για αυτά τα επιτεύγματα που επέτυχαν σε αυτούς τους δύο τομείς. Ευχαριστώ κύριε Χάουιτ. Για δύο λεπτά ο κύριος Λάμστορφ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ την κυρία Ομεν Πράγματι έθεσε μια πάρα πολύ καλή βάση για την εργασία μας, ξεκάθαρη και ισορροπημένη. Οπωσδήποτε σε κάποια ζητήματα θα τα συζητήσουμε περισσότερα, π.χ. αυτό που έχει ιδιαίτερη σημασία για την ομάδα μου, η ελευθερία της ε, έκφρασης. Θέλουμε περισσότερη πρόοδο. Εδώ πέρα νομίζω πως ε, έχουμε μια κάπως ασυνήθιστη και μη διπλωματική γλώσσα όσον αφορά αυτές τις ε, ανησυχίες που εκφράζει η Κομισιόν. Πρέπει να το σκεφτούμε. Είναι ένα παράδοξο. Απ' τη μία υπάρχουν ανοιχτές συζητήσει για πάρα πολλά κρίσιμα ζητήματα, απ' την άλλη δεν υπάρχει επαρκές νομικό πλαίσιο. Και ισχύει το αντίστροφο για την ε, θρησκευτική ελευθερία βεβαίως δεν είναι τόσο σημαντικό αυτό για εμάς τους φιλελεύθερους όσο για το ΕΛΚΑ αλλά παραμένει η θεμελιώδης ε, ελευθερία. Επίσης ε, πρέπει να γίνει μια διάκριση μεταξύ διπλωματίας και δημοκρατίας. Πράγματι έχετε δίκιο, είναι θετικό το ότι επιτυγχάνεται πρόοδος με την ε, Αρμενία, αλλά σημαντική είναι η δημοκρατική εξέλιξη εντός της χώρας. Αυτό είναι το θέμα μας και για το ζήτημα της διπλωματίας να κάνω δύο ακόμα παρατηρήσεις. Πρώτον, ναι, πολύ καλή υπόθεση με την Αρμενία, η πρόοδος αυτή. Εγώ θα ήθελα και κάποια ανάλογη πρόοδο στην εφαρμογή του πρωτοκόλλου της Άγκυρας που δυστυχώς δεν έχει συμβεί και ακριβώς ε, με ανισχύει αυτό από διπλωματική σκοπιά όταν ο πρόεδρος ε, Αχμαντίνετζάντ ε, περιγράφεται από τον Τούρκο πρόεδρο ως ε, φίλος ε, και το ίδιο ε, υποδέχονται και τον πρόεδρο του Σουδάν ο οποίος αναζητείται για εγκλήματα πολέμου. Δεν ξέρω ποιες είναι οι προθέσεις της Τουρκία, Τουρκίας στην περιοχή. Νομίζω όμως πως θα μπορέσουμε να εργαστούμε με βάση αυτό το σχέδιο έκθεσης. Ευχαριστώ. Βάιγκελ για δύο λεπτά. Ο κύριος Βάιγκελ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Το τραπέζι μπροστά μας έχουμε μια έξοχη έκθεση. Είναι αναλυτική έκθεση και χρησιμοποιεί διπλωματική διατύπωση. Είμαστε πολιτικοί. Μας ενδιαφέρει πρωταρχικά η πολιτική αξιολόγηση. Πιστεύω λοιπόν ότι στην πρόταση ψηφίσματος υπάρχει καλή ισορροπία μεταξύ ενός πραγματικού γεγονότος, δηλαδή ότι η Τουρκία είναι μια περίπλοκη πολυπολιτισμική κοινωνία όπου έχουμε παράδοση και η εναρμόνιση μακροπρόθεσμα είναι κάτι που απαιτείται στη χώρα αυτή. Από πλευράς Ευρωπαίων πολιτικών έχουν γίνει μία-δύο λυπηρές αξιολογήσεις έναντι της Τουρκίας και η Τουρκία έχει παρατηρήσει αυτές τις αξιολογήσεις. Πιστεύω ότι θα πρέπει να αποφεύγουμε τέτοιου είδους αξιολογήσεις και χαίρομαι που αυτές οι εκτιμήσεις δεν τις βρίσκουμε σε αυτή την έκθεση. Όπως και ο κύριος Λάμπστορφ και εγώ Λέω ότι πρέπει να είμαστε ευαίσθητοι απέναντι στι ελευθερίε. Τι θεωρούμε δεδομένε τι ελευθερίε στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά το συμβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δικαιωμάτων τα δικαιώματα των μειονοτήτων, την ελευθεροτυπία, την ισότητα ανδρών, γυναικών κλπ. Και κάτι άλλο το οποίο αναφέρεται στην έκθεση. Η Τουρκία είναι εταίρος μας στον κόσμο, σε ειρηνευτικές επιχειρήσεις και σε άλλες δραστηριότητες όπου συνεργαζόμαστε και στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δηλαδή Ευρωπαϊκή Ένωση με την Τουρκία και τον ΝΑΤΟ. Μάωρο, κύριος Μάωρο έχει το λόγο για δύο λεπτά. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Λαμβάνοντας υπόψη ότι ο χρόνος είναι πολύ περιορισμένος, θα ήθελα να επικεντρωθώ επί της μίας πτυχής στα πλαίσια τη έξοχη δουλειά που έκανε η κυρία Όμεν Ρόιτεν. Δηλαδή, θα ήθελα να αναφερθώ στην αξιολόγηση τη περιφερειακή πολιτική τη τουρκική κυβερνήσεω. Εκμεταλλεύεται η κυβέρνηση ότι υπάρχει μεγάλη σταθερότητα εδώ και πολλά χρόνια και αναπτύσσει αυτή την πολιτική. Επεξηγούμε, εξηγούμε. Από τη μία πλευρά έχουμε μια Τουρκία η οποία χτυπά τις πόρτες της Ευρώπης και κάνει μεγάλη πρόοδο για να πετύχει αυτό το αποτέλεσμα. Από την άλλη όμως έχουμε μια Τουρκία η οποία με αναφορά την πολιτική της έναντι των Βαλκανίων, της Κίνας, του τορκόφωνων πληθυσμών Μεσοποταμίας και Σιβηρίας δείχνει ότι θέλει να είναι χώρα που ε, έχει ηγετική θέση στην ε, κεντρο Ασία. Όπως είπε και ο κύριος Λάντορφ, οι σχέσεις με χώρες όπως είναι το Ιράν, το Ιράκ και η Συρία, Τουρκία με αυτές τις χώρες, θα πρέπει να μας δημιουργεί ερωτηματικά όσον αφορά τη συμβατότητα της ανάπτυξης αυτών των στρατηγικών με τις πιο γενικές πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, το σύνολό της. Πιστεύω ότι θα πρέπει να το προσέξουμε αυτό, θα πρέπει να αξιολογήσουμε αυτές τις κινήσεις και να τις πλαισιώσουμε στις παρατηρήσεις όσον αφορά την πρόοδο της Τουρκίας προς την προσχώρηση στην Ευρώπη, να βλέπουμε τι κάνει στον κόσμο η Τουρκία. Διότι ε, προφανώς οι συνέπειες δεν περιορίζονται απλώς σε φιλικούς τόνους στις σχέσεις με τον Αχμαντινετζάτ και με άλλους, αλλά μπορεί να καθορίζονται και στατηγικά οι τοποθετήσεις. Και μπορεί να έχουν συνέπειες αυτές οι κινήσεις της Τουρκίας που ε, δεν μπορούμε να τι καθορίσουμε. Είναι μια θωμανική προσέγγιση, θα έλεγα. Ο κύριος Μάουρο, τελείωσε ο κύριος Άτκιν έχει το λόγο για δύο λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να επιμείνω σε μία πτυχή αυτής της εξαιρετικής έκθεσης της ΡΙΑ. Χθες ε, συνάντησα τον ε, Ελληνοκύπριο δήμαρχο της Αμοχώστου με κάποιους συναδέλφους του και παρόλο που υπήρχε κάποια αφησιμία εκ μέρους μου για την προσχώρηση της Τουρκίας. Επαφωτερίζουσα είναι η στάση μου. Δεν έχω πιστεί ούτε προ τη μία ούτε προ την άλλη κατεύθυνση. Αλλά νομίζω ότι η θέση τη Τουρκία απέναντι στην Κύπρο και η αδιαλαξία είναι χαρακτηριστική. Όχι μόνο στο ε, στο νησί, αλλά και με τους Έλληνες και Κυπρίους συναδέλφους. Και νομίζω ότι θα πρέπει εμείς να καταστήσουμε απόλυτα σαφές ότι μας ενοχλεί και μας δυσταριστεί ιδιαίτερα ότι η κατάσταση αυτή έχει αποτελματωθεί. Γίνονται κάποιες μικροκινήσεις, αλλά εν γέννη η κατάσταση είναι αποτελματωμένη. Γνωρίζω από προσωπική μου εμπειρία και γνωρίζοντας και τους Ελληνοκύπριους και τους Τουρκοκύπριους, βάζουν πρώτα την Κύπρο και δεύτερη στην Ελλάδα και την Τουρκία. Και εσωτερικά δεν έχουν και προβλήματα ιδιαίτερα, γιατί ο Δήμαρχος της Αμοχώστα είπε ότι η σχέση με τους ε, Τουρκοκυπρίους γενικώ είναι καλές. Αλλά πρέπει να μας κάνει μια χειρονομία η Τουρκία. Και δεν ξέρω αν κατά τη συζήτηση της έκθεσης μπορούμε να υποβάλουμε μια τροπολογία για να ενισχύσουμε και να κάνουμε πιο επίμονη την έκκλησή μας προς την Τουρκία να μην είναι πια αδιάλακτη, να αναγνωρίσει ότι αυτό είναι κρίσιμο θέμα και η Λευκοσία είναι η μόνη διχασμένη, διχοτομημένη πόλη στην Ευρώπη. Δεν μπορούμε να παραδεχόμαστε μια τέτοια κατάσταση, να την ανεχόμαστε. Θα πρέπει να επιληθεί αυτό το θέμα. Δεν μπορεί να μένει ατέρμονα έτσι αμφίσιμο. Και επίσης ε, θα μπορούσαμε να συντάξουμε και μια τροπολογία κατά τη γνώμη μου, κάνοντας πιο επίμονη αυτή την έκκληση. Ευχαριστώ κύριε Άτκινς. Ευχαριστώ κυρία Φλότρε. έχει το λόγο η πρόεδρος της Επιτροπής Ευρωπαϊκή Ένωση Τουρκία. Ευχαριστώ. Ήθιστε στο Κοινοβούλιο να δίνουμε πρώτα το λόγο στους ε, συντονιστές ή στους προέδρους των ε, κοινοβουλευτικών αντιπροσωπιών. Η έκθεση της κυρίας Ομενρόιτεν είναι εξαιρετική βάση συζήτησης ε, για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και για την Επιτροπή και την ευχαριστώ θερμά για τις προσπάθειές της. Η έκθεση λέει ήδη από τις πρώτες παραγράφους αλλά και στα συμπεράσματα ότι υπήρξαν εξελίξεις θετικές και ενθαρρύνσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς τις τουρκικές αρχές αλλά και την τουρκική κοινωνία. Νομίζω ότι αυτές οι θετικές εξελίξεις είναι πραγματικά ψυχοτικές. Σε ό,τι αφορά τα προτινόμενα κριτήρια της Κοπεχάγης, καλό θα ήταν να γίνει μια αναδιοργάνωση γιατί οι εκθέσεις μας σχολιάζονται εκτενώς και στον τουρκικό τύπο. Οπότε καλό θα είναι να είναι χρήσιμες από αυτή την άποψη και να ενισχύουν τους διάφορους φορείς, τα πολιτικά κινήματα, τα συνδικαλιστικά κινήματα που δίνουν μάχη για περισσότερη δημοκρατία και σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών στην Τουρκία. Οπότε εύστοχο και σκόπιμο θα ήταν να δώσουμε στους διάφορους άξονες των θεμελιωδών ελευθεριών καλύτερη διάσταση. Για παράδειγμα, δεν είναι συνετό κατά τη γνώμη μου να έχουμε πέντε παραγράφους για τις θρησκευτικέ μειονότητες, ενώ το ουσιώδες ζήτημα της συνδικαλιστικής ελευθερίας, το θεμελιώδες αυτό δικαίωμα, αναφέρεται μόνο προς το τέλος των κριτηρίων της Κοπεχάγης και σε μία μόνη παράγραφο. Ενώ αφορά τι συλλογικέ δράσει, το δικαίωμα τη απεργία, τη συνδικαλιστική ελευθερία, αυτέ είναι οι προποθέσει για το άνοιγμα ενό κεφαλαίου και νομίζω ότι αξίζει μια καλύτερη θέση, ακόμη και η ελευθερία έκφραση. Γιατί γίνεται τέτοια διαφοροποιημένη μεταχείριση τόσο θεμελιωδών ελευθεριών όπως η θρησκευτική, η ανεξιθρησκεία μάλλον, η συνδικαλιστική ελευθερία, η ελευθερία έκφραση. Θα πρέπει να αποκαταστήσω μια ισορροπία μεταξύ των ελευθεριών αυτών. Τώρα στα πλαίσια της συζήτησης Έχετε εξαντλήσει το χρόνο σας παρακαλώ κυρία μου, ολοκληρώστε. Ακούστε, συζήτηση κάνουμε, η πρώτη συζήτηση επί τη βάση ενός σχεδίου έκθεσης. Ναι, αλλά πρέπει να σεβαστούμε το χρόνο μας, λέει ο Πρόεδρος. Νομίζω ότι δικαιούμαι να υποβάλω και τις δικές μου απόψεις εδώ. Και επιτρέψτε μου να ολοκληρώσω. Δεν ολοκλήρωσα. Χρειαζόμαστε και μία παράγραφο για το δικαίωμα των μεταναστών και των ετούντων άσυλο. Μας λείπει μία τέτοια παράγραφος. Ξέρετε ότι το Συμβούλιο της Ευρώπης ε, έχει καταρτήσει εκθέσεις για το θέμα αυτό. Πολύ μεστές. Και μια και έχουμε διαπραγματεύσεις για μια συμφωνία επανεισδοχής, μια τέτοια παράγραφος είναι ουσιώδης για την έκθεση αυτή. Ολοκληρώνω κύριε Πρόεδρε. Μια στιγμή, μια στιγμή τελειώνω. Χρειαζόμαστε ρητή μνήα της προοπτικής της ένταξης. γιατί χθες μιλήσαμε για το ενισχυμένο καθεστώς του Μαρόκου και νομίζω ότι οι προσπάθειες, η παρακολούθηση και ο έλεγχος που απαιτείται από την Τουρκία θα πρέπει να στηριχθούν σε μια πραγματική γνήσια ενταξιακή προοπτική της Τουρκίας. Οι δεμή θα μας επικρίνουν και δικαίως ότι χρησιμοποιούμε δύο μέτρα και δύο σταθμά στις εταιρικές μας σχέσεις, γιατί το ενισχυμένο καθεστώς είναι αρκετά δεσμευτικό. Σας ευχαριστώ για την υπομονή σας. Σας ευχαριστώ. Ε, τελευταία φορά όμως. Ε, γνωρίζετε την υπομονή μου τελευταία φορά. Χάτζη Γεωργίου, δύο λεπτά. Να συγχαρώ και εγώ καταρχήν την κυρία Όμεν για την έκθεσή της, η οποία είναι πράγματι εμπολής αντικειμενική σειρά στοιχείων τη έκθεση για την Τουρκία αντικατοπτρίζουν την πραγματικότητα, είναι θετικέ επισημάνσει για σειρά αρνητικών δεδομένων και πρέπει το Κοινοβούλιο μα να συνεχίσει να τα υποδεικνύει. Δυστυχώ, οι Τούρκοι εργαζόμενοι δεν έχουν βασικά δικαιώματα κατοχυρωμένα από συμβάσει και τον Διεθνή Οργανισμό Εργασία, όπω το δικαίωμα στην απεργία, χωρί εκφοβισμού και φυλακίσει. Ο στρατό, αγαπητοί συνάδελφοι, δεν είναι σε πλήρη πολιτικό έλεγχο. Ακόμα ορίζει ζητήματα εξωτερική πολιτική η ομαλοποίηση των σχέσεων με Αρμενία δεν πρέπει να αποτελέσει επικοινωνιακό τρίκ, αφού θα πρέπει να υλοποιηθούν αποφάσεις και είναι εδώ που θα κριθούν όλοι. Δεν είναι αλήθεια ότι το ΠΚΚ κατεφεύγει σε όποιες αιματοχυσίες, ιδιαίτερα τον τελευταίο χρόνο. Χαιρετίζομαι προσπάθειες για αποδοχή των δικαιωμάτων των Κούρδων, αλλά αυτές πρέπει να υπερβούν το πρώτο βήμα και να περάσουν σε στάδιο που δεν τους καταδιώκει, με απόσυρση αντιδημοκρατικών και κατασταλτικών μέτρων θα πρέπει οι νομικές δομές του τουρκικού κράτους να γίνουν τέτοιες που να ενσωματώνουν και να προεσπίζονται το δίκαιο. Για το Κυπριακό, αγαπητοί συνάδελφοι, τι ζητούμε. Η Τουρκία να κάνει ό,τι έχει υπογράψει. Έχει υπογράψει απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση ότι θα ανοίξει τα αεροδρόμια και τα λιμάνια της στην Κύπρο. Δεν το έχει κάνει. Έχει υπογράψει ότι θα ομαλοποιήσει τη σχέση της με την Κύπρο. Δεν το έχει κάνει και έχει υπογράψει ότι θα βοηθήσει στην επίλυση του Κυπριακού. Να μην μείνουμε στα λόγια. Ένα σπρόξιμο προ την Τουρκία είναι αναγκαίο και χρήσιμο για να επιληθεί ένα πρόβλημα που ταλανίζει όλου. Τέλο, δεν πρέπει να αφαιθεί να νοηθεί ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση επιβραβεύει την Τουρκία για τη στάση τη ανοίγοντα το κεφάλαιο τη ενέργεια επειδή έχει συμφωνίε με κάποια κράτη-μέλη. Τι γίνεται με τα άλλα κράτη στα οποία η Τουρκία παρεμποδίζει την άσκηση των κυριαρχικών του δικαιωμάτων πράξη που σχετίζεται με το υποσυζήτηση κεφάλαιο. Κλείνω. Υπάρχουν θετικέ εξελίξει στην Τουρκία, συνάδελφοι. Αλίμονο αν εμεί δεν τη βλέπουμε. Εμεί ιδιαίτερα οι Κύπροι τι παρακολουθούμε και τι βλέπουμε και σα καλούμε να πάρετε όχι από τι ευαισθησίε μα, αλλά από την εμπειρία μα σαν γείτονη χώρα αυτού του κράτου που αιτείται την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Κόβατσεφ για δύο λεπτά παρακαλώ. Κύριος Κόβατσεφ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Όμεν Ρόιτεν. Είναι πολύ ισορροπημένη, καλή η έκθεσή της. Δεχόμαστε και αναγνωρίζουμε την πρόοδο της Τουρκίας σε κάποιους τομείς όπως είναι ο οικονομικός τομέας, ο τομέας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων έχει επιτευχθεί η πρόοδο στι σχέσει με τι γειτονικέ χώρε. Να σα επιστήσω την προσοχή σε δύο πτυχέ. Γνωρίζετε ότι υπάρχουν κάποια προβλήματα μεταξύ Τουρκίας και Βουλγαρίας. Υπάρχει παλιά συμφωνία μεταξύ Τουρκίας και Βουλγαρίας που δημιουργεί κάποια προβλήματα και υπάρχει πρόβλημα με τους βούλγαρους πρόσφυγες. Θα ήθελα η κυρία Ρόιτεν να τα συμπεριλάβει αυτά στην έκθεσή της. Κατά την άποψή μου, είναι ανησυχητικό όταν ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών που επισκέπτεται κάποιες βαλκανικές χώρες και πάει, παραδείγματος χάρη στο Σεράγεβο, λέει ότι η Οθωμανική παρουσία στα Βαλκάνια ήταν θετικό στοιχείο, θετικό μήνυμα και όταν ένας υπουργός εξωτερικών δηλώνει ότι η Τουρκία προστάτευε ένα μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού των Βαλκανίων. Αυτό είναι κάτι που δεν ισχύει. Δεν πιστεύω ότι ένας Τούρκος υπουργό έπρεπε να λέγει αυτά τα πράγματα όταν χτυπάει τις πόρτες της Ευρώπης η Τουρκία. Σας ευχαριστώ. Ο κ. Μαυρονικόλας για δύο λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να αναφέρω στο σημερινό ψήφισμα ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό να αναφερθούμε στις σχέσεις καλής γειτονίας της Τουρκίας με τις χώρες που την περιβάλλουν. Πιστεύω το σημερινό ψήφισμα είναι αρκούντος ικανοποιητικό και ισορροπημένο. Θα ήθελα όμως να επισημαίνω ότι κάποιες από τις ενέργειες και πράξεις της Τουρκίας εμπεριέχουν τον κίνδυνο να αποτελούν απλά ενέργειες καλής θέλησης. Τέτοιες ενέργειες έχουν γίνει με το Κουρδικό και με την Αρμενία, αλλά δεν βλέπουμε οποιασδήποτε ουσιαστικές αλλαγές στις ε, σχέσεις της Τουρκίας με τις γειτονικές χώρες. Στο Κυπριακό θα ήθελα να αναφέρω ότι θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε τον πρώτη των κίνδυνων που αντιμετωπίζει σήμερα η Κύπρος και ο κίνδυνος αυτός είναι ο επικισμός από την Τουρκία. Πιστεύω ότι η αγαπητή συνάδελφος θα μπορούσε με δύο-τρεις λέξεις να συμπεριλάβει την ανάγκη να σταματήσει ο επικισμός στην Κύπρο. Επίσης, θα πρέπει να ισχυριστούμε με κάθε ειλικρίνεια ότι πραγματικά δεν έχει κάνει απολύτως τίποτε η Τουρκία σε σχέση με την, με την Κύπρο. Ούτε ένα από τα θέματα τα οποία έχει υπογράψει. Αναφέρθηκε προηγούμενο ο συνάδελφος στη συζήτησή του με τον Δήμαρχο Αμοχώστου. Έχουμε μία πόλη φάντασμα στην Κύπρο. Κύριε Πρόεδρε, η πόλη φάντασμα αυτή ονομάζεται Αμόχωστος και είναι πόλη φάντασμα εδώ και από το 1974 Επίσης θα μπορούσε στο κείμενο να γραφτεί ότι πρέπει άμεσα να εφαρμοστεί το πρωτόκολλο της Άγκυρας και τελειώνοντας θα ήθελα να δηλώσω και εγώ ότι το άνοιγμα του κεφαλαίου της ενέργειας με βρίσκει σε αυτή τη φάση τουλάχιστον όπως προχωρούμε και όπως βλέπουμε αντικειμενικά τα γεγονότα εντελώς αντίθετο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ κύριε Μαυρονικόλα. Μπότσκουρ για δύο λεπτά. Κυρία Μπότσκουρ. Σας ευχαριστώ. Θα ήθελα καταρχήν να ευχαριστήσω θερμά την κυρία Όμεν Ρόιτεν, γιατί η έκθεσή της, το σχέδιο έκθεσής της είναι μια πολύ σωστή βάση εργασίας. Είναι ισορροπημένη όπως κάθε πόνημα της κυρίας Όμεν Ρόιτεν. Εγώ θα ήθελα να πω δύο λόγια για την ισότητα των ευκαιριών μιλάμε για τα δικαιώματα των ομοφιλοφίλων. Ωραία. Αλλά να μιλήσουμε και τα δικαιώματα των ε, φιλομεταβατικών. Transgender. Υπάρχουν κάποια, κάποιες θετικές εξελίξεις για την Αρμενία για παράδειγμα. Η κατάσταση με τους Κούρδους έχει βελτιωθεί και στο Κοινοβούλιο το επισημαίνουμε αυτό χρόνια ολόκληρα. Είναι σαφές ότι υπάρχουν κάποιες δυσκολίες, αλλά οι τουρκικές αρχές έχουν επιδείξει θάρρος και τόλμη και θα πρέπει να τις ε, υποστηρίξουμε. Σε ό,τι αφορά τώρα την ανεξιθρησκεία, είναι πολύ σημαντικό αυτό το δικαίωμα, αυτή η ελευθερία και θα πρέπει τα δικαιώματα της χριστιανικής, ε, των χριστιανικών θρησκευτικών ε, μειονοτήτων να υπερασπίζονται, να τη χάνουν υπεράσπιση μάλλον, αλλά όταν μιλούμε για ανεξιθρησκεία, μην ξεχνάτε ότι υπάρχουν και άλλες θρησκευτικέ ενότητες, όχι μόνο η χριστιανική. Η ανεξιθρησκεία ε, θα πρέπει να ισχύει σε ολόκληρη την Ευρώπη και για όλες τις θρησκευτικέ μειονότητες. Ο Ευρωπαίος Επίτροπος ε, για τα θέματα διεύρυνσης έκρινε ότι οι διμερείς σχέσεις μεταξύ Σλοβενίας και Κροατίας θα πρέπει να βελτιωθούν χάρη στην διαπραγμάτευση. Ίσως αυτό το θέμα το δημερώσει, ίσως θα πρέπει να το αναφέρουμε και στην έκθεση. Δεν ξέρω τι γνώμη έχει η κυρία Μποσκούρτη. Κυρία Κοπάκια, δύο λεπτά. Ε, πρώτα απ' όλα θέλω και εγώ να συγχαρώ την εισηγήτρια, η οποία για μία ακόμα χρονιά παρουσίασε ένα πάρα πολύ ισορροπημένο κείμενο. Δύο μόνο σημεία θέλω να επισημάνω στην οποία, στα οποία θα ήθελα τα σχόλιά της το ένα αφορά το πρωτόκολλο της Άγκυρας. Στην περσινή της έκθεση είχε ζητήσει μια καταληκτική ημερομηνία για, την εφαρμογή και επικύρωση και εφαρμογή του πρωτοκόλλου αυτού. στο φετινό κείμενο όχι μόνο δεν υπάρχει αυτή η καταληκτική ημερομηνία, αλλά προτείνει και το άνοιγμα του κεφαλαίου της ενέργειας. Και ε, ερωτώ πώς είναι δυνατόν με μια χώρα που διαπραγματεύεται με τις 26 από τις 27 χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης να ζητάμε να ανοίξει ένα ακόμα κεφάλαιο. δεύτερη ερώτηση, το θέμα δύο μικρών νησιών, τη Σύμβρου και τη Στενέδου. Στην περσινή της έκθεση είχε αναφορά, πολύ σημαντική κατά τη γνώμη μου, στην ανάγκη διατήρησης του πολυεθνικού χαρακτήρα των δύο νησιών. Στη φετινή έκθεση δεν υπάρχει αυτή η αναφορά και θα ήθελα να ρωτήσω γιατί. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ κυρία Κοπά για δύο λεπτά. Ο κύριος Τάνοκ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα είμαι πάρα πολύ σύντομος. Δεν θα χρειαστώ καν δύο λεπτά. Ήθελα να συγχαρώ εκ μέρους της ομάδας μου, της ομάδας CCR, την κυρία Όμεν Ρόιτερ... που εξεπώνησε φέτος μια ιδιαίτερα σύντομη και πλήρη έκθεση, που είναι εξαιρετικά ισορροπημένη και καλύπτει όλους τους βασικούς ε, τομείς. Θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή της Επιτροπής στην παράγραφο 32, όπου εκεί νομίζω ότι ίσως να χρειάζεται κάποια μικρή ενίσχυση του μηνύματος. Είναι απογοητευτικό, πιστεύω, δοθέντος του πολιτικού κεφαλαίου και ενέργειας που καταναλώθηκαν για τη λήξη του εμπάργκο με την Αρμενία και ε, ε, ο πρόεδρος Σαρκοζή αγνώρισε και τη διασπορά της Αρμενίας για να γίνει αυτό και υπεγράφει το επόμενο συνεννόησης και τα πρωτόκολλα και την επόμενη μέρα ο Πρωθυπουργό της Τουρκίας είπε ότι παρά τα όσα έγιναν δεν ήταν έτοιμος να προωθήσει το έγγραφο αυτό μέσα στην τουρκική εθνοσυνέλευση που έχει πολύ μεγάλη πλειοψηφία και θα μπορούσε να το κάνει εύκολα εκτός εάν είχε επιληθεί το πρόβλημα του Ναγκόρνο Καραμπάχ. Και αυτό είναι παιχνίδι στα χέρια των εθνικιστικών δυνάμεων στον Πακού και στο Αζερμπαϊτζάν ε, στους οποίους ασκούνταν πίεση να ε, συμβιβαστούν και μπαίνουν χρήματα στην κυβέρνηση της Αζερία και έχουμε τώρα πολεμοχαρεί δηλώσεις που γίνονται ότι επιφυλάσσουν του δικαιώματο να ξανακατακτήσουν διαδυνάμες στον Αγκόρνο Καραμπάχ. Θα πρέπει χωρί να θέσουμε προποθέσει να είμαστε πιο στεναροί στη διατύπωσή μα. Να πούμε, εκφράζουμε τη λύπη μα διότι η κυβέρνηση τη Τουρκία υπαναχώρησε από τι συμφωνίε. Τέλο πάντων, τούτου λεχθέντο, όλε οι άλλε πτυχέ εκθέσεω είναι άκρο ικανοποιητικέ, καλύπτονται όλα τα θέματα από τις δολοφονίες γυναικών μέχρι θρησκευτικέ μειονότητες, τους χριστιανούς, τους ε, Σύριους, τους, ε, τον κλήρο των Ορθοδόξων, Ελληνοορθοδόξων Πολύ καλά τα κατάφερες Ρία, είναι μια έξοχη έκθεση. Ευχαριστώ κύριε Τάνοκ. Κλείνουμε τις παρεμβάσει με τα δύο λεπτά του κυρίου Παπαδόπουλου. Κύριε Πρόεδρε. Κύριε Είναι διπλωματική όντω η έκθεση τη κυρία Χόμεν. Επισημαίνει πρόοδο σε κάποια θέματα, όμω υπάρχουν αρκετά προβλήματα τα οποία η Τουρκία πρέπει να δει χρειάζεται άσκηση πιέσεων επιτάχυση μεταρρυθμίσεων εφαρμογή της νομοθεσίας υλοποίηση δεσμεύσεων και όχι επικοινωνιακή πολιτική. Υπάρχει πρόβλημα στα θέματα των γυναικών, στην ισότητα των φύλων, στην ελευθερία του τύπου, στο ρόλο που διαδραματίζει ο στρατός στην Άγκυρα. Τα ανοίγματα στους Κούρδους και στους Αρμενίους μας βρίσκουν σύμφωνους, όμως δεν πρέπει να είναι επικοινωνιακά τεχνάσματα. Στο Κυπριακό η Άγκυρα δεσμεύτηκε αλλά δεν υλοποίησε το πρωτόκολλο της Άγκυρας, δεν ομαλοποίησε τις σχέσεις της με την Κύπρο, παραμένει αδιάλακτη στο Κυπριακό, διατηρεί διαρκώς και ενισχύει την παρουσία τουρκικού στρατού στο 37% των κυπριακών εδαφών που είναι ευρωπαϊκά εδάφη. Συνεχίζει τον επικισμό των κατεχομένων, το σφετερισμό των περιουσιών των Ελληνοκυπρίων στα κατεχόμενα. Παρεμποδίζει με δικά τη πλοία τι έρευνε τη Κύπρου στην νότια οικονομική ζώνη για πετρέλαιο δεν άνοιξε την πόλη της αμοχώς του όπως λένε τα ψηφίσματα του οργανισμού ηνωμένων εθνών. εξακολουθεί να παραβιάζει τα δικαιώματα των συγγενών των αγνωμένων και εμάς των προσφύγων. η τουρκία πρέπει να πιεστεί. διαφωνούμε να ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο για το περιβάλλον ή την ενέργεια και ας μην θοπεύουμε την τουρκία είναι σημαντικό να ασκηθούν κυρώσει τον Δεκέμβρη. Συγχαίρω την κυρία Νόουμε και ελπίζω αρκετά από αυτά που συμβαίνουν στην Κύπρο να ενσωματωθούν στην έκθεσή τη, στην πρόταση ψηφίσματο. Σας ευχαριστώ. Κυρία Παπαδοπούλου, έχουμε τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Όχι πάνω από ένα πεντάλεπτο παρακαλώ. Ευχαριστώ, πρόεδρε. Δεν θα χρειαστώ καν ολόκληρο πεντάλεπτο για να σας εκθέσω τη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έκθεση Omen Reuters. Κατά τη γνώμη είναι άκρος ισορροπημένη και αντικατοπτρίζει με σαφή τρόπο την κατάσταση στην Τουρκία. Κάνει έναν σωστό και ακριβή απολογισμό των τελευταίων χρόνων και δίνει και συγκεκριμένες προοπτικές για το τι θα πρέπει να γίνει στην Τουρκία προκειμένου να σημειωθεί πρόοδος ε, στους διάφορους τομείς που πραγματεύεται η έκθεση. Ίσως ε, θα μπορούσαν να γίνουν κάποιες σκέψεις για την ανισορροπία που υπάρχει σε ό,τι αφορά την αντιμετώπιση κάποιων ελευθεριών ε, δίνεται μεγαλύτερο βάρος σε ορισμένες από τις άλλες όπως επισήμανε και η κυρία Φλότρ. Εκεί ίσως θα μπορούσε να γίνει μια επανισορρόπηση μεταξύ των διαφόρων θεμελιωδών ελευθεριών. Κάποιες θεμελιώδεις ε, ελευθερίες, ε, έχουν τη θέση στο κείμενο και αξίζουν να είναι εκεί όπως και άλλες. Ρία, σας ε, διαβίβασα τις απόψεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την αιτιολογική σκέψη που αφορά την έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Παρακαλώ ε, εξετάστε τις παρατηρήσεις μας, γιατί εφόσον αναφέρεστε στην έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα να πείτε ότι καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι ήταν περιορισμένη η πρόοδος των προηγούμενων ετών, μάλλον δεν είναι πιστή μεταφορά των συμπερασμάτων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μια τέτοια δήλωση. Παρ' όλα αυτά η έκθεση σας είναι εξαιρετική και σας συγχαίρουμε θερμά. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κύριε Φιλόρη. Όπως πάντα κλείνει τη συζήτηση με την παρέμβασή της η συγγήτρια. Η κυρία Ομενρόιτεν έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να επανέλθω σε κάποιες παρατηρήσεις που, που ακούσαμε και θα προσπαθήσω να είμαι λακωνική. Είναι αδύνατο κύριε Πρόεδρε σε μια έκθεση που εκ των πραγμάτων είναι περιορισμένη και έχει συγκεκριμένη έκθεση, να συμπεριληφθούν ε, όλα αυτά τα σχόλια που ακούσαμε σήμερα. Όταν μου λέτε αυτά που ακούσαμε για τη Βουλγαρία από τον ε, Βούλγαρο συνάδελφο, ήδη πέρυσι είχαμε παρόμοιες παρατηρήσεις ε, στην έκθεση. Εγώ προσπαθώ να αποκαταστήσω μια ισορροπία στην έκθεση. Δεν μπορώ να περιλάβω όλα τα σχόλια. Θέλουμε να είμαστε και κριτικοί, αλλά και ενθαρρυντικοί ταυτόχρονα. Και να επισημαίνουμε ε, τα σημεία που υπάρχουν αδυναμίες και που επιδέχονται περισσότερες βελτιώσεις και πρόοδο. Γι' αυτό σας παρακαλώ αγαπητοί συνάδελφοι, ας μην διαταράξουμε αυτή την ε, έθραυστη ισορροπία στην οποία έχει καταλήξει η έκθεση. Σε ό,τι αφορά τα πολιτικά κριτήρια, είχα πει ανέκαθεν ότι τα κριτήρια της Κοπεχάγης είναι η πεμπτουσία της συνεργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μια πολιτισμένη κοινωνία οφείλει να σέβεται και τα ατομικά και τα συλλογικά δικαιώματα. Και όλα αυτά τα δικαιώματα θα πρέπει να κατοχυρώνονται και από το κράτος δικαίου, αλλά να αποτελούν και αναπόσπαστο τμήμα της νοοτροπίας μιας κοινωνίας. Η κυρία Φλότρ απουσίαζε τη στιγμή που έκανα την εισαγωγή της έκθεσής μου. Αν ήταν όμως στην αίθουσα, θα είχε ακούσει ότι... Είχα πει είχα κάνει αναφορά των συνδικαλιστικών δικαιωμάτων και του δικαιώματο της απεργίας. Είναι απόλυτο σημαντικό, κυρία Φλότρ, να γίνουν σεβαστά τα θρησκευτικά δικαιώματα. Και αποτελούν πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι και μιλάμε για μικρές μειονότητες. Αν δούμε τους αλεβίτες και αν δούμε τη συζήτηση, πράγματι μπορούν να συμβούν ακόμη πολύ περισσότερα πράγματα Αντιλαμβάνομαι πως θα κατατεθούν ε, τροπολογίες, αλλά ελπίζω να γίνει σεβαστική βασική άποψή μου από τους συνάδελφους. Τώρα, για τα ΜΜΕ, προσπάθησα να το δω το θέμα όσο το δυνατόν πιο σοβαρά, για να κρίνω το τι συμβαίνει, αλλά δεν βρίσκω απαραίτητο να διαλέξω πλευρά. Είπα ήδη πως ε, το πρόστιμο στον όμιλο εκείνο είναι εξοντοτικό. Αλλά εγώ δεν μπορώ να ε, γνωρίζω το τι έχει κάνει αυτός ο όμιλος. Πρέπει λοιπόν να αποκτήσει η Τουρκία μια δομή ΜΜΕ που η οποία θα είναι υγιή για την ίδια τη χώρα και συγκρίσιμη με τις υπόλοιπε χώρες. Τώρα, για την ε, κυρία Μποσκούρτ και τα δικαιώματα των γυναικών. Όταν μιλάμε για τα δικαιώματα των γυναικών, ναι, είναι συμπιεσμένα σε μία παραγραφό. Μπορώ να προσθέσω άλλες δέκα παραγράφους, αλλά το να λέμε περισσότερα παραδείγματα δεν θα προσθέσει περισσότερο στην ουσία του πράγματος που αναφέρεται εκεί πέρα. Και ελπίζω και εδώ πέρα να μην έχουμε πάρα πολλές ε, τροπολογίες κατόπιν. Η σχέση με τους γείτονες, με την Κύπρο και με την Ελλάδα. Πέρσι, στην περσινή έκθεση και σας υπενθυμίζω πως Είχαμε αναφέρει εκεί πέρα τα δεδομένα για το τι θα γίνει το 2009. Εγώ διάλεξα λοιπόν εδώ πέρα στην παράγραφο 28 την εξή διατύπωση. Να την εφαρμόσει πλήρω την ε, σχετική συμφωνία χωρίς καθυστέρηση. Νομίζω αυτό είναι το σωστό. Κύριε Πρόεδρε, υπάρχουν κάποιες ε, παράγραφοι για το ΝΑΤΟ, επίση, για την Κύπρο. Ε, αν αναγνωρίσει η Τουρκία την ε, Κύπρο έχουν λυθεί όλα τα προβλήματα. Λύνονται πάρα πολλά πράγματα. Και, το, και ενεργειακή πολιτική και πάρα πολλά άλλα πρέπει να γίνουν κάποια βήματα. Κάποια βήματα από το τουρκικό κράτος και πραγματικά αυτό συζητιέται συνέχεια, αλλά ελπίζω τα βήματα αυτά να γίνουν και από την ελληνοκυπριακή κοινότητα και λέω στους Τούρκους ε, φίλους μου πως θα γίνουν πολύ ευκολότερα τα πράγματα εάν δείξετε πως έχετε καλές προθέσεις, αν κάνετε πραγματικά κάτι. Γιατί έτσι θα μπορέσουν και οι διαπραγματεύσεις στο νησί να κλείσουν επιτυχώς. Ε, και αυτό νομίζω είναι σκοπός ε, όλων μας. Νομίζω κύριε Πρόεδρε πως οι γενικές γραμμές ε, Αναφέρθηκα στα όσα είπαν οι συνόδελφοι. Σας ευχαριστώ και για τα καλά σας λόγια και ελπίζω πως θα μπορέσουμε τον Φεβρουάριο όταν θα ψηφίσουμε αυτή την έκθεση να έχουμε μια πλειοψηφία νομίζω γύρω στο 90% γιατί θα δώσουμε έτσι και ένα σαφές μήνυμα στην Τουρκία. Σας ευχαριστώ. Καλώς. Ευχαριστούμε την εισηγήτρια. Σας ευχαριστούμε για την τελική σας αυτή παρουσίαση. Ακριβέστατη υπήρξατε. Μπορούμε σύντομα να περάσουμε στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διατάξεως που προβλέπει ανταλλαγή απόψεων με την κυρία Άστον, ύπατη εκπρόσωπο της Ενώσεως και αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Χρησιμοποιώ αυτά τα λίγα λεπτά που μας χωρίζουν από την εξέταση του δεύτερου σημείου της ημερήσιας διάταξής μας για να σας δώσω κάποιες πληροφορίες όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο θα εξελιχθούν οι εργασίες. Βλέπω ότι κάποιος ζητά μια παρέμβαση. Ο κύριος Άτκινς, διαδικαστικό. Για το διαδικαστικό, συγγνώμη Πρόεδρε, σύντομα, όσον αφορά το τελευταίο σημείο που συζητήσαμε, έχουμε κάποιο χρονοδιάγραμμα για την υποβολή τροπολογιών και άλλα συναφή τέτοια. Πάμε να τι πληροφορίες σωστό. Προθεσμία υποβολή τροπολογιών είναι 15 Δεκεμβρίου στις 12 το μεσημέρι. Ναι, ήταν αναγκαία αυτή η διευκρίνηση. Τώρα στρέφομαι προς το δεύτερο σημείο που ήθελα να σας πω εκεί ότι, ότι ζήτησαν πολλοί να πάρουν το λόγο και εξαντλείται έτσι ο χρόνος που είχε καθοριστεί από τη διάσκεψη των Προέδρων. Και από τι υποχρεώσει τη κυρία Ήπα τη εκπροσώπου δεν μπορεί να ξεπεράσει το δίωρο παρουσία στη συνεδρίαση αυτή. Ζήτησαν παρέμβαση οι ομάδε. χρησιμοποιεί το σύστημα DONT οπότε κάθε ομάδα έχει σύμφωνα αυτού του όρους το χρόνο που τους διατίθεται και ζητώ συγγνώμη από τώρα από εσά διότι θα πρέπει να σεβαστώ αυτό το πίνακα με, και να επιβάλλω ιδιαίτερη πειθαρχία χρονική. Εάν ξεπεράσετε το χρόνο, εκ των προτέρων ζητώ συγγνώμη, δεν μπορώ να ξεπεράσω τον κανόνα, θα πρέπει να το κάνω, είναι αντιπαθητική κίνηση, αλλά θα πρέπει να σας αφαιρέσω το λόγο. Λοιπόν, αυτές είναι οι προϋποθέσεις και ζητώ από την κυρία Άστον να εισέλθει και να ξεκινήσουν οι εργασίες μας μαζί της. Λοιπόν, παρακαλώ, καθίστε, ούτως ώστε να ξεκινήσουμε τις εργασίες μας, την ημερίδα των εργασιών μας, με την κυρία Άστον, την οποία υποδεχόμεθα με μεγάλη ευχαρίστηση, μεγάλη τιμή για μας, να μπορούμε να τη φιλοξενούμε στην Επιτροπή μας λίγες μέρες μερικές ώρες σχεδόν ε, μετά την ανάλυση των καθηκόντων της. Αναζωογονείται έτσι η εξωτερική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και ισχυροποιούνται τα οικονομικά μέσα που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει διαθέσει για τον ρόλο αυτό για τη διπλωματική δράση δηλαδή, συντονισμένη διπλωματική δράση των 27 κρατών μελών, των πολλών ειρηνευτικών αποστολών που εκτελεί η Ευρωπαϊκή Ένωση στα πλαίσια των σχέσεων γειτονία και στα πλαίσια άλλων πολιτικών. Όσον αφορά λοιπόν αυτή την πολιτική που με την εφαρμογή της συνθήκης της Αβώνας θα ακολουθηθεί, βλέπουμε μια νέα όθηση που δίνεται από αυτό, την, αυτή τη θέση. Αναζωογονείται αυτός ο ρόλος και συνέβαλαν όμως οι προκάτοχοι της, ο κ. Ξαβιέ Σολάνα και η κυρία Μπενίτα Φερέρο Βάλτνερ που μαζί με όλους μας, όλοι μαζί θα θέλουμε να τους ε, χαιρετήσουμε και να θυμηθούμε τα όσα έκαναν. Κυρία Άστον, ο διορισμός σας στη θέση της ΥΠΑ της εκπροσώπου και αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι κάτι που θέλαμε να συμπέσει με την έναρξη της θητείας της Νέας Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θητεία που θα αναμιμοποιηθεί από δημοκρατική ψηφοφορία του νέου Κοινοβουλίου που έχει εκλεγεί ελεύθερα και εσείς πιστεύω θα θέλατε αυτή η συνάντηση να μπορούσε να εξελιχθεί σε αυτό το πλαίσιο. Όμως υπήρξαν καθυστερήσεις όπως γνωρίζουμε όσον αφορά την κύρωση της συνθήκης της Λισαβόνας και αυτό μας οδήγησε σε κάποια καθυστέρηση, σε κάποιες καθυστερήσεις και έτσι στην ανάγκη εξέβρεσης θεσμικής ισορροπίας που προβλέπεται τη συνθήκη. Κάτι που εφαρμόζεται με κάποια πρακτικά μέτρα προσαρμογής Ζητήσαμε λοιπόν στα πλαίσια αυτού του διορισμού σα, αναλήψη των καθήκοντων σα, να έρθουμε σε επαφή μαζί σα, σε αυτή την επιτροπή, για να συζητήσουμε στο δίωρο που θα μας αφιερώσετε τις διάφορες προκλήσεις που σας ε, περιμένουν. Μία παρατήρηση όσον αφορά το είδος του διορισμού που έλαβε χώρα, έχει 100 και κυβερνήσεων αποφάσισαν να διορίσουν ως ύπατη εκπρόσωπο ένα μέλος της ε, παρούσης Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και πιστεύω ότι μπορώ να υπογραμμίσω ότι αυτή είναι μια επιλογή που μπορούμε να θεωρήσουμε ότι είναι καλός ιονός για την δημιουργία μιας εξωτερικής πολιτικής που είναι πράγματι κοινοτική διότι νομιμοποιείται από την κοινοβουλευτική εμπιστοσύνη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή που εξέρχεται την είχε αποκτήσει αυτή η ψήφο εμπιστοσύνη. Αυτή η εμπιστοσύνη προέρχεται από ειλικρινή συνεχή διάλογο που σέβεται τις διάφορες απόψεις. Και εσείς η κυρία Άστον ως Επίτροπος δείξατε αυτό το σεβασμό για τα θεσμικά μας όργανα και για το ρόλο του δικού μας θεσμικού όργανου και εύχομαι και στα νέα σας καθήκοντα εσείς να δείξετε την ίδια ευαισθησία και την ίδια προσοχή που δείξατε μέχρι τώρα και ε, αυτό είναι εξυπηρετή και τις δικές σας εργασίες και τις δικές μας. Τις επόμενες εβδομάδες εσείς θα πρέπει να προετοιμάσετε τη δημιουργία της ε, Ευρωπαϊκής Διπλωματικής Υπηρεσίας. Για αυτή τη δημιουργία προβλέπει η συνθήκη τη διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο πνεύμα θεμητής συνεργασίας και σεβασμού των θεσμών, κάτι που προανέφερα και εσείς θα συμμετάσχετε την προσπάθεια. Πιστεύω ότι εσείς θα εξασφαλίσετε τη συμμετοχή, πλήρη συμμετοχή της Επιτροπής μας στις συζητήσεις που θα προηγηθούν και θα συνοδεύουν τις διάφορες νομοθετικές προτάσεις που θα υποβληθούν. Και τώρα, χωρίς περαιτέρω καθυστερήσεις, θα ήθελα να σας δώσω το λόγο ζητώντας από εσά, όπως ζήτησα και από όλους τους παρόντες συναδέλφους, να περιορίσετε το χρόνο των παρεμβάσεών σας σε περίπου ένα δεκάλεπτο. Αυτό πιστεύω είναι προς όφελος των καλών εργασιών της συνεδριάσεως μας. Έχετε το λόγο εσείς κυρία Άστον. Ε, Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμη Ευρωβουλευτέ, καταρχήν θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά για το προνόμιο που μου δώσατε να με προσκαλέσετε στη συνεδρίασή σας και χάρηκα ιδιαίτερα όταν επισημάνατε ότι ε, τρέφω ιδιαίτερο σεβασμό και εκτίμηση για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και αυτό το αναγνωρίσατε. Χαίρομαι ιδιαίτερο γι' αυτό και σας διαβεβαιώ ότι θα συνεχίσω να εμπλέκω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και θα έρχομαι όσο πιο συχνά γίνεται ενώπιόν σας. Θα ήθελα επίσης να πω όπως είπα και στην ε, Επιτροπή ΙΝΤΑ, στην οποία είχα πάει πολύ συχνά, και σε όλους τους ευρωβουλευτές. Ελπίζω να μου επισημαίνετε τις ανησυχίες σας ε, όποτε τις αισθάνεστε και να μην έχουμε μόνο τέτοιες ιδιαίτερες ευκαιρίες ε, για συζήτηση. Είναι πολύ σημαντική αυτή τη στιγμή η θέση σα σε ισχύ τη ηθίκη Λισαβόνα και χαίρομαι που έχουμε την ευκαιρία να το τονίσουμε και εδώ. Δέχτηκα αυτή την, αυτό το αξίωμα με τη φιλοδοξία να τηρήσω τι υποσχέσει μου και θα σέβομαι πιστά και τα κράτη-μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση και του Ευρωπαίου πολίτε. Και προσβλέπω σε στενή συνεργασία με τον πρόεδρο του Συμβουλίου, τον πρόεδρο τη Επιτροπή και του ε, υπουργού εξωτερικών και των 27 χωρών μέλων. Και φυσικά ε, με τους συναδέλφους της ε, Επιτροπής ως Αντιπρόεδρος, ε, αν και εφόσον επιβεβαιωθεί και η νέα τη σύνθεση. Αυτό είναι το νέο πνεύμα με το οποίο ήρθα σήμερα της καλύτερης ανάπτυξης και αξιοποίησης των σχέσεών μας και θα συνεχίσω την επικοινωνία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με ανοιχτό και ρεαλιστικό τρόπο. Πολλά αναφέρθηκαν για το κατά πόσο οι εμπειρίες μου ήταν σχετικές με το αντικείμενο που αναλαμβάνω. Πάντως, ε, ποτέ δεν ήμουν άνθρωπος που υιοθετούσε μια πολύ στενόμυαλη προοπτική. Έχω 27 χρόνια, 28 χρόνια εμπειρίας, ε, διαπραγματεύσεων, αναζήτηση συνένεσης και μάλιστα το τελευταίο χρόνο αναγνωρίστηκε και στο Ευρωπαϊκό, Συνοβου... στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ότι ήμουν κατάλληλη για αυτό το ρόλο. Μάλιστα πιστεύω στην σιωπηρή και, και διακριτική διπλωματία και όταν βλέπουμε τις προκλήσεις που μας περιμένουν γνωρίζουμε ότι το να δημιουργήσουμε την εμπιστοσύνη, να ανακτήσουμε την εμπιστοσύνη των πολιτών είναι πολύ σημαντικό και θα πρέπει φυσικά να κρατήσουμε τη μοίρα στα χέρια μας και γι' αυτό χρειαζόμαστε ανθρώπους που δεν θα μιλάνε μόνο αλλά θα ακούν και όλα, θα διδάσκονται και θα διδάσκουν και θα μπορούν να εργάζονται τόσο στο φως των προβολέων αλλά και στην, στο παρασκήνιο και ως υπουργό Δικαιοσύνης και ως μέλος της Βρετανικής Κυβέρνησης και στην Προεδρία της Βουλής των Λόρδων άσκησα με αυτό το πνεύμα τα καθήκοντά μου και ως επίτροπος, πρώην επίτροπος εμπορίου νομίζω ότι έχω συγκεντρώσει πολλά, πολλές γνώσεις και προσόντα και μάλιστα συνεργάστηκα ε, και θα συνεργαστούμε και στο μέλλον με τις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Ρωσία και την Κίνα και αισθάνθηκε ιδιαίτερη τιμή όταν ομόφωνα 27 χώρες μέλη με ενέδειξαν ως τον κατάλληλο άνθρωπο για το αξίωμα αυτό. Και ε, ε, βέβαια εξεπλάγει και κάπως. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να εξασφαλίσω μία συνέχεια της εξωτερικής πολιτικής μας και θα ήθελα να ποτίσω φόρο τιμή στο Χαβιέρ Σολάνα και στη Φενή, Μπενίτο Φερέρο Βάλτνερ, γιατί πραγματικά ήταν πολύ σημαντική η συνεισφορά τους ε, για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μια και είναι περιορισμένος ο χρόνος, θα ήθελα να πω ότι έχουμε μια πολύ σημαντική φήμη στον κόσμο, χάρη στις αξίες μας, ε, στις αρχές που μας είναι προσφυλείς. Και ήδη έχω ακράδαντη υπεποίθηση στις αρχές αυτές και πιστεύω ότι θα πρέπει να συνεχίσουμε με την ανθρωπιστική μας βοήθεια. Είμαστε ε, μισό δισεκατομμύριο άνθρωποι που συνεργαζόμαστε και θα πρέπει ε, να δείξουμε το πολιτικό μας βάρος ε, και να έχουμε πρωταγωνιστική θέση. Θα δείτε λοιπόν και συνέχεια αλλά και δυνατότητα αναθεώρησης ε, και αξιοποίησης του έργου που έχουμε σε ολόκληρο τον κόσμο και βλέπετε ότι είναι σαν ψηφιδωτό όλα αυτά τα διάφορα καθήκοντα που θα τα συγκεράσω μαζί. Και τις επόμενες εβδομάδες θα καταρτήσω κάποιες προτάσεις για την εξωτερική διπλωματική υπηρεσία και πιστεύω ότι ε, μπορούμε να διεκδικήσουμε μια ηγετική θέση, αξιοποιώντας ήδη το έργο του Συμβουλίου και της Επιτροπής και να διαμορφώσουμε μια νέα διπλωματική υπηρεσία που θα επιφέρει τη θεαμένη αξία στα κράτη-μέλη και θα είναι και μοναδική στις προτάσεις της. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κυρία Άστον. Είναι πολύ καλή αυτή. Ε, βολεύει το ότι ήσασταν συνοπτική για τη συνέχιση τη συζητήσεω. Τέσσερι παρεμβάσει δύο λεπτών θα ακολουθήσουν και μετά θα ακολουθήσει η απάντησή σα και έτσι θα πάμε μέχρι το τέλο, μέχρι ότου εξαντληθεί ο κατάλληλο των αγορητών. Ο κύριο Αλαφράγκα είναι ο πρώτος συντονιστής της ομάδας του ΕΛΚ για δύο λεπτά. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Άστον, εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος θα ήθελα να σας, να θερμά για το διορισμό σας και να, ευχαριστήσω, σας ευχαριστήσω για το ότι ήρθατε αμέσω στην ε, Επιτροπή, κάτι που δείχνει τη βούλησή σας να εμπλέξετε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θα έχουμε μέχρι τον Ιανουάριο το χρόνο να σας στείλουμε το αριθματολόγιο και να μάθουμε τις προθέσεις και τις προτάσεις σας ε, στα θέματα της εξωτερικής διπλωματικής υπηρεσίας. Αυτό που ενδιαφέρει την πολιτική μου ομάδα είναι αν είστε διατεθειμένοι να αναμίξετε πλήρω αυτή τη μεταβατική περίοδο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ιδιαίτερα στα θέματα των αρμοδιοτήτων που λαμβάνουμε από τη συνθήκη. Επίση, έχετε αποσαφηνίσει τι γεωγραφικέ υπηρεσίε ε, θα βρίσκονται άμεσα υπό τη δική σα ε, αιγίδα και ποιε θα εξαρτώνται από του άλλου επιτρόπους. Έχετε συγκεκριμένε. Ε, απόψη για το πού θα, που θα εδρεύσει το γραφείο σας, το Συμβούλιο στην Επιτροπή. Κάποιος συμπατριώτης σας είπε δεν θα πρέπει να... Ε, για και το Συμβούλιο να μην προκαλέσει συμφόρηση στην, ε, στη Ουάσιγκτον, ε, στη Μόσχα ή στο Τόκιο. Εμείς δεν έχουμε τέτοια φιλοδοξία. Θέλουμε μια κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας που θα είναι ορατή, δίκαιη και κυρίως θα συνάδει με τις αρχές και τις αξίες που όλοι προασπίζουμε. Επίσης θα ήθελα να σας δείσω να έχετε οραματικότητα, πεποίθηση, φιλοδοξία, δέσμευση προς τα ευρωπαϊκά πράγματα και το ευρωπαϊκό όραμα, αλλά και πίστη και θεσμική αφοσίωση. Τα 27 κράτη-μέλη δεν κατάφεραν ομόφωνα να υποστηρίξουν την υποψηφιότητα ε, στην ε, ε, Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών ένα ευρωβουλευτή και συμπατριώτη σα. Ευχαριστώ κύριε Σαλαφράγκα που ήσασταν σχολαστικό στην τήρηση του χρόνου, συντονιστή τη ολιστική ομάδα Βίγκενινγκ. Για δύο λεπτά ακολουθεί. Μπορείτε να πάρετε το λόγο, κύριε Βίγκενινγκ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Λέδη Άστον, εξ ονόματος ε, της ομάδας ε, των Σοσιαλιστών και των ε, Δημοκρατών σας καλωσορίζω στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με την ιδιότητά σας της είπα της εκπροσώπου εξωτερικής πολιτικής και αντιπρόεδρο της Κομισιόν που είναι δύο πτυχές της ίδιας δουλειάς και δεν μπορούν να διαχωριστούν. βεβαίω οι, ακροασει οι ακροάσεις θα γίνουν τον Ιανουάριο, αλλά νομίζω ότι μπορούμε ήδη να συζητήσουμε για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το γεγονός πως τη δεύτερη ημέρα των καθηκόντων σας βρίσκεστε εδώ πέρα δείχνει την διαθεσή σας να συνεργαστείτε και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί η συνθήκη της Λισαβόνας που ετέθη χτες ε, σε ισχύ δεν δημιούργησε μόνο το δικό σας αξίωμα αλλά μας έδωσε εμά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο νέες ευθύνες και νέες αρμοδιότητες και τις επόμενες εβδομάδες ε, και μήνες θα δεχτείτε πολλές πιέσεις γιατί εργαζόμαστε με ένα νέο σύστημα και θα πρέπει να μπορέσετε να βρείτε κι εσείς ε, μια ισορροπία μεταξύ της ε, κοινοτικής και της διακυβερνητικής ε, μεθόδου και δεν χρειάζεται να σας πω ποια προτιμούμε. Σας εύχομαι καλή επιτυχία λοιπόν. Τώρα να περάσω στις ερωτήσεις. Υπάρχουν κάποια θετικά ζητήματα στις ευρωρωσικές σχέσεις. Συμφώνησε όσον αφορά το ιρανικό πρόγραμμα μαζί μας ο κύριος Μετβέντεφ ε, και μίλησε για την καταπολέμηση διαφθορά και τι δίκαιε εκλογέ. Τι πρέπει να κάνει λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση για να λύσει τις ενεργειακές διαφορές Ευρωπαϊκή Ένωση Ρωσία που αποτελούν σημείο και ευκαιρία και πρόκληση και τι σκοπεύει να κάνει για να ξαναξεκινήσει ο διάλογο με τη Ρωσία για δημοκρατία, κράτο δικαίου και ανθρώπινα δικαιώματα. Ευχαριστώ. Σα ευχαριστώ κύριε Βίγκενινγκ. Η συντονίστρια της ομάδας Άλτε, η κυρία Νέιτς, έχει το λόγο για δύο λεπτά. Κύριε Πρόεδρε, κυρία εκπρόσωπε, αγαπητοί συνάδελφοι, το βράδυ του διορισμού σας ε, έλειψαν πάρα πολλές φωτογραφίες και μία από αυτές έκανε το γύρο του κόσμου και είναι ταυτόχρονα και καθησυχαστικό και ανισχυτικό. Ήταν τέσσερα άτομα, ήταν εκεί πέρα και ο πρόεδρος Κομισιόν στο κέντρο και ο πρόεδρος Συμβουλίου ο κύριος ε, Ράινφελτ και στις άκρες ο κύριος ε, Φαν Ρόμπα, μόνιμος πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και στην άλλη άκρη εσείς. Θεωρώ πως ε, βεβαίως το πως ήσασταν τοποθετημένοι δεν σημαίνει ακριβώς και την σημασία των ε, καθηκόντων σας, αλλά πράγματι δείχνει πως η Προεδρία θα προσπαθήσει να διαφυλάξει τα δικαιώματά της. Πώς σκοπεύετε να εργαστείτε εσείς σε αυτό τον ε, λαβύρινθο για να αποφύγετε έτσι πολέμους όσον αφορά τις αρμοδιότητες. Τέλος, όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικών Σχέσεων, είπατε κάποια πράγματα. Ε, τον ε, Απρίλιο θα υποβάλει μια πρόταση το Συμβούλιο μετά από δική σας βεβαίως ε, μετά από ένα δικό σχέδιο πρόκειται λοιπόν για μια ευκαιρία μοναδική για οικοδόμηση μιας πραγματικά ευρωπαϊκής διπλωματίας και υπάρχουν και εδώ πέρα βεβαίως κάποια κεκτημένα ε, δικαιώματα αν θέλετε υπάρχουν εθνικά Φέουδα. Πώς σκοπεύετε λοιπόν εσείς να εργαστείτε εδώ πέρα, κυρία εκπρόσωπε. Ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ κυρία Νέιτς. Τώρα η συντονίστρια των Πρασίνων, η κυρία Λούνατσεκ, για δύο λεπτά. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Εκ μέρους των Πρασίνων θα ήθελα να σας καλωσορίσω εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Σας ευχαριστώ που ήρθατε για να μοιραστείτε αυτό το δύο ώρο μαζί μας. Κυρία Βαρόνη, πρώτα απ' όλα η Ευρώπη χρειάζεται ενιαία και ισχυρή φωνή και κοινό πρόσωπο το οποίο θα εμφανίζεται και προς τα μέσα και προς τα έξω για να τελειώσει επιτέλους αυτή η κατακαιρματισμένη κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας και να έχουμε πρόληψη των ε, συγκρούσεων όπως αναφέρεται και στην συνθήκη της ε, Λισαβόνας. Πρέπει λοιπόν αυτό το ευρωπαϊκό συμφέρον να αντιπαρατηθεί στα εθνικά στους εθνικούς ε, μονόδρομους όπως είχαμε παραδείγματος χάρη ε, στην περίπτωση του πολέμου του Ιράκ. Είστε στην χώρα σας ε, γνωστοί ως φιλοευρωπαία και ελπίζω το ίδιο να δείξετε εδώ πέρα. Πώς θα διασφαλίσετε λοιπόν το ότι δεν θα γίνεται πραγματικά το μακρύ χέρι του Foreign Office. Ελπίζω να τα καταφέρετε, έχετε την στήριξή μας. Επίσης, η συνοχή εσωτερική και εξωτερική της ευρωπαϊκής πολιτικής ασφάλειας ε, αφορά πολλούς ε, επιτρόπους, ε, διεύρυνση, αναπτυξιακή βοήθεια κτλ. Τι σκοπεύετε να κάνετε προς τα έξω, π.χ. η μεταρρύθμιση του ΟΗΕ που θα οδηγήσει μακροπρόθεσμα σε μια ενιαία έδρα στο Συμβουλίο Ασφαλείας τη Ευρωπαϊκής Ένωση, τέλο για τα Βαλκάνια. Εδώ πέρα στη Βοσνία η συνταγματική διαδικασία έχει κολλήσει, δεν προχωράει. Τι σκοπεύετε να κάνετε για να οδηγηθούμε σε μια λύση για να υπάρξει μια δυνατότητα ένταξης της Βοσνίας και για το κοσφοπέδιο είστε υπέρ του άμεσου διαλόγου για την βίζα, για την απελευθέρωση της ε, βίζας για τους κατοίκους του Κοσμοβιδίου όπως αποφάσισε και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ. ευχαριστώ κυρία Λουνάτσεκ. Η κυρία Άστον έχει το λόγο. Παρακαλώ και εσείς κυρία Άστον να τηρήσετε το πεντάλεπτο για την απάντηση στις πρώτες τέσσερις ερωτήσεις. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Εντός πενταλέπτου Αναγκαστικά θα είμαι σύντομη. Κύριε Σαλαφράγκα, σας ευχαριστώ για τις ευχές σας. Νομίζω ότι σωστά περιμένετε να δείτε τι σχέση θέλω να έχω με το Κοινοβούλιο. Θέλω να σεβαστώ πλήρω τη συνθήκη και να σεβαστώ πλήρω το Κοινοβούλιο. Τώρα πώς θα λειτουργήσει αυτό. Εμείς θα πρέπει να το καθορίσουμε μαζί. Οι τελικές αποφάσεις και ευθύνε είναι ξεκάθαρο που ανήκουν. Διάβασα λεπτο σε κάθε λεπτομέρεια τη συνθήκη για να την περάσω το κοινοβούλιο μου. Αλλά ποτέ δεν δίστασα από το να αναλάβει τη σωστή θέση, τη θέση που τα αρμόζει το κοινοβούλιο αυτό το διάλογο. Πρέπει να συζητήσουμε πώς θα εφαρμοστεί αυτό. Τώρα, κατά πόσο θέλω να σταματήσω την κυκλοφορία του ΣΥΠΗΝ. Θέλω να ρέει η κυκλοφορία. Αυτό που έχει σημασία για μας είναι ποικιλοτρόπος και με συντονισμένη φωνή καμιά φορά και καμιά φορά με πιο ησυχή φωνή να ξεκαθαρίζουμε τη θέση της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, ποιες είναι οι αξίες μας. Να παίξουμε το ρόλο μας για να λειτουργήσουν καλύτερα τα πράγματα. Ρωτήσατε για τη διαφωνία στον αφορά το Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ. Δεν με εκπλήσει αυτό. Με 27 κράτη-μέλη να έχουμε διαφορετικές απόψεις και μέσα προκλήσει που αντιμετωπίζουν είναι η συνεργασία με τα 27 κράτη-μέλη. Για να βρούμε το κοινό νήμα, όχι τον ελάχιστο κοινό παρονομαστή, τον ε, υψηλότερο, το υψηλότερο δυνατό επίπεδο συνεργασία. Ευχαριστώ που οι σοσιαλιστέ με όρισαν Συμφωνώ. Ε, πρέπει να συνεργαστούμε όσο πιο στενά γίνεται. Είμαι ο σύνοδο κορυφή στη Στοκχόλμη. Παρέστην σε όλε τι συνόδου κορυφή με τη Ρωσία τον τελευταίο χρόνο. Αυτό που λέει ο πρόεδρο Μετβέτεφ είναι αρκετά ενδιαφέρον. Δηλαδή το πώ προσεγγίζει το μέλλον της Ρωσίας. Θα πρέπει να συνεργαστούμε στενά μαζί τους. Συζητήσαμε ενεργειακά θέματα, βεβαίως, και θα πρέπει να συνεχιστεί αυτό. Πιστεύω όμω ότι όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα, κράτο δικαίου κλπ. όλα αυτά τα θέματα θα πρέπει να συνεχιστούν οι συνομιλίε με τη Ρωσία και ήδη όπω προανέφερα είχα την δυνατότητα να παρακολουθήσω του διαλόγου και ω Επίτροπο Εμπορίου να διεξαγάγω διαλόγο ε, και με τον πρόεδρο και της Ρωσίας και με τον πρωθυπουργό και θα συνεχίσω συνομιλίες. Ευχαριστώ επίσης και την ομάδα του Άλτε. Αναφερθήκατε στη φωτογραφία. Δεν ήξερα πού βρισκόμουν όταν μου πήραν τη φωτογραφία. Μπήκα σε μια αίθουσα, μια φωτογραφία. Φεύγω για τη Μαδρίτη το απόγευμα. Πάνω να συναντηθώ με την νέα Προεδρία, να διπνήσω με, τον υπουργό, με του Υπουργού Εξωτερικών, να συνομιλήσω με τον Πρωθυπουργό τη Ισπανία το απόγευμα. Θα μπορέσω να συνομιλήσω με εκείνους. Θα πρέπει να συνε... χρησιμοποιήσουμε την ενέργεια της εναλλακτική προεδρίας, να χρησιμοποιήσουμε τι δυνατότητες που προσφέρουν τα κράτη-μέλη σοφά και καλά. Ξέρω τι, σημαίνει αυτό για το δικό μου ρόλο, αλλά μπορούμε να κερδίσουμε πολλά αν βρούμε τη σωστή διαδικασία. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Δεν έχω καμία αμφιβολία ότι μπορώ να τα καταφέρω. Μπορώ να συνεργαστώ στενά με του συναδέλφου, αλλά πρέπει να είναι ξεκάθαρος και ο ρόλος μου. Όσον αφορά την υπηρεσία εξωτερικής δράσης, Υπάρχουν πολλά σχέδια που έχω ε, να βρω τρόπους ούτως ώστε να μπορούμε να ηγηθούμε στον κόσμο. Και θέλω να βρω τη μοναδική πρόταση που πουλάει, όπως την αποκαλώ. Κύριε Νόνατσεκ, ευχαριστώ ξανά. Θέλετε να μιλάμε με μία φωνή, συμφωνώ. Εγώ δεν θα είμαι επέκταση της Βρετανικής κυβερνήσεως. Διορίστηκα από τα 27 κράτη-μέλη και όπως έκανα και με το εμπόριο θα αντικατοπτρίζω πιστά τι απόψει τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχετε δίκιο. Είμαι, είναι γνωστό στη χώρα μου ότι είμαι υπέρ τη Ευρώπη και είμαι υπερήφανη που αυτή είναι η φήμη που με ακολουθεί. Είναι πολύ σημαντικό να είναι συνεπεί οι δράσει μα. Όσον αφορά τον ΟΗΕ τώρα, το ρόλο τη ΕΕ τη εκπροσώπου είναι να μιλά εκ μέρου των 27 κρατών μελών όταν υπάρχει συμφωνία. Αυτή είναι η θέση. Και έτσι θα παραμείνει όσον αφορά τη Βοσνία. Πολλά πρέπει να γίνουν. Τα συζήτησα, συζήτησα το θέμα αυτό ήδη, τη Συμφωνία Βερολίνο-ΣΥΝ και πώ μπορεί να χρησιμοποιηθεί αυτή η συμφωνία. Υπάρχουν πάρα πολλά που μπορούν να γίνουν, δεν έχω χρόνο να μπω σε Ε, Διάλογο για το κοσυφοπίδιο θα πρέπει να γίνει πάρα πολύ δουλειά ακόμα όσον αφορά και αυτό το θέμα. Σας ευχαριστώ κυρία Άστον. Τώρα θα στραφούμε ίσως και σε κάποιες απαντήσεις που ίσως να μην κάλυψαν πλήρως ερωτήσεις. Ίσως προς το τέλος θα σας υποβάλω κι εγώ κάποια ερώτηση. Δύο λεπτά, Συντονίστε του ECR, ο κύριος Τάνοκ. Έχετε δυνατόν να παλεύετε κύριε Τάνοκ. Κύριε Πρόεδρε, λέει Άστον, πρώτα απ' όλα η συνάδελφός σας από τους εργατικούς η Μεριχάνιμπολ μου είπε ότι δεν θέλω να γίνει γυναίκα είπατε εκπρόσωπος. Δεν με απασχολεί αυτό. Το αυτό που με απασχολεί είναι η εμπειρία και τα προσόντα σας. Εγώ δεν είχα κανένα πρόβλημα για την ε, κυρία Φέρερο Βάλτνερ, η οποία βεβαίως είχε πάρα πολλά προσόντα ως ε, σας. Ο δε κύριος ε, Χαβιέ Σολάνα ήταν υπουργό Εξωτερικών ε, της Ισπανίας και Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ πριν αναλάβει τα καθήκοντά του. Εδώ μέσα σε αυτή την Επιτροπή υπάρχουν πολλοί πρώην Υπουργοί Εξωτερικών. Οπότε η ομάδα μου θέλει να γνωρίζει γιατί θεωρείτε ότι εσείς ε, πρέπει να καταλάβετε αυτή τη θέση ενώ υπάρχουν άλλοι πιο ικανοί. Τώρα για την πολιτική, για την ε, κοινή πολιτική έμνες και ασφαλείας. Τι θα, κατα... τι θα κάνετε στην προσπάθεια Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, Ουκρανίας να προειδοποιήσετε την ε, ρωσική κυβέρνηση να μην παρέμβει στις ε, Ουκρανικές εκλογές και πόσο θεωρείται ότι αποτελεί σημείο τριβής η Κρυμαία. Τώρα για τον Νότιο Κάφκασο, τον Αγκόρνο Καραμπάχ, τι θεωρείται ε, ότι πρέπει να γίνει σχετικά με τις δηλώσεις ε, του Προέδρου του Αζερβαϊτζάν που απειλήσε με χρήση βίας για ανακατάληψη του θυλάκου και για το ότι η Τουρκία είπε πως πρέπει να λυθεί αυτή η κατάσταση ως προϋπόθεση για την ομαλοποίηση των σχέσεων ε, με την Αρμενία, δεδομένης επίσης ε, της αποστολής ε, δυνάμεων του ΝΑΤΟ στο κέρας Αφρικής, τι θεωρείτε ότι είναι η προσθέμενη αξία της αποστολής της Αταλάντα. Και τέλος, ποιο είναι το νόημα του να έχουμε εδώ πέρα στρατιωτική δομή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και τέλος, ως εργατική πολιτικός θεωρείτε ότι θα μπορέσετε να αντισταθείτε στις πιέσεις ε, των συνδικάτων που θέλουν να σταματήσουν την εμπορική συμφωνία με την ε, Κολομβία και επίσης με την κοινότητα των Αμήλα από το Ηνωμένο Βασίλειο που θέλουν να σταματήσει την αντίστοιχη συμφωνία με τη Σρι Λάνκα. Ευχαριστώ κύριε Τάνοκ. Για την ΚΟΕ. Λέζινγκ. Κυρία Λέζινγκ, συντονίστρια. Εξ ονόματος των, αριστερών, με συγχωρείτε, σας ε, καλωσορίζω. Να περάσω στις ε, ερωτήσεις. Μέχρι τον Απρίλιο του 2010 θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η δομή της εξωτερικής υπηρεσίας. Η Σουηδική ε, Προεδρία είπε πως θα πρέπει να είναι ένα σουηγενερής οργανισμός ανεξάρτητος από Συμβούλιο και Κομισιόν. Όμως νομίζω ότι θα έπρεπε εδώ πέρα να εκμεταλλευτούμε την ευκαιρία για έναν εκδημοκρατισμό της ΚΕΠΑ. Ποια επιλογή προτιμάτε εσείς επίσης. Βλέπετε πως ε, θα εκπροσωπούνται περισσότερο τα πλούσια κράτη-μέλη στη στελέχωση αυτής της ε, υπηρεσια Δεν θεωρείτε λοιπόν πως υπάρχει εδώ πέρα παραβίαση του ευρωπαϊκού ιδεώδους ε, και ένα δημοκρατικό έλλειμμα και ένα συγκεκριμένο ερώτημα για την Σομαλία, γιατί αναφέρθηκε ήδη η Αταλάντα. Υπάρχουν πληροφορίες πως ε, η Σομαλία θα λάβει κονδύλια από το μέσο σταθερότητας ε, για συμβούλους. Αυτό σημαίνει πως θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε την ε, τωρινή μεταβατική κυβέρνηση η οποία συνεχίζει να εφαρμόζει όλο και περισσότερο την Σαρία και την ταπείνωση των γυναικών. Αυτό είναι το αποτέλεσμα της ε, μέχρι τώρα επιμόρφωσης. Τι εννοεί η Ευρωπαϊκή Ένωση όταν λέει σταθεροποίηση. Το γεγονός επίσης ότι έχετε το δικαίωμα να προτείνετε τον προϋπολογισμό της υπηρεσίας σας. Πόσο θα είναι αυτός, ε, επίσης σκοπεύετε να τον εκμεταλλευτείτε και για στρατιωτικές ε, κινήσεις και αντιλαμβάνομαι σωστά, προτείνετε εσεί τον προπολογισμό και μετά θα τον εγκρίνει με ειδική πλειοψηφία το ε, Συμβούλιο και δεν έχει εδώ πέρα κανένα ρόλο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κυρία Λούζιν. Εν ονόματι του FD, Μπάνερμαν για δύο λεπτά. Ο κύριος Μπάνερμαν βαρώνει αν σας αρέσει η επιστημονική φαντασία, κυρίως η σειρά Dr. Who του BBC, η σειρά, και έχετε και ένα από τα ρομπότα, Dalek στο σπίτι σας, αυτό έχει σημασία. Τώρα, ο δόκτορας έχει τη χρονομηχανή του και εσείς εμφανιστήκατε κάπως έτσι, από το πουθενά. Ε, ε, πρέπει να σας ρωτήσουμε ποιο είναι το παρελθόν σας και η παρουσία σας εδώ πέρα. Είσαστε ικανοί, αλλά υπάρχουν κάποια σοβαρά ερωτήματα τα οποία θα πρέπει να απαντήσετε και θέματα να καλύψετε. Μπορείτε να ξεκαθαρίσετε λοιπόν, όταν είσαστε υπουργός, ε, όταν υπεύθυνοι για την αφοπλισμό, πυρηνικό 1982 στο Ηνωμένο Βασίλειο, δεν πήγατε χρήματα από χώρε του Σοβιετικού μπλοκ ή από το Κομμουνιστικό Κόμμα του Ηνωμένου Βασιλείου άμεσα ή έμεσα μέσω άλλων διάβλων. Γι' αυτό δεν εννοώ άμεσα από τη Ρωσία τη Σοβιετική Ένωση. Αυτό το αποκλείεται. Αλλά τότε πήρατε χρήματα από κάποια άλλη χώρα της Σοβιετικής Ένωσης ή φορέα κομμουνιστικό ή οργάνωσης που ε, ε, ήταν πλησίον στο Κομμουνιστικό Κόμμα. Το ότι ήσασταν ε, ταμείας του CND ε, και δαρνηθήκατε να ονομάσετε κάποιο δωρητή και λέγεται μάλλον ερευνητές σοβιετικοί πήραν χρώματα από το CND και υπάρχει τεκμηρίωση ότι υπήρχαν, ήρθαν και πόροι στο CND από την KGB και έγινε έλεγχος το 1993 που είδαν ότι οι πόροι του CND 40% των πόρων του CND δεν μπορούσαν να βρεθούν από πού προερχόταν όλες οι χώρες που εκπροσωπούνται εδώ που είχαν την ατυχία να ζουν υπό κομμουνιστικό καθεστώς και όλες οι χώρες του ΝΑΤΟ που εκπροσωπούνται εδώ ε, ήταν στόχος του CND και το CND προσπαθούσε να υπονομεύσει αυτές τις χώρες και γι' αυτό χρειαζόμαστε μια σαφή απάντηση για το Campaign for Nuclear Disarmament. Ευχαριστώ κύριε Μπάνεμαν για τους μη εγγεγραμμένου. Μάντλενερ για δύο λεπτά. Eh, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ακούσαμε πολλές ερωτήσεις κυρίως από τους Βρετανούς ε, συναδέλφους και η ερώτηση την οποία θα ήθελα να κάνω και εγώ είναι ότι θα εκπροσωπείτε προσεχώς 27 χώρες με 27 διαφορετικά οράματα. Και μιλήσατε μίλησε μόνο με συγχωρείτε πρόσφατα η Σουηδική Προεδρία για την Ιερουσαλήμ ως ε, πιθανή πρωτεύουσα ενός ε, ανεξάρτητου Παλαιστινιακού κράτους. Ε, έχετε την δυνατότητα εσείς να κάνετε επιλογές και τι γίνεται με τα συμφέροντα των μικρότερων χωρών όπως η Ολλανδία. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κύριε Μάτνερ. Κυρία Άστον, βλέπω ότι είναι δύσκολο να απαντήσετε σε πέντε λεπτά αυτά που σας διαθέτω σε ρηπές ερωτημάτων που είναι πολλές και κάθε ερώτηση έχει υποερώτηση αλλά δείξατε την ικανότητά σας και δείχνει την ικανότητά σας και σε αυτό. Σε πέντε λεπτά λοιπόν, λέει Άστον. Ευχαριστώ. Θα κάνω ό,τι μπορώ. Κύριε Τάνοκ, ρωτήσατε καταρχήν γιατί εγώ θα πρέπει να καταλάβω αυτό το αξίωμα. Η απάντηση είναι γιατί 27 αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων με διόρισαν. Μπορεί να μην με διαλέγατε εσείς, αλλά με διάλεξαν οι 27 και θα αναλάβω αυτό το έργο με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Σε ό,τι αφορά τα προσόντα και την εμπειρία μου ε, ως προς το Κοινοβούλιο, τρέφω ιδιαίτερο σεβασμό για το Κοινοβούλιο και υπάρχουν άνθρωποι που είχαν πραγματικά τεράστια πείρα και πολύ πλούσια πείρα και ευρωβουλευτέ και θα προσπαθήσω να την αξιοποιήσω και θα ζητήσω τη βοήθειά του για το έργο μου. Πάντω τα προσόντα μου πιστεύω ότι είναι κατάλληλα για το αξίωμα αυτό. Σε ό,τι αφορά την Ουκρανία, έγιναν κάποιε συζητήσει ε, μεταξύ του Πρωθυπουργού τη Ουκρανία και του Προέδρου τη Ρωσία. Δεν ξέρω ποια ήταν η έκβαση αυτών των συνομιλιών. Θα δούμε τι θα γίνει και με τι εκλογέ. Πάντως θα είναι καλό, καλή σφιγμομέτρηση για τη δημοκρατία αυτές οι εκλογές. Δεν προλαβαίνω να απαντήσω σε όλες τι ερωτήσει. Ό,τι αφορά την επιχείρηση Αταλάντη και τον Άβαρχο Χάτσον, το έργο του, νομίζω ότι θα συμβάλλει αυτή η επιχείρηση. Φυσικά δεν είναι επαρκή. Θα πρέπει να συνεργαστούμε με την Αφρικανική Ένωση και να δούμε τι θα γίνει στην επόμενη διάσκεψη κορυφή με την Αφρική γιατί θα έχουμε και κάποιε χερσαίε επιχειρήσει Πάντω, ο στρατηγό Λίκη χθε με ενημέρωσε για τα θέματα αυτά. Δεν φοβάμαι που προέρχομαι από το Εργατικό Κόμμα. Φυσικά θα ε, έχουμε και το θέμα της ε, Συμφωνίας Ελεύθερου Εμπορίου με την Κολομβία. Υπάρχουν περιπτώσεις ε, όπου πρέπει να δεσμευτούμε και αλλού να αποδεσμευτούμε. Στην περίπτωση της Κολομβίας πιστεύω ότι καλό θα ήταν να δεσμευτούμε, να εμπλακούμε στο θέμα αυτό. Τώρα για το θέμα της εξωτερικής υπηρεσίας που θα είναι ανεξάρτητη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ποια είναι η δική μου προτίμηση, μα μην ξεχνάτε ότι μας δεσμεύει η συνθήκη και είναι πολύ σημαντικό ο, στις πρώτες αποστολές του, της, εκπροσώπου να προσέξουμε να τηρήσουμε αυτή τη συνθήκη που μετά από πολύ κόπο εγκρίθηκε. Και ε, η μελλοντική διπλωματική υπηρεσία πιστεύω θα έχει τέτοια μορφή που θα καθιστά υπερήφανους και τους ευρωβουλευτές και τα κράτη-μέλη. Τα μικρότερα κράτη-μέλη είναι εξίσου σημαντικά και θα πρέπει να εξασφαλίσουμε την ανάμειξή τους και στην ε, υπηρεσία εξωτερικών δράσεων και γενικώ στο έργο μας. Ήδη ε, γευμάτισα με ε, προσώπους της ΜΕΑ και θα εξασφαλίσω συμμετοχή όλων των κρατών ε, στις προσπάθειες αυτές για τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Εξωτερικής Υπηρεσίας. Για τη Σομαλία μίλησα, δεν πρόκειται να αναφερθώ. Τώρα κονδύλια δεν τα γνωρίζω, τα συγκεκριμένα. Κύριε Καμπεμπάνεμαν, ήταν πολύ ωραία όταν ήπιαμε στη Γενέβη τη Δευτέρα ένα ποτήρι σαμπάνιας και τότε με είχατε προειδοποιήσει για αυτές τις ερωτήσεις. Και είναι λογικό να μου θέτετε τέτοιε ερωτήσει για το παρελθόν μου και το ιστορικό μου. Αλλά το 1992 ε, είναι χρόνια ολόκληρα πριν. Θα προσπαθήσω να απαντήσω όσο καλύτερα μπορώ. Πάντως δεν έλαβα ε, χρήματα άμεσα από καμία σοβιετική χώρα. Ήμουν μέλος του Εργατικού Κόμματος. Η εκστρατεία για τον πυρηνικό αφοπλισμό ήταν μια οργάνωση και αυτό είναι το καλό της δημοκρατίας. Ότι τόσα χρόνια μετά μπορείτε να μου θέτε τέτοια ερωτήματα και να σας απαντώ. Τα 38% των κονδυλίων ε, δεν υπησέρχονται ε, στον έλεγχο και μάλιστα εγώ διέταξα τον πρώτο έλεγχο και γινόταν ε, ε, διαδηλώσεις και γίνονταν έρανοι εκεί και τότε ως ναι είχαμε τέτοια πολύ σημαντικά ιδανικά και νομίζω ήταν πολύ σημαντικό και τα χρήματα μαζεύουμε σε κουβάδες δεν ξέρω από πού προέρχονταν φαντάζομαι δεν σας εκπλήσει Ελπίζω την επόμενη φορά να με <laughs> θέσετε ερωτήσει για την εξωτερική πολιτική. Τώρα για τις 27 διαφορετικές προοπτικές και τα 27 διαφορετικά οράματα εξωτερικής πολιτικής. Ναι, θα πρέπει όμως να βρούμε τρόπους συνεργασίας μεταξύ μας. Και αυτό που είναι πολύ ενδιαφέρον για πάρα πολλά θέματα, ακόμη και αν υπάρχουν διαφωνίες ε, σε διάφορες πτυχές της εξωτερικής πολιτικής, για το Κωσυφοπέδιο, για παράδειγμα, όλοι υποστήριξαν τις ε, αποστολές της ΕΠΑ. Και η συνεργασία με τα κράτη-μέλη είναι πολύ σημαντική. Για παράδειγμα, το χαρτοφυλάκιο του εμπορίου, πολύ δύσκολα οικονομικά θέματα, πολύ δύσκολες βιομηχανίες. Θα πρέπει να βρούμε κοινούς παρανομαστές για να προχωρήσουμε. Και αυτό είναι το ζητούμενο. Αλλά το στόχος μας είναι αναβάθμιση και εναρμόνιση προς τα πάνω, όχι κατά ανάγκη προς τον ελάχιστο κοινό παρανομαστή. Σας ευχαριστώ κύριε Άστον. Περνάμε στην τρίτη ομάδα ερωτήσεων. Προβλέπει παρέμβαση ενός λεπτού και μόνο για κάθε αγορητή. Θα σας πρότεινα να Πηγαίνετε κατευθείαν στο ερώτημα. Πρέντα. Ελκ. Ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κυρία Άστον, έχω δύο ερωτήσεις. Καταρχήν, ποιο κατά τη γνώμη σας είναι το μέλλον των διατελετικών σχέσεων και στα πολιτικά θέματα αλλά και στα θέματα άμυνας. Πιστεύετε ότι θα υπάρξουν δυσκολίες στην πολιτική συνεργασία ή περισσότερες δυσκολίες στα θέματα άμυνας στις διατλαντικές σχέσεις. Δεύτερη ερώτηση για την ε, ανατολική εταιρική σχέση. Παρακαλώ δείξτε λίγη φαντασία. Ποια πιστεύετε θα είναι η μορφή αυτής της ανατολικής εταιρική σχέσης τα επόμενα δύο χρόνια. Και για τη δημοκρατία τη Μολδαβία. Εκεί μια... ανέλαβε μία φιλοευρωπαϊκή ευρωπαϊκή κυβέρνηση μετά τις τελευταίες εκλογές ε, μια κυβέρνηση που θέλει να υλοποιήσει τους στόχους της εταιρικής σχέσης. Και θα είναι η Μολδαβία η Λιδία ηλίθος κατά τη γνώμη σας για αυτή την ε, ανατολική εταιρική σχέση. Σας ευχαριστώ κύριε Πρέντα. Ο κύριος Χάουιτ έχει το λόγο για ένα λεπτό. Κύριε εκπρόσωπε, συγχαρητήρια για τον διορισμό σας. Ε, κύριε Τάνοκ, θα ήθελα να γνωρίσω το ποια είναι η προσθεμένη αξία στον ευρωπαϊκό τουρισμό ε, αυτών των ζητημάτων που αναφέρατε. Επίσης να ρωτήσω και εγώ κάτι για τις ε, διατλαντικές σχέσεις ε, γιατί βεβαίως κάποιος ανέφερε πώς θα μπορούσε να είστε η ευρωπαϊκή εκδοχή της ε, Hillary Κλίντον. Εν πάση περιπτώσει, πώς θα έχουμε καλές σχέσεις διατλαντικές και όχι μόνο με την ε, άλλη πλευρά και με τον Ειρηνικό ωκεανό. Τέλος πάντων, ποια είναι τα μαθήματα που έχουμε αντλήσει μετά από την διαμάχη για το βοδινό κρέας με τις ε, ορμόνες και γενικότερα για τις εμπορικές σχέσεις και θα προσπαθήσετε πάντα να έχουμε αρμονικές σχέσεις με τις ΥΠΑ ανεξαρτήτως κόστους. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κύριε Χάουιτ. Ο κύριος Αροσβόλης και έχει το λόγο για ένα λεπτό. Uh, uh, Καταρχά, συγχαρητήρια, Λέδη στον για το διορισμό σα και προσβλέπουμε σε πλήρη πλαγματική και πάει εξωτερική δράση τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω υπό την ηγεσία σα. Έχω δέσεις ερωτήσει. Το πρώτο ερώτημα, πόσο σημαντική για σας είναι το πρόγραμμα για την εταιρική ανατολική σχέση και πώς προτίθεστε να το εφαρμόσετε αυτό το πρόγραμμα και πώς προτίθεστε να εξασφαλίσετε ότι θα εξυπηρετήσει τα συμφέροντα και της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και των ανατολικών γειτόνων μας και κανέναν άλλον. Δεύτερο ερώτημα αφορά τον ασφαλή ενεργειακό εφοδιασμό όσον αφορά τμήμα τη εξωτερική πολιτική. Εδώ το Κοινοβούλιο, πέρα από την ίδια την ενεργειακή πολιτική τη Ενώσεω, θέλει να υπάρχει εξωτερική πολιτική ενεργειακή που θα εφαρμόζεται στα πλαίσια τη εξωτερική πολιτική, στα πλαίσια τη συνθήκη Λισαβόνα. Εσεί πώ προτίθεστε να εξασφαλίσετε ότι αυτό θα, η ενεργειακή πολιτική θα ενταχθεί στην εξωτερική πολιτική τη Ευρωπαϊκή Ενώση, πώ θα εξασφαλίσετε ότι οι αρχέ τη χάρτα ενεργεία θα εφαρμόζονται στην πράξη. Τρίτο ερώτημα. Ευρωπαϊκή Ένωση Ρωσία, πώ προτίθεστε να συνδυάσετε τα ανθρώπινα δικαιώματα εξωτερική πολιτική που βασίζεται στα ανθρώπινα δικαιώματα και οικονομικέ και πολιτικέ πτυχέ και συμφέροντα. Τέταρτον, γεωγραφική ισορροπία και κοινή εξωτερική υπηρεσία, μάλλον εξωτερική υπηρεσία, Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερική Πολιτικής. Παρακαλώ να τηρείτε το χρόνο σας. Ο κ. Γκαλτιέρη, για ένα λεπτό ευχαριστώ. Κυρία Άστον, η ιστορία αυτών των πρώτων δέκα ετών της ΚΕΠΑ σίγουρα είναι ιστορία μιας επιτυχίας επιτυχίας ε, ε, επιχρησιακής των 22 αποστολών, επιτυχία που απορρέει από τη δυνατότητα της ε, ΚΕΠΑ να συντονίζει μέσα πολιτικά και στατιωτικά διαχειρίσεως κρίσεων. Όμως αυτή η επιτυχία επιβάλλει αντιμετώπιση κάποιων προκλήσεων, όχι αυτών της ανάπτυξης και δημιουργίας των σωστών ε, δομών, αλλά διπλής νομιμότητας εσωτερικής της ΚΕΠΑ και της σχέσης με τους εξωτερικούς φορείς και το διεθνές σύστημα. Θα ήθελα να σας ρωτήσω υπό το φως αυτών του σεβασμού που δείχνετε προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, πώς συγκεκριμένα θα δημιουργήσετε τις επαφές, τις σχέσεις με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, σε αυτή την ε, ΚΕΠΑ, κυρίω για τη δρομολόγηση νέων επιχειρήσεων πρώτα απ' όλα. Και δεύτερο, θα σα ρωτήσω, μπορείτε να μα πείτε ποιο είναι το όραμά σα όσον αφορά τι σχέσει μεταξύ ΝΑΤΟ και ΚΕΠΑ και τι είδου συμπληρωματικότητα μπορεί να υπάρχει μεταξύ αυτών. Ευχαριστώ κύριε Γκουαλτιέρη. Η κυρία Άστον έχει μόνο τέσσερα λεπτά για να απαντήσει. Θα είσαστε τόσο γενναία και ικανή να το καταφέρετε. Έχετε το λόγο. Θα προσπαθήσω αλλά να είστε επικείς δεν μπορώ να επισέλθω σε πολλές λεπτομέρειες για τις ε, διατηλαντικές σχέσεις. Έχετε δίκιο, το Διατελετικό Οικονομικό Συμβούλιο και το έργο μου εκεί ε, μου δίνει πλούσια πείρα για το θέμα αυτό και μάλιστα ε, την Παρασκευή συνάντησα την Υπουργό Εξωτερικό Κλίντον ε, και μιλήσαμε και τηλεφωνικά. Θα έχουμε πάρα πολλές συνομιλίες. Θα χαρακτήριζα τις σχέσεις μας ως στρατηγικά σημαντικές. Για πολλά θέματα θα, θα έχουμε την ίδια γραμμή πλεύσης, σε άλλα θα διαφωνούμε, αλλά εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ για τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η Υπουργός Κλίντον για τα συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτειών. Σε ό,τι αφορά τη Μορδαβία, κύριε Πρέντα, η ανατολική εταιρική σχέση θα έχει ουσιώδη σημασία για πολλές εργασίες μας και αυτό θα το συζητήσω και τις επόμενες εβδομάδες με την Μπενίτα Φερόρο Βάλντνερ που θα αναλάβει το χαρτοφυλάκιο του εμπορίου που θα εμπλουτίσει με την πύρα της. Κύριε Σάριος Βόλσκι, το θέμα της ενεργειακής ασφάλειας και του, της ασφάλειας του ενεργειακού ανεφοδιασμού εντάσσεται στο διάλογό μας. Πάντως ε, θα συνεργαστούμε και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που έχει ευθύνες για αυτά τα θέματα αλλά και στο διάλογο και στις διασκέψεις κορυφής. Το θέμα της ασφάλειας του ενεργειακού εφοδιασμού θα είναι παρόν. Στη Στοκχόλμη, στη διάσκεψη κορυφής, ασχοληθήκαμε με όλα αυτά τα θέματα για τη Ρωσία, τα ανθρώπινα δικαιώματα, την ανάγκη διαλόγου με τη Ρωσία, την ενίσχυση και εμβάθυνση αυτής της σχέση ε, για το μέλλον και Πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να ενισχύσουμε αυτό το διάλογο, να τον εντατικοποιήσουμε τους επόμενους μήνες και χρόνια και νομίζω ότι χρειαζόμαστε μια τέτοια ενίσχυση του διαλόγου. Την τελευταία σας ερώτηση δεν την άκουσα γιατί με διάκο... σας διάκοψε ο πρόεδρος, αλλά μπορείτε να μου τη θέσετε κάποια άλλη στιγμή. Ε, σε ό,τι αφορά τα χαρακτηριστικά της ε, σχέσης αυτής, κύριε Γκαλτιέρα, Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό αυτό το θέμα. Ήδη έχει ξεκινήσει μια σειρά συναντήσεων με τους ε, ηθήνοντες ε, και τους επικεφαλείς και στις στρατιωτικές και σε μη στρατιωτικές επιχειρήσεις για να δούμε πώς θα τα δρομοδολογήσουμε όλα αυτά. Και χθες μάλιστα είχαμε σχετική συνάντηση. Θα συμμετέχουμε έχω την Πέμπτη και Παρασκευή σε σχετικές συνομιλίες με τον ΝΑΤΟ και με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ θα ξεκινήσουμε ένα πολύ σημαντικό διάλογο. Σας ευχαριστώ κυρία Άστον. Σεβαστήκατε τέλεια το διάστημα αυτό. Τέταρτη ομάδα ερωτήσεων. Βάιντερ για ένα λεπτό. Ε, Η κυρία after Κυρία Άστον, μετά την εισβολή της Ρωσίας στη Γεωργία τον Αύγουστο του 2008, ε, χιλιάδες ε, Γεωργιανοί 147.000 χρειάστηκε να φύγουν από τη Γεωργία και δεν μπόρεσαν ακόμη να επαναπατριστούν γιατί δεν υπάρχει ασφαλής επιστροφή. Και μάλιστα η κατάσταση όσων έμειναν στα κατεχόμενα της Γεωργίας είναι πολύ κακή. Πώς αντιμετωπίσετε αυτή την κατάσταση που καταστρατηγεί τα ανθρώπινα δικαιώματα. Σε ό,τι αφορά την ενεργειακή πολιτική, χρησιμοποιήθηκε ως εργαλείο της εξωτερικής πολιτικής. Τι σκοπεύετε να κάνετε ώστε τα μεμονωμένα συμφέροντα κάποιων ευρωπαϊκών χωρών να μην έρθουν σε αντίθεση με τα ευρωπαϊκά συμφέροντα για την ενεργειακή ασφάλεια. Υπάρχει πιθανότητα επικάλυψης ε, κάποιων καθηκόντων σας ε, ως Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πώς θα αντιμετωπίσετε τα συγκρόμενα συμφέροντα που σου μερικέ μερικές φορές. Ο κ. Βουάτσον έχει για ένα λεπτό. Παρακαλώ, συνάδελφοι, μόνο ένα ερώτημα. Διότι σε ένα λεπτό, αν κάνετε πάνω από, μία ερώτηση, η κυρία Άστον δεν μπορεί πραγματικά να απαντήσει στο χρόνο που έχει στη διάθεσή σα. Ορίστε. Ε, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Βαρόνι θα μας πείτε κάποια πράγματα για τις στρατηγικές σας προτεραιότητες για την ε, υπηρεσία εξωτερικής δράσης. Θα προωθήσετε τις αξίες της Ευρώπης και αν ναι, πώς θα προωθήσετε την δημοκρατία, το κράτος δικαίου, τα ανθρώπινα δικαιώματα και την κατάργηση της ανατικής ποινής. Δεύτερον, θα πείτε κάτι για το Αφγανιστάν. Συμφωνείτε με τον ε, πρόεδρο Ομπάμα πως ε, κινδυνεύει η ασφάλεια του πλανήτη και αν ναι, τι ρόλο θα παίξει η Ένωση και τα κρατη της. Σας ευχαριστώ κύριε Βάτσον. Για ένα λεπτό, η κυρία Γιαννάκο έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Καλωσορίζω ορίζω ε, την Βαρονέσα Άστον. Ε, επιζητούσαμε πάντοτε μέσω της συνθήκης της Λισαβόνας να έχουμε μια κοινή έκφραση προς τα έξω και αυτό επιτάσσει και η ενιαία νομική προσωπικότητα της Ένωσης. Θέλω να τη ρωτήσω και θέλω να έχω μια απάντηση με ένα ναι ή με ένα όχι. Σκοπεύει να θέσει τα ατομικά και ανθρώπινα δικαιώματα ως προϋπόθεση βασική καλών σχέσεων με οποιαδήποτε χώρα του κόσμου και ιδίως με τις χώρες της Αφρικής με τις οποίες, τις οποίες η Ένωση χρηματοδοτεί. Σας ευχαριστώ κύριε Γιαννάκου. Ράουτσεκ, για ένα λεπτό, κύριος Ράουτσεκ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Βαρώνη Άστον, πρώτα απ' όλα για την Κίνα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ανάγκες για στατική εταιρική σχέση και επικοδομητικές σχέσεις με την Κίνα για διμερή και παγκόσμια θέματα όπω εμπόριο, καταπολέμηση αλλαγή του κλίματο, φτώχεια, μη διάδοση πυρηνικών όπλων κλπ. Αυτό που εξισορροπείται με τη μέρημνα για ανθρώπινα δικαιώματα, τι σχετικέ ανησυχίε και για κάποιε πολιτικέ τη Κίνα σε αναπτυσσόμενε χώρε, όπω την Αφρική. Τι γίνεται με την ισορροπία. Πρώτο ερώτημα. Δεύτερο ερώτημα. Ιράν. Ο πρόεδρος Αχμαντίνε Τζάντ ανακοίνωσε την περασμένη Κυριακή απόφαση να οικοδομήσει άλλε 10 μονάδε εμπλουτισμού ουρανίου. Η απόφαση αυτή ελήφθη αμέσω μετά την απόφαση τη διεθνού υπηρεσία ατομική ενέργεια που καταδίκασε η Ισλαμική Δημοκρατία αυτή. Κατά άποψή σα, τι περαιτέρω βήματα θα πρέπει να λάβουμε ούτω ώστε το Ιράν να συμμορφωθεί με τι υποχρεώσει του και τα ψηφίσματα, τα πολλά του ΟΗΕ, του Συμβουλίου Ασφαλεία. Και τι μπορούμε να κάνουμε και την Ουνία των πολιτών στο Ιράν, για του φοιτητέ, για τι γυναίκε και άλλου. Σα ευχαριστώ. Κυρία Άστον, μπορείτε να απαντήσετε για ένα τετράλεπτο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ ξανά. Όσον αφορά αυτό που κύριε Βεντέιρα, το θέμα της γεωργίας. Νομίζω ότι απαντήσαμε γρήγορα και αποτελεσματικά πέρσι. Θέσατε εντό του ερωτήματό σας και άλλο ευρύτερο θέμα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι αυτό θα είναι ένα κομμάτι των αξιών. Θα συμπεριλαμβάνεται στις αξίες που ανέφερε ο κύριο Βάτσον, που έχουμε στην καρδιά μας. Είναι στον πυρήνα της προσέγγιση που ακολουθούμε ρωτήσατε για τον πρόεδρο εξωτερική πολιτική. Η συνθήκη είναι ξεκάθαρη. Θα λειτουργεί στο δικό του επίπεδο ο πρόεδρο. Οπότε δεν νομίζω ότι θα υπάρξει κάποιο πρόβλημα, διότι πράγματι ήδη με την αναλλακτική προεδρία, αναλασσόμενη προεδρία, ε, λειτουργούμε ως ομάδα, όπου αυτό ενδείκνεται. Θα το ρυθμίσουμε, αλλά σίγουρα θα είμαστε αποτελεσματικοί. Κύριε Βάτσον, ρωτήσατε οι στατικέ προτεραιότητε τη Υπηρεσία Εξωτερική Δράσεω και νομίζω ότι οι αξία είναι στο επίκεντρο αυτών των δράσεων. Αυτό που προσπαθώ να κάνω διότι είχα, επισκέφθηκα και της, ε, με αντιπροσωπείς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όλο τον κόσμο είναι να χρησιμοποιήσω τις ικανότητες τις ηγετικές για να δω ότι είναι μοναδικό που προσθέτει αξία σε αυτά που κάνει τα, κάνουν τα κράτη-μέλη. Να δώσω θέμα τη είναι αξία. Πού δημιουργούνται δυνατότητες να μιλά η Ένωση με μία φωνή, να ηγείται σε συνομιλίες με αυτές τις χώρες, σε συγκεκριμένα θέματα που μας απασχολούν. Τώρα, αν είναι παρόμοια αντιμετώπιση σε κάθε χώρα, αυτό είναι κάτι που μπορούμε να το εξετάσουμε. Αλλά σίγουρα θα είναι μοναδική και διαφορετική αυτή η υπηρεσία. Όσον αφορά το Αφγανιστάν, μελετούμε αυτά που είπε ο πρόεδρο. Εγώ θα ήθελα να εργαστούμε αποτελεσματικά, να συνεργαστούμε στα πλαίσια τη UPOL. Εκεί μπορούμε να δώσουμε προστιθέμενη αξία να δώσουμε στη θέμα θέμενη αξία όσον αφορά την κατάρτιση και υποστήριξη. Αυτό είναι κάτι που αναγνωρίζεται όχι μόνο στο Αφγανιστάν, αλλά ε, και σε άλλα μέρη του κόσμου. Και θα πρέπει αυτό να συνεχιστεί, να είναι αποτελεσματικό. Θα το συζητήσουμε από τα πρώτα θέματα που θα συζητηθούν στι διατλαντικέ σχέσει, θα είναι αυτό. Με ρωτήσατε, ναι. Δεν είναι, η ερώτησή σα δεν απαντάτε με ναι, ναι, όχι, δυστυχώ. Γιατί? Διότι ήμουν υπουργό για τα ανθρώπινα δικαιώματα και νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουμε πού μπορούμε να προσθέσουμε αξία για να πάρουν αυτά τα θέματα στα σοβαρά οι χώρες αυτές μέσω διαλόγου και μέσω της σχέσης που έχουμε και πού είναι καλύτερο να πούμε ότι κοιτάξτε σε κάποιες περιστάσεις η Ευρωπαϊκή Ένωση λέει δεν μπορούμε να έχουμε διάλογο μέχρι να αλλάξετε κάτι. Ποια είναι η άποψή μου. Ότι υπάρχει ένα ολόκληρο φάσμα. Η πρόκληση για εσά σαν Ευρωβουλευτέ είναι να, να με να με ρωτάτε σε αυτό το φάσμα που βρίσκομαι. Άκουσα διάφορε απόψει σχετικά με τι διάφορε αντιμετωπίσει. Εγώ δεν προσπαθήσω να κάνω. Να είμαι ξεκάθαρη απέναντί σα. Γιατί πρέπει να κάνουμε κάτι συγκεκριμένο. Έχουμε συγκεκριμένη ε, θέση και πώ ταιριάζει με την επιθυμία μα να προωθούμε τα ανθρώπινα δικαιώματα. Κύριε Ρούτσεκ, όσον αφορά την Κίνα, ήδη προείδευσα ω επίτροπο Εμπορίου τον ε, διάλογο με την Κίνα συναντήθηκα τη Δευτέρα σύντομα με τον Υπουργό Εμπορίου τη Κίνα, στη Γενέβη ε, είναι πάρα πολύ σημαντική στατική σχέση αυτή που θα πρέπει να έχουμε με την Κίνα, διότι η Κίνα θα πρέπει να βλέπει προς την Ευρωπαϊκή Ένωση όπως και προς τις ΗΠΑ. Εγώ έχω ισχυρές ε, σχέσεις με τον Υπουργό Εμπορίου, τον Υπουργό Εξωτερικών και τον Πρωθυπουργό. Προείδρευσα σε αυτή την ε, πρωτοβουλία μαζί του, οπότε θέλω να το, να το καλλιεργήσω αυτό θα πρέπει να δούμε και τη σχέση αυτή όχι μόνο της Κίνας με την Αφρική αλλά εν γέννη με την Αφρική. Πώς μπορούμε να προωθήσουμε την ανάπτυξη στην Αφρική με κάθε σημασία του όρου. Ιράν, βεβαίω λυπούμε για την απόφαση που έλαβε το Ιράν και θα πρέπει να είμαστε ενωμένοι και νομίζω ότι ήδη υπάρχει αυτή η ενότητα της διεθνούς κοινότητας όσον αφορά τις απόψεις μας για τα επόμενα βήματα έναντι του Ιράν και τα βήματα που κάνει το Ιράν στο τέλος θα πρέπει να βρούμε μια διαπραγματευτική λύση ή δυνατόν, αλλά θα πρέπει να συνεχιστεί και η εξέταση ενδεχομένων κυρώσεων. Σας ευχαριστώ κύριε Άστον. Ξεκινάμε τη, το πέμπτη ομάδα παρεμβάσεων. Βίλερ για ένα λεπτό. Κυρία Βίλερ. Αξιότιμη Άστον. αναφερθήκατε ήδη στο θέμα της πυρηνικής ενέργειας του Ιράν. Σωστό. Να μας πείτε ποια σχέδια έχετε για τις μελλοντικές σχέσεις ε, με την Ευρωπαϊκή Ένωση που είναι πολύ ευρύτερες ε, από αυτό το ζήτημα. Π.χ. η χρήση του μεγάλου δυναμικού της κοινωνίας των πολιτών. Σωστό είναι το ότι υπάρχουν ε, διαπραγματεύσεις, να μην υπάρχει πρόγραμμα πυρηνικών όπλων του Ιράν. Επίσης θετικό είναι να υπάρξει ένας ε, πυρνικός αφοπλισμός και βρίσκεται τώρα επιθύρες ε, η Επιτροπή της Συμφωνίας Μη Διάδοσης Πυρνικών Όπλων και θα ήθελα να ξέρω ποια σχέδια έχετε εσείς για εφαρμογή αυτής της συνθήκης. Ευχαριστώ κύριε Λοχμπίλερ. Το λόγω για ένα λεπτό και ο Σβάν Όρντεν. στον του ότι εκ των υστέρων ε, διοριστήκατε από τον Βρετανό Πρωθυπουργό και τους σοσιαλιστές συνοδοιπόρους του στην Ευρώπη. Όταν αλλάξει η κυβέρνηση στη Μεγάλη Βρετανία θα ζητήσετε μία νέα εντολή. Δεύτερον, είπατε πως είμαστε στο Αφγανιστάν για να γίνουν ασφαλέστεροι οι δρόμοι στην πατρίδα μας. Τι σημαίνει αυτό όταν κάθε μέρα έρχονται στις χώρες μας παράνομα άνθρωποι από το Ιράν, το Αφγανιστάν και από άλλες χώρες όπου εκολάπτεται η τρομοκρατία και όταν λέτε πως υποστηρίζετε την κυβέρνηση και τον λαό της Σρι Λάγκα που χρειάζονται γενικευμένο σύστημα προτιμήσεων για να αναδικοδομηθεί η χώρα μετά από 30 χρόνια. Τι άποψη έχετε. Ευχαριστώ για ένα λεπτό κύριο Σκόβατσεκ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κυρία Άστον πρώτα απ' όλα να σας συγχαρώ για τον διορισμό σας. Εμένα το ερώτημα μου είναι πιο θεσμικό. Πώς σκοπεύετε να συντονίσετε το έργο σας με τους επιτρόπους εκείνους που έχουν πτυχές εξωτερικής πολιτικής όπως π.χ. ανάπτυξη, διεύρυνση, ανθρωπιστική βοήθεια και πώς σκοπεύετε να γίνει αυτό με την μελλοντική υπηρεσία εξωτερικής δράσης. Ε, θα έχετε κάποιο ομάδα εξωτερικής πολιτικής εντός του σώματος ε, των Επιτρόπων. Και η συνεννόηση θα γίνει ευθύς εξ ad hoc ανάλογα με το τι προκύπτει. Ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ κύριε Κόβατσεκ. Για ένα λεπτό Μούνιτς, κυρία Μούνιτς. Ευχαριστώ. Και σας ευχαριστούμε κυρία Άστα. Ως ε, γυναίκα και προοδευτική είμαι ιδιαίτερα χαρούμενη και ικανοποιημένη για το διορισμό σας σε αυτό το αξίωμα. Ε, ο πρόεδρος Ομπάμα παρουσίασε την ε, στρατηγική του για το Αφγανιστάν και Πέμπτη και Παρασκευή θα συνέλθουν οι Υπουργοί Εξωτερικών των Συμμάχων στις Βρυξέλλες. Στις 28 Ιανουαρίου θα γίνει η Παγκόσμια Διάσκεψη για το Αφγανιστάν και γίνεται προσπάθεια συνένεσης ή συντονισμένης θέσης για το Αφγανιστάν. Σε ό,τι αφορά την επιχείρηση Αταλάντη και την ναυτιλιακή ασφάλεια στον ειδικό. Χαιρόμαστε για την επιχείρηση Αταλάντη, αλλά δεν νομίζω ότι είναι μια βιώσιμη λύση. Πώς θα συμβάλλετε σε μια βιώσιμη λύση για την ανάπτυξη της Σομαλίας και την ασφάλεια στη θάλασσα Πώς επίσης θα συντονιστείτε με τους, με τους επιτρόπους για την ανάπτυξη. Στην, ε, φαίνεται ότι χαλαρώνει το ενδιαφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Λατινική Αμερική. Έχετε κάποια, κάποιο συγκεκριμένο σχέδιο για την Λατινική Αμερική. Σας ευχαριστώ κυρία Μούνης. Άλλα τέσσερα λεπτά σε εσά ε, για να απαντήσετε κυρία Άστον. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Λαμπιλίου, με ρωτήσατε για ε, την ε, κοινωνία των πολιτών του Ιράν. Είναι μια σημαντική πτυχή της ε, πολιτικής μας όσον αφορά αυτό το πάζλ των σχέσεων με τις άλλες χώρες που βασίζεται σε διαφορετικές πτυχές και πολιτικές, ενίοτε στρατιωτικές και οπωσδήποτε οικονομικές. Και οι σχέσεις αυτές δεν περνάνε μόνο μέσω εμού αλλά και μέσω των βουλευτών ηγετών, υπουργών εξωτερικών και ενισχύεται έτσι ο διάλογος και συμφωνώ πως αυτό είναι σημαντικό κομμάτι του όσων πρέπει να γίνουν. Όσον αφορά δε την αναθεώρηση της συνθήκης περί μη πυρηνικών δεν έχω αυτή τη στιγμή κάποιες ιδέες για την εφαρμογή. Σημαντικό είναι να συνεχιστούν οι πρωτοβουλίες. Κύριε Φανόρντεν, Χαίρομαι που είπατε πως εκ των υστέρων το σκέφτηκε ο Πρωθυπουργό. βεβαίως δεν ήταν αυτές οι συζητήσεις που είχα εγώ μαζί του. Ο δε ηγέτης σας ήταν ένας από του πρώτου με συνεχάρη. Και χάρηκα για τα συγχαρητήρια αυτά. Δεν νομίζω πως ζητάει την ε, παρέτησή μου. Έχω το μήνυμα στον τηλεφωνητή αν θέλετε να τα ακούσετε. Αλλά χάρηκα που με καλωσόρισε τόσο θερμά και όπως το είπε και ο ίδιος αντιπολίτευση ή όχι ε, θα συνεργαστούμε και βεβαίως ε, να είστε σίγουροι πως όταν ήμουν Βρετανίδα Επίτροπος Εμπορίου ενημέρωνα όλα τα πολιτικά κόμματα και η πόρτα μου και για εσάς όπως και για κάθε βουλευτή όσον αφορά άλλα ζητήματα. Τα μεταναστευτική πολιτική δεν είναι ζήτημα δικό μου για τις γενικευμένες προτιμήσεις ε, να το εξετάσω, αλλά έχει ένα πολύ συγκεκριμένο σκοπό το καθεστώς αυτό και ξεκινάει με κάποιες συγκεκριμένες αξίες, ε, κριτήρια εν πάση περιπτώσει. Και υπό την προηγούμενη μου ιδιότητα φρόντιζα για την εφαρμογή αυτών των κριτηρίων. Οπότε ο διάλογος συνεχίζεται και θα δούμε τι θα γίνει. Κύριε Κόβατσεκ, πώς θα συνεργαστούν οι επίτροποι. Δεν θα τους κατευθύνω, αλλά ελπίζω να έχουμε μια στενή συνεργασία ως Επίτροπος Εμπορίου συνεργαζόμουν με τους Επιτρόπους Ανάπτυξης, Βιομηχανίας για την κλιματική αλλαγή κτλ. Αυτό σκοπεύω να το κάνω. Νομίζω πως ε, όσο περισσότερο συνεργαζόμαστε τόσο περισσότερο επιτύχουμε και το αναμένω αυτό. Δεν θέλω τώρα εγώ να πω πως θα έχουμε κάποια ομάδα εργασίας της Εμένα είναι διοργανική η εργασία μου. Αλλά οπωσδήποτε θα παίξουμε έναν σημαντικό ρόλο εντός της Κομισιόν μόλις ε, ενημερωθούμε. Κύριε Μουνίθ, ευχαριστώ για τα καλά σας ε, λόγια. Η δε συνάντηση του ΝΑΤΟ, του Συμβουλίου, όλα αυτά, το Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων, θα αποτελέσουν ευκαιρίες να συζητήσουμε εντός και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης τα δύσκολα αυτά ζητήματα όσον αφορά το Αφγανιστάν και αυτό το οποίο είπατε για την Αταλάντα όπως είπα είναι πολύ σημαντικό να φροντίσουμε να έχουμε και κάποιες πρωτοβουλίες στην ξηρά για να ε, έχουμε ειρήνη στην Σομαλία. Σε συνεργασία με την Αφρικανική Ένωση. Κεντρική Αφρική, ε, Αμερική δεν την έχουμε ξεχάσει. Περισσότερα σε λίγο. Σας ευχαριστώ κύριε Άστον. Έκτη ομάδα ερωτήσεων. Παρεμβάσεις των Προέδρων των Υποεπιτροπών και των εκπροσώπων των Επιτροπών. Χάουταλα της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για 1,5 λεπτό. Σας ευχαριστώ. ευχαριστώ. Λέιδη Άστον. Έχω την αίσθηση ότι το βιογραφικό σας α, ε, μας α, ε, δίνει καλούς ιονούς για την ε, ισχυρότερη θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως προς τα ανθρώπινα δικαιώματα σε εξωτερικές σχέσεις. Δεν ξέρω όμως πώς η διπλωματία μπορεί να ευνοήσει τα ανθρώπινα δικαιώματα. Γιατί οι προσπιστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων ε, ρισκάρουν την ίδια τους τη ζωή. Στην περίπτωση χωρών όπως η Ρωσία και η Κίνα, πολλές φορές ε, χρειάζεται μία στεντόρια φωνή και όχι μία χαλαρή διπλωματία. Ευχαριστώ. Τώρα, σας ευχαριστώ κυρία Αουτάλα, πρόεδρος της Υποεπιτροπής Αμήνης, Jean. Ο κύριος Ντονζόν. Ευχαριστώ. Κυρία Άστα, καταρχήν συγχαρητήρια για το διορισμό σας στο αξίωμα της ύπατης εκπροσώπου εκ μέρους Επιτροπής, της Υποεπιτροπής Ασφάλειας και Άμυνας θα είστε επικεφαλή τη υπηρεσία εξωτερική ε, δράση, που θα είναι σημαντικό μηχανισμό και εργαλείο για την κοινή εξωτερική πολιτική ασφάλεια και Άμυνα. Και ε, αυτή η δομή, όπω ζήτησε το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο, θα περιλαμβάνει πολλού μηχανισμού ε, διαχείριση κρίσεων, που μέχρι στιγμή ανήκαν σε αρμοδιότητες Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη Γραμματεία του Συμβουλίου, άσχετα αν έχουν στρατιωτικό ή μη στρατιωτικό χαρακτήρα. Ποια είναι η δική σας ε, πρόθεση για το πώς θα διαρθρωθούν οι διάφοροι μηχανισμοί εντός της εξωτερικής υπηρεσίας σε ό,τι αφορά τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνας. Όσοι είπατε εκπρόσωπος θα είστε και επικεφαλής αυτού του οργανισμού που δημιουργήθηκε πριν από πέντε χρόνια για να καλυφθούν οι ανεπάρκειες ως προς τον εξοπλισμό που παρατηρήθηκαν σε διάφορες επιχειρήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ένα από τα προβλήματα που έχει ο οργανισμός αυτός άμυνας είναι η χρηματοδότηση και ο πολιετής προϋπολογισμός του κάποια προβλήματα και κολλήματα οφείλονται στη δική σας πατρίδα. Πώς σας σκοπεύετε να υπερκεράσετε αυτές τις δυσκολίες. Σας ευχαριστώ κύριε Ντανζάν για την Επιτροπή Ανάπτυξης ο κύριος Ντέβα για ένα μισή λεπτό. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Η Βαρόνη Άστον ανέλαβε πολύ δύσκολη δουλειά. Καλή τύχη της εύχομαι. Της... Ε, η Λέδη Άστον ε, τελικά έδειξε μεγάλη αυτοπεποίθηση. Σαν δεύτερο αντιπρόεδρος Επιτροπής Ανάπτυξης, θα σας ρωτήσω, Λέδη Άστον, βλέπετε διάκριση μεταξύ συντονισμού εξωτερικής πολιτικής των κρατών μελών και του ξεχωριστού ε, θέματος ε, ανακούφισης της στόχιας στον κόσμο. Επιβεβαιώνετε ότι το ρόλο σας τον βλέπετε σαν ισότιμο με τον ρόλο με τους υπουργούς εξωτερικών των κρατών μελών και με τον, τον κύριο Πίμπαλτς επίσης που είναι τον, ε, τον Επίτροπο Ανάπτυξης. Ισότιμο ρόλο. Ευχαριστώ κύριε Ντέβα. Για 1,5 λεπτό κυρία Μουσκαρντίνη για την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Βαρώνει Ευχόμεθα ότι εσεί μαζί με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να μπορείτε να μιλάτε, να αντιδράτε, να συζητείτε. Όπω είπατε και εσεί στην παρέμβασή σα, όσον αφορά τι ευθύνε σα για τη διαχείριση των αντιπροσωπιών τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή στι τρίτε χώρε, ε, που αυτέ οι αντιπροσωπείε ασχολούνται βασικά με το εμπόριο. Πιστεύετε ότι μπορείτε να συμφιλιώσετε το, τη διοργάνωση των αντιπροσωπιών εξωτερικού εμπορίου της Ευρωπαϊκής Ενώσεως εν ώψη της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικών Υπηρεσιών και συνεργασία με τις δικές μας πρεσβείες στο εξιστήτες χώρες. Πρέπει να υπάρχουν περισσότεροι υπάλληλοι όχι μόνο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αλλά και του Ευρωπαϊκού Κοινοβούλιου σε αυτές τις πρεσβείες που θα έχουν σημαντικά καθήκοντα. Εμείς θα θέλαμε να έχετε περισσότερο, περισσότερες δυνατότητες ελέγχου, να μπορείτε να ελέγχονται οι εμπορικές δραστηριότητες, οι πρακτικές dumping και να μην περνάνε τα παραποιημένα προϊόντα για να μειωθούν οι διαφορές με τους εξοκοινωτικούς μας εταίρους. Για να γίνει αυτό, πρέπει η πολιτική να εφαρμόζεται και μέσω του εξωτερικού εμπορίου με προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων θύσιο όμως και των δικαιωμάτων του εμπορίου εν γέννη παράλληλα. Ευχαριστώ κυρία Μουσκαρντίνη. 1,5 λεπτό είχε ο καθένας και γι' αυτό σας ε, δίνουμε ένα λεπτό παραπάνω, μερικά δευτερόλεπτα παραπάνω για να μπορέσετε να απαντήσετε. Πέντε λεπτά σας δίνουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ γενναιόδωρος ε, κύριε Πρόεδρε. Ε, ρωτήθηκα καταρχά για το ρόλο τη ήπια διπλωματία και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Προσπάθησα να κάνω τη διάκριση αυτή, όταν χρησιμοποίησα τη φράση αυτή, διάκριση μεταξύ πάντα σαν κάτι, σαν ένας εγωισμός με πόδια να παρουσιάσω σαν εικόνα. Πολλές φορές και στα πλαίσια καθηκόντων μου, στα πλαίσια εμπορίου, ήξερα ότι άμα κάνει κάτι έξω από το φω των προβολέων, ότι πετύχει καλύτερα αποτελέσματα. Αυτό δεν σημαίνει ότι πάντα αυτό ισχύει. Σωστά το θέτε σαν ερώτημα. Και όσοι με είδατε να δουλεύω, υπήρξατε μάρτυρες ότι όταν χρειάζεται θα πρέπει να είμαστε στην πρώτη γραμμή με πολύ χειρή φωνή, στεντόρια φωνή, εκφράζοντας ανησυχίε, ε, προβληματισμό για τα τεχνόμενα στον κόσμο. Και σα διαβεβαιώνω ότι όπω είπατε έχω ιστορικό σε αυτό το τομέα και αυτό θα κάνω. Για τον κύριο Σονζάν τώρα. Δίκιο έχετε. Πρέπει να δούμε μακροπρόθεσμα τι γίνεται. Διότι η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Άμυνα στα πέντε χρόνια που υπάρχει ε, έχει πολλά να κάνει ακόμα. Ήταν επιτυχέστατο φορέα, πέτυχε πολλά αλλά πρέπει να επιδιώξουμε στενότερη συνεργασία με την υπηρεσία διαστήματο, με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κλπ. Και μια από τι φιλοδοξίε μου για τι επόμενε εβδομάδε είναι να μπορέσω να συνομιλήσω με όλου του εμπλεκομένου σε αυτού του δύο φορεί να δούμε ε, πώς μπορούμε να θέσουμε μακροπρόθεσμα στρατηγικούς στόχους και πώς μπορούν να εφαρμοστούν και να πετευχθούν αυτοί. Ε, ο νέος τρόπος λειτουργίας σημαίνει ότι μπορούμε να εξετάσουμε προσεκτικά ποια θέλουμε να είναι το αποτέλεσμα και πώς θα το επιδιώξουμε στρατηγικά. Το έχω υπόψη μου αυτό και έχω υπόψη μου αυτή την υπηρεσία άμυνας και πώς θα κινηθεί. Κύριε Ντέβα, ανάπτυξη το ερώτημά σας αφορά δύο πράγματα. Η ανάπτυξη να μην χάσει τη φωνή της, συμφωνώ με αυτό απόλυτα. Ακόμα και αν συνδυάζουμε τη δράση της Ευρωπαϊκής Ενώσεως στην προσπάθεια ανάπτυξης, εσεί σαν Επιτροπή Ανάπτυξη και όσοι ασχολούνται με την ανάπτυξη πάντα θα μπορούν να βλέπουν, θα πρέπει να βλέπουν το κομμάτι τη ανάπτυξη, να είναι ορατό. Συμφωνούμε, θα το ξεκαθαρίσω όμω πρέπει η ανάπτυξη να εντάσσεται στην ευρύτερη εικόνα των σχεσιών μας με άλλες χώρες. Σαν επίτροπος εμπορίου, το εμπόριο τέριαζε με την ανάπτυξη. Όπως και τα θέματα του κλίματος ταιριάζουν την ανάπτυξη. Όπως και τα θέματα ασφάλειας πάνε παράλληλα με την ανάπτυξη. Αν οι γεωργοί συνέχεια πρέπει να μετακινούνται διότι α, τους κυνηγάει ο πόλεμος, δεν μπορούν να σπείρουν, δεν μπορούν να αναπτύξουν την οικονομία τους. Άρα είναι ένα κομμάτι τη γενικότερη εικόνα, αλλά και κάτι ξεχωριστό, κυρία Μοσκαρντίνη. Θέλω του ικανότερου στην υπηρεσία εξωτερική δράση, του καλύτερου, από όπου και αν έρχονται. Άνθρωποι που πρέπει να προωθήσουν αυτό το ρόλο. Το εμπόριο ήταν πάρα πολύ σημαντικό από τη δική μου εμπορία σε πολλέ αντιπροσωπείε και έχουμε έξοχου ανθρώπου σε όλο τον κόσμο που μπόρεσαν να προωθήσουν το θέμα. Και αυτό θα εξακολουθήσει να αποτελεί κομμάτι των προσπαθειών. Σωστά μου το θέσατε. Και οι βουλευτέ ταξιδεύουν. Και αυτοί μπορούν να μου δώσουν πληροφορίε Πού πετύχαμε περισσότερο, όπως τα βλέπετε εσείς. Πού θεωρείτε ότι χρειάζεται περισσότερη προσπάθεια. Σας ευχαριστώ κύριε Άστον. Έβδομη ομάδα παρεμβάσεων. Πρώτη παρέμβαση, Στράσερ, για ένα λεπτό. Κύριο Στράσερ. Καλώς ήρθατε, Ελένη Άστον, και συγχαρητήρια και καλή επιτυχία. Να επανέλθω τώρα στις σχέσεις ε, με την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, με τις ΗΠΑ και ειδικά την ε, συνεργασία στον τομέα της ασφάλειας. Αυτή είναι αναγκαία όχι μόνο από την 11η Σεπτεμβρίου και μετά, είναι ζήτημα αρχών. Αλλά αυτό το οποίο ανισχύει περισσότερο τους ε, ευρωβουλευτές και τους πολίτες είναι η προστασία προσωπικών δεδομένων και δικαιωμάτων. Και εκεί πέρα έχουμε ανησυχητικές ε, πληροφορίες. Έχουμε τα τέλη των 10 ε, δολαρίων για είσοδο, το πρόγραμμα πληροφοριών αεροπορικών ε, επιβατών κτλ. Θα ήθελα λοιπόν να τοποθετηθείτε σχετικά. Σας ευχαριστώ κύριε Στράσερ. Για ένα λεπτό. Ο Ιουλαντ. Η κυρία Ιουλαντ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Α, Όμεν Ρόιτεν άκουσα, με συγχωρείτε. Έδωσα το λόγο στην κυρία Ιουλάντ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Βαρόνι Άστον, η ερώτησή μου αφορά τη διαμάχη Ρωσίας-Γεωργίας. Εσείς, ως είπατε εκπρόσωπος, τι σκοπεύετε να κάνετε προκειμένου να αποτραπεί επανάληψη αυτής της ε, διένεξης στο μέλλον και στην υπερτριστερία και στον Ακόρνο Καραμπάχ. Τι θα πράξετε προκειμένου να διορθωθεί εκεί η κατάσταση και πώς θα αποφύγουμε περαιτέρω διαμάχες ε, Ρωσίας-Γεωργίας γιατί πέρυσι μιλήσαμε για το τι θα μπορούσε να είχε κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση για να αποφύγει τη διένεξη. Αλλά σας ε, διαβεβαιώ ότι σήμερα η κατάσταση στη Γεωργία εξακολουθεί να είναι πολύ λεπτή και επικίνδυνη. Γιατί δεν δέχτηκε η Ρωσία ε, Ευρωπαίους παρατηρητές στη Νότια Οσετία και Απχαζία. Σας ευχαριστώ κυρία Ογιολάντ. Για ένα λεπτό. Παλέκης. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Άστον. Οι σοσιαλιστές ήταν και είναι υπέρ του αφοπλισμού. Σημερίζεται το όραμα του Αμερικανού Προέδρου Ομπάμα για έναν κόσμο χωρίς πυρηνικά όπλα. Και τι δράση θα μπορούσε να αναλάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση προς αυτή την κατεύθυνση. Ακούγοντας τις απαντήσεις σας, διαμόρφωσα την εντύπωση ότι Όσο πιο ε, δύσκολες είναι οι ερωτήσεις που σας κάνω, τόσο καλύτερα απαντάτε. Έχω μία απλή ερώτηση. Ποια είναι κατά τη γνώμη σας ε, η ικανότητα και η πιθανότητα της Τουρκίας να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέσα σε 10-15 χρόνια. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κύριε Παλέκης. Η κυρία Όμεν Ράιτεν έχει το λόγο για ένα λεπτό. Λοιπόν, τώρα είναι η σειρά μου. Καλώς ήρθατε. Δεύτερον, σε μία από τις ε, απαντήσεις καταλάβαμε πως ήσασταν Βρετανίδα ε, Επίτροπος. Σας επαναλαμβάνω, δεν έχει εθνικότητα Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κατόπιν, όταν ταξιδεύετε ανά τον κόσμο θα ε, εκπροσωπείτε τις ε, κοινέ μας αξίες όπως αναφέρονται στη Χάρτα Θεμελιωδών Δικαιωμάτων στην οποία, την οποία δεν έχει προσυπογράψει το Ηνωμένο Βασίλειο. Πώς θα την υπερασπίσετε λοιπόν. Και στη συνθήκη της Λισαβόνας ε, ζητάμε την υπογραφή της σύμβασης της σχετικής του ΟΗΕ. Πόσο θα επιδιώξεις την υπογραφή αυτή. Σε ευχαριστώ κύριε Αμέν Είπατε εκπρόσωπος έχει το λόγο για τέσσερα λεπτά απαντήσουν. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Στράσερ. Μιλήσατε, ρωτήσατε και πάλι για τις διατελετικές σχέσεις και το θέμα της προστασίας και ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων. Ο Επίτροπος Ζακ Μπαρό ασχολήθηκε με το θέμα αυτά και είναι πιο αρμόδιος. Πάντως ως ε, υπουργό ε, Δικαιοσύνης ε, είχα ασχοληθεί με το θέμα αυτό και από ό,τι θυμάμαι είχαμε πολύ ε, τακτικό διάλογο με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και τότε ήμουν ε, υπουργό όταν ε, η, την Προεδρία την ασκούσε η Μεγάλη Βρετανία. Και φροντίζουμε και στη συλλογή των δεδομένων να αναγνωριστούν τα δικαιώματα των πολιτών. Δεν ξέρω τι τροπή έχουν πάρει οι συζητήσει αυτέ τώρα, γιατί εκπίπτει αυτό το θέμα πια των αρμοδιοτήτων μου. Πάντω είναι πολύ σημαντικό και σα ευχαριστώ που το θέσατε. Κύριε Όγιουλαντ, Ρωσία και Γεωργία. Δεν μπορώ να σας εκθέσω όλες τις λεπτομέρειες ε, για το προς τα που θα πρέπει να οδεύσουμε. Πάντως, ε, θα πρέπει να αναγνωριστούν δύο τινά. Καταρχήν, θα πρέπει να συνεχίσουμε το διάλογο και να έχουμε επίγνωση αυτών των θεμάτων, ακόμη και αν ε, έχουμε ξεπεράσει το θέμα των διενέξεων. Έχουν παραμείνει εκκρέμει κάποια ζητήματα και θα αποτελέσουν τμήμα του στενού διαλόγου που θα έχουμε στο μέλλον. Και θα ήθελα να αποκρισταλωθούν οι απόψει μα στου επόμενου μήνε. Δεν μπορώ τη δεύτερη μέρα τη ανάληψης των καθηκόντων μου και χωρί να έχω προβεί σε κάποιες διαβουλεύσεις ε, ή με προκατόχου ή με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να λάβω θέση για το θέμα αυτό από τώρα. Κύριε Παλέτσκη, για τον κόσμο χωρί ε, πυρηνικά. Ε, μου είπατε ότι προτιμώ τις δύσκολες ερωτήσεις και μια τέτοια μου θέσατε. Σίγουρα ε, ένα κόσμο χωρί πυρηνικά είναι η προσδοκία του κάθε ανθρώπου. Αλλά η, διαδικασία είναι πολύ σύνθετη, περίπλοκη και χρονοβόρα. Ο πρόεδρος Ομπάμα εξέθεσε την αμερικανική θέση για το θέμα αυτό. Με ρωτήσατε και για την Τουρκία. Από ό,τι ξέρω, 33 είναι τα κεφάλαια των διαπραγματεύσεων και μόνο ένα έχει ολοκληρωθεί θα είναι χρονοβόρη διαδικασία και υπάρχει διάσταση απόψεων στο Συμβούλιο και για το θέμα της διεύρυνσης και για το πώς ε, θα προχωρήσουν καλύτερα οι σχέσεις με την Τουρκία. Θα πρέπει να το συζητήσουμε αυτό. Αλλά τόσος χρόνος πέρασε και μόνο ένα κεφάλαιο έκλεισε. Αλλά θα συνεχιστούν οι συζητήσεις για το θέμα αυτό. Και τέλος, κυρία Ομέν Ρόιτεν. Δεν ε, εννοούσα ότι ήμουν επίτροπος της Βρετανίας. Εννοούσα ότι κατάγομαι από τη Βρετανία. Δεν έχω ηθαγένεια. Είμαι Ευρωπαία πάνω απ' όλα και αυτή είναι η σχέση που έχω και με το αξίωμά μου. Είμαι Ευρωπαία και φυσικά έχω και δραστηριότητα στα εθνικά πράγματα και είμαι υπερήφανη γι' αυτό, αλλά είμαι ιδιαίτερα περήφανη που είμαι Ευρωπαία και με αυτό το πρίσμα θα εργαστώ και στο νέο αξίωμα. Και φυσικά Όλα, όλα τα κράτη-μέλη θέλω να συμμετέχουν στη διαδικασία αυτή όσο μπορεί ο καθένα Ευχαριστώ. Για το χάρτη, για το χάρτη. Είπα, θέλω όλα τα κράτη-μέλη να συμμετέχουν στο θέμα αυτό. Είχα συγκεκριμένη ερώτηση για το χάρτη και για την υπογραφή τη συνθήκη τη Γενέβη. Μήπω θα είχα την καλοσύνη να την επαναλάβετε. Ναι, σα υπέβαλα μια συγκεκριμένη ερώτηση. Είπα πώ θα ε, προσπίσετε το χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων και δεύτερον πώς ε, θα προωθήσετε την υπογραφή της Ευρωπαϊκής ε, Σύμβασης για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Μα το ξεκαθάρισα ήδη ότι οι λεπτομέρειες για το πώς θα προχωρήσουμε θα έρθουν αργότερα. Πάντως, ως πρώην υπουργό Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, αλλά και ως πρώην Επιτροπός Εμπορίου, έδωσε ιδιαίτερη σημασία και έμφαση στα ανθρώπινα δικαιώματα. Τώρα, αν επειδή κατάγομαι από τη Βρετανία, δεν έχω διαφορετική άποψη. Έχω το ευρωπαϊκό πρίσμα, γιατί με είπατε εκπρόσωπος Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σας ευχαριστώ, κύριε Άστον. Για ένα λεπτό, Μποτσκούρ. Κυρία Μποτσκούρ. Ευχαριστώ. Συγχαρητήρια, Λέβη Άστον, για τον διορισμό σας. Με ικανοποιεί ως ε, επικεφαλής της ε, αντιπροσωπείας ε, με την ε, Κεντρική Αμερική. Θα ήθελα να σας ρωτήσω πώς θεωρείτε ότι μπορούν να προωθήσουν τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα οι διαπραγματεύσεις για την Ονδούρα. Η κρίση δεν έχει περάσει. Πώς μπορεί η Ευρώπη να παίξει έναν ρόλο πρωτοποριακό σε συνεργασία με τον Οργανισμό Αμερικανικών Κρατών και να φροντίσει να καταλήξουμε σε μια βιώσιμη κατάσταση στην ε, Κεντρική Αμερική. Τέλος, για τη Μέση Ανατολή, υπό το φως της έκθεσης Goldstone, πώς ε, βλέπετε την εφαρμογή των ε, συμπερασμάτων και την παρακολούθηση και τη συνέχεια που πρέπει να δοθεί. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, κύριε Μπότσκουρτ. Για ένα λεπτό, ο κύριος Λαντσμπέργκης. Ευχαριστώ. Αξιότιμη κυρία ενώ στην ε, Ένωση συνεχίζουμε να μιλάμε για την Ευρωπαϊκή Αλληλεγγύη, το σύνθημα αυτό απομακρύνεται όλο και περισσότερο από την πραγματικότητα. Η συμφωνία η ρωσογερμανική κρατικών εταιριών περιαγωγού στη Βαλτική έγινε πίσω από την πλάτη κρατών μελών και θα συνεχιστεί αγνοώντας το σχετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για μια σωστή αξιολόγηση των περιβαλλοντικών απειλών με καμία εγγύηση για τους λαούς μας. Αλλά το χειρότερο είναι ότι βράχει πρόθεσμα θα φρουρείται ο αγωγός από το ρεσικό ναυτικό. Και τα πρώην ουδέτερα ύδατα της Βαλτικής θα γίνουν πλέον γειτονιά του στρατηγικού άρχοντά μας, του Κρεμλίνου. Πρέπει να το αγνοούμε το ζήτημα ή θεωρείτε πως πρέπει να ασχοληθείτε επιτέλους με αυτό. Σας ευχαριστώ. Κάτσιν για ένα λεπτό. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Βαρόνι Άστον, η Βοσνία Ζεγοβίνη έχει δύσκολο πλαίσιο, δύσκολο ιστορικό και αβέβαιο μέλλον. Υπάρχει ύπατος εκπρόσωπος στο Σεράγεβο, αλλά θέλετε να τον απολύσετε. Η Βοσνία Ζεγοβίνη δεν μπορεί να γίνει μέλος της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Η, η Γερμανία που ήταν προτεκ... δεν έγινε τελικά παρόλο που είχε προβλήματα στο παρελθόν δεν έγινε μέλος της Ευρωπαϊκής Ενώσεως η Βοσνία Ζεγοβίνη εξακολουθεί να χρειάζεται εκεί έναν ύπατο εκπρόσωπο μέχρι ότου να γίνει μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι ντόπιοι πολιτικοί περιμένουν να τελειώσει ο χρόνος του ύπατου εκπροσώπου για να κλείσει το γραφείο του ύπατου εκπροσώπου και γι' αυτό οι πολιτικοί δεν θέλουν να επενδύσουν στο μέλλον, στις μελλοντικέ πολιτικές η μία ενωμένης Βοσνίας Αζεγοβίνης. Εγώ προτείνω να ενισχύσετε το ρόλο, τη θητεία μάλλον, να επεκτείνετε τη θητεία του είπα το εκπροσώπου εκεί και έτσι να σταθεροποιηθεί η Βοσνία Ζεγοβίνη, όλη η περιοχή και να προωθηθούν οι ευρωπαϊκές προσπάθειες ε, σε όλη την περιοχή των Δυτικών Βαλκανίων. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο κ. Πέτερινγκ έχει το λόγο για ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Βαρόνι Άστον. Φαίνονται σε σπάν και οι δύο ιδιότητες και τις είπα της εκπροσώπου και τη αντιπροέδρου. Συγχαρητήρια θερμά. Ερωτώ λοιπόν, ποιες είναι οι προτεραιότητές σας για να ενισχυθεί ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον κόσμο. Ε, τι σημασία δίνεται στον διαπολιτισμικό διάλογο και για το ιστορικό πλαίσιο. Πριν από 20 μόλις χρόνια η Σλοβενία ανέκτησε την ανεξαρτησία της. Και όταν ξεκίνησε τις προσπάθειές της, χαρακτηρίστηκε ανίκανη. Μας είπαν τότε ότι δεν επρόκειτο να καταφέρουμε τίποτα. Και αυτά μάλιστα ήταν τα λόγια πεπειραμένων ανθρώπων. Αυτά ως προς το ιστορικό. Ε, τελείωσε λοιπόν η συστάδα των ερωτήσεων, οπότε ήρθε η ώρα να απαντήσετε, λέει Διάστον. Έχετε τέσσερα λεπτά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κυρία Μποσκούρτ, όσον αφορά τις διαπραγματεύσεις ε, με την Κεντρική Αμερική και την χρήση συμφωνιών για την προώθηση περιφερειακής ολοκληρώσης, συμφωνώ μαζί σας. Υπάρχουν πραγματικές δυνατότητες να χρησιμοποιήσουμε τις συμφωνίες αυτές για να υποστηρίξουμε τη σωστή ευρω... Ε, περιφερειακή ολοκλήρωση. Όχι να την επιβάλλουμε, αλλά να δημιουργείται αυτή η ολοκλήρωση που είναι καλή για αυτές τις χώρες. Όσον αφορά τώρα την Ονδούρα, μια κοινοβουλευτική αντιπροσωπεία είναι εκεί ακόμα ή επιστρέφει. Δεν ξέρω ποια είναι η άποψή του. Ε, θα πρέπει να γίνει συζήτηση στο Συμβούλιο την επόμενη εβδομάδα για την Ονδούρα, να δούμε ποια είναι η θέση του. Δεν χρειάζεται να σα εξηγήσω Γνωρίζετε πολύ καλά πώ έχουν τα πράγματα, αλλά θα πρέπει να το συζητήσουμε αρκετά γρήγορα το θέμα. Και όσον αφορά τη Μέση Ανατολή, ήδη ξεκίνησα προσεκτική ανάλυση του θέματος και ανησυχώ πολύ για την ανθρωπιστική κατάσταση εκεί, κυρίως τη λωρίδα της Γάζας και έχουμε προκλήσεις για να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα. Την Παρασκευή το απόγευμα είχα βιντεοδιάσκεψη με τα μέλη του κουαρτέτου που εδρεύουν στην Ιερουσαλήμ για να προσπαθήσω να ξεκινήσω μια συνεργασία μαζί τους για να καθορίσουμε τη θέση μας. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να εξασφαλίσουμε ότι δεν θα κινηθούμε προς τα πίσω, να, προοδεύσουμε. Έχουμε τον οδικό χάρτη, ξέρουμε που πρέπει να φτάσουμε και πρέπει να εξασφαλίσω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα παίξει το ρόλο της. Κύριε Λαντσμπέργκης, είπατε κάτι πολύ σημαντικό, ήταν πολύ ένθερμος ο λόγος σας. Ένα λεπτό δεν μπορώ εγώ να σας δώσω μια οριστική άποψη όσον αφορά ένα θέμα που είναι τόσο ε, καινούριο για μένα. Είμαι ειλικρινής σε αυτό που λέω και ένα θέμα που θα υπάρχουν πολλές απόψεις, όχι μόνο στο Κοινοβούλιο αλλά και εκτός. Αυτό θα σας πω είναι ότι θα πρέπει να καταλάβω τις λεπτομέρειες καλύτερα, να συνεργαστώ με τους συναδέλφους μου που επεξεργάζονται το θέμα και στα κρατημέλη και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ελπίζω ότι εσείς και εγώ θα έχουμε τη δυνατότητα διαλόγου επί του θέματος. Όσον αφορά ε, το θέμα του γραφείου του είπατε εκπροσώπου στη Βοσνία, ε, προτείνατε να ενισχύσουμε την εντολή, να επεκτείνουμε την εντολή. Κύριε Κατσίν, η δουλειά που ο Καλ Μπίλτ έκανε, κυρίως και το θέμα της πρωτοβουλίας 5 συν 2, είναι κάτι που εξεταστεί διεξοδικότατα, να δούμε πώς μπορούμε να προχωρήσουμε από εδώ και πέρα στη Βοσνία. Εγώ έχω κάποιε ανησυχίε όσον αφορά την κατάσταση. Θα έχετε και εσεί τι δικέ σα ανησυχίε. Και ο Καλ Μπίλτ και εγώ ήδη ξεκινήσαμε συζητήσει. Και ξεκινήσαμε συζητήσει και με του Αμερικανού ομολόγου του, προσπαθώντα να δούμε πώ μπορούμε τον καλύτερο δυνατό τρόπο να εξασφαλίσουμε ότι θα επικρατήσει σταθερότητα εκεί. Ξέρω πόσο σημαντικό είναι το θέμα. Αυτό έχω να σα πω. Σα ευχαριστώ. Α, ξέχασα κάτι, λέει κυρία Άστον. Τον κύριο Πίτερ λησμόνησα. Ζητώ συγγνώμη, συγγνώμη. Έχω τόσα χαρτάκια με ονόματα εδώ. Προτεραιότητες για την Ευρωπαϊκή Ένωση και το διαπολιτισμικό διάλογο. Υποθέτω ότι με αυτό εννοείται τη δυνατότητα που έχουμε να συνομιλούμε με όλου όλο τον κόσμο σε διαφορετικά πολιτισμικά πλαίσια με διάφορε ομάδε τη κοινωνία. Αν αυτό εννοείται, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, έχει τεράστια σημασία, είναι ιδιαίτερα σημαντικό ο ρόλο των κοινοβουλίων. Σω να μην κάνουμε αρκετά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κάνει, αλλά πολλά άλλα κοινοβούλια δεν κάνουν αρκετά. Όσον αφορά να προωθήσουμε αυτό το διάλογο, να δημιουργήσουμε το διάλογο, είναι πάρα πολύ σημαντικό να δούμε ότι εδώ μιλάμε για τη σημείο διαπαφής μεταξύ Ευρώπης και των εταίρων μας στην παγκόσμια οικονομία και των εταίρων μας στην αντιμετώπιση πολιτικών δυσκολιών. Αλλά να μπορούμε επίσης όπου χρειάζεται να προωθούμε τις απόψεις μας βάσει των αξιών που μας ενώνουν ως ε, Ευρωπαίους. Σας ευχαριστώ κύριε Άστον. Περνάμε στην ένατη ομάδα ερωτήσεων. Παρέμβαση ενός λεπτού. Κράισελ Ντόρφλερ. Και εγώ θα ήθελα να σας συγχαρώ Βαρονιάστον. Η Βραζιλία βεβαίως δεν έχει σημαντικό ρόλο μόνο στην οικονομία και στο κλίμα αλλά και στην διεθνή πολιτική και διπλωματική σκηνή. Ο πρόεδρος Λούλα δέχτηκε τον πρόεδρο του Ιράν, τον κύριο Αχματινιτζάντ και ακούστηκαν κάποια σχόλια. Θεωρείτε λοιπόν πως η Βραζιλία παίζει ήδη και θα μπορούσε να παίξει σημαντικότερο ρόλο στη Μέση Ανατολή δεδομένων των ε, διπλωματικών αντιπαραθέσεων και με το Ιράν και βλέπετε μια ενίσχυση της ε, υπηρεσίας σας ακριβώς στη Λατινική Αμερική μέσω της εμπλοκής αυτών των ε, χωρών και συμφωνείτε με την άποψή μου πως ο πρόεδρος Λούλα μπορεί να παίξει ένα εξαιρετικό ρόλο ως ένας νέος παγκόσμιος παίκτη στην αντιμετώπιση των προβλημάτων που έχουμε. Ευχαριστούμε κύριε Κράιστερφλερ. Το λόγο τώρα έχει ο κύριος Τούνα Κέλαμ για ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Κυρία, είπατε, είπατε εκπρόσωπα. Η συνθήκη της Λισαβόνας ε, είναι δύο ημερών. Δεν υπάρχουν πια ε, δικαιολογίες για να απέχει κανείς από τις εξωτερικές πολιτικές όπως ε, την πολιτική ασφάλειας ε, και ενέργειας. Πώς θα ξεπεράσετε τον, την επικρατούσα διμέρη, τον διμερή χαρακτήρα στις σχέσεις για να δώσετε ένα πιο κοινοτικό χαρακτήρα σε εξωτερικές σχέσεις. Η κυρία Ογιολάντ μίλησε για τη Γεωργία. Εγώ δεν είμαι ικανοποιημένο με την παρούσα κατάσταση στην Γεωργία, γιατί δεν τηρήθηκαν οι συμφωνίες και οι, Ευρω... εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν μπόρεσαν να εισχωρήσουν στα εδάφη ε, των, ε, των... των οπαδών της απόσχησης. Καλώς, ευχαριστώ. Ο κύριος Μάουρ έχει το λόγο για ένα λεπτό. Κύριε Αντιπρόεδρε Άστον, ο διορισμός σας είναι καρπός μιας λογικής που και ο πρόεδρος Μπαρόζο τη χαρακτήρισε ως κοινοτική. Τα κράτη-μέλη έδειξαν ότι πιστεύουν σε μια ευρωπαϊκή εξωτερική πολιτική. Για να αντιληφθεί κανεί καλύτερα πώ μπορεί να λειτουργήσει μια κοινή εξωτερική πολιτική, σα ερωτώ. Εσεί που είστε η έκφραση μια κυβέρνηση που έστειλε στρατεύματα στο Ιράκ, πώ κρίνετε τι χώρε που δεν έστειλα στρατεύματα εκεί και ποια από τις δύο πολιτικές ε, χαρακτηρίζεται ως ευρωπαϊκή. Δεύτερη ερώτηση. Αναγνωρίζετε ή όχι ως είπατε εκπρόσωπος τον νέο εκλεγέντα πρόεδρο της Ονδούρας. Τρίτη ερώτηση. Στην πατρίδα σας, την τελευταία πενταετία, ε, έγιναν κάποιες ε, πολιτικές δολοφονίες ίσως εξαιτίας ρωσικών μυστικών υπηρεσιών που δημιούργησαν τεράστιες εντάσεις μεταξύ της κυβέρνησής σας και της Μόσχας. Ποια κατά τη γνώμη σας πρέπει να είναι η ευρωπαϊκή προσέγγιση απέναντι στη Ρωσία. Ευχαριστούμε κύριε Μάουρο. Το λόγο τώρα έχει για ένα λεπτό η κυρία Γιακονσάρη. Κυρία Άστον, συγχαρητήρια για το διορισμό σας. Είστε πλέον το δημόσιο πρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είστε και τα μάτια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και ο ρυθμός τηλεφώνου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για πολλούς Ευρωπαίους, για πολλές γυναίκες στην Ευρώπη και για πολλές γυναίκες σε ολόκληρο τον κόσμο, ο διορισμός σας είναι πάρα πολύ σημαντικός. Πώς θα συμβάλλετε στην πρόθεση της θέσης της γυναίκας στον κόσμο. Σε ό,τι αφορά την αρκτική ζώνη, την αρκτική περιοχή, είναι μια πολύ ευάλωτη περιοχή και ανοίγει όλο και περισσότερο, μετατρέπεται σε ένα ελντοράντο πετρελαίου και φυσικού αερίου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση όμως δεν συμμετέχει στο Αρκτικό Συμβούλιο. Πώς ε, σκοπεύετε να προωθήσετε την ευρωπαϊκή πολιτική της ε, Ένωσης στην Αρκτική. Ευχαριστώ, κυρία Γιακονσουάρη. Σβέμπ για ένα λεπτό. Ο κύριο Σβέμπ. Κύριε Αντιπρόεδρε, μιλήσατε για την ήπια διπλωματία και απαντώντας στην κυρία Χαουτάλη είπατε ότι δεν είναι αρκετή ίσως για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Θα ήθελα να αναφέρω το θέμα της Λευκορωσίας. Ποια είναι η γνώμη σας για τις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης Λευκορωσίας, γιατί εκεί η ελευθερία και των πολιτικών κομμάτων και των μέσων μαζικής ενημέρωσης είναι συρρυκνωμένη και πολλοί φυλακίζονται για τις πολιτικές τους ε, απόψεις. Ε, Ποια είναι η γνώμη σα για τη Λευκορωσία στα πλαίσια και τη ανατολική εταιρική σχέση. Έχω και δεύτερη ερώτηση. Ποια είναι η γνώμη σα σε ό,τι αφορά την ρωσική προσφορά ότι είναι πρόθυμη να λάβει μέρος στην ανατολική εταιρική σχέση. Πώ κρίνετε αυτή την προσφορά της Ρωσίας. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Επιτρέψτε μου να πω κάτι εν συντομία. Κάποιες ερωτήσεις ίσως να μην καλύφθηκαν ή σας πολύ περιορισμένοι όσον αφορά την κοινή εξωτερική υπηρεσία. Κάποιοι συνάδελφοι ζήτησαν να μας πείτε ποιε είναι οι προθέσεις σας όσον αφορά τις αρμοδιότητες της υπηρεσίας αυτής. Γεωγραφικές αρμοδιότητες, θεματικές αρμοδιότητες. Θα συμπεριλάβει μετά την πολιτική γειτονία ή όχι. Δεύτερον, πώς προτίθεστε να οργανώσετε την υπηρεσία σας θα είναι, θα είναι εκεί οι εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του Συμβουλίου θα είναι ένα κοινό γραφείο ή θα είναι δύο ξεχωριστά γραφεία. Α σας δώσουμε πέντε λεπτά αυτή τη φορά για να δώσετε απαντήσεις. Έχετε το λόγο. Γενεοδορία, γενεοδορία σας είναι απεριόριστη, Πρόεδρε. Τα καλά νέα είναι πως ε, βεβαίως αυτή είναι η πρώτη μας συνάντηση Οπότε τη δεύτερη μέρα των καθηκόντων μου δεν μπορώ να τα ξέρω όλα, αλλά δεν θέλω και να σπαταλήσω τον, τον χρόνο σας όταν υπάρχουν τόσε πολλέ ερωτήσει, οπότε θα επανέλθουμε σε αυτά τα ζητήματα πολλές φορές ελπίζω. Κράισλερ Ντέρφλερ, με ρωτήσατε για την ε, Βραζιλία και βεβαίω έχω συνεργαστεί και ως υπουργό Εξωτερικών και ως Επίτροπος Εμπορίου και έχετε δίκιο, ο πρόεδρος Λούλα τον συνάντησα πρόσφατα στην ε, Σύνοδο, έχει ένα πολύ σημαντικό ρόλο, αλλά έχουμε και εκλογές ε, και είναι ενδιαφέρον να δούμε τι θα γίνει στην Βραζιλία. Πράγματι έχετε δίκιο για τον πιθανό ρόλο της Βραζιλίας, αλλά μπορεί να έχουμε και αλλαγές που θα επηρεάσουν και το πώς θα παίξουν αυτόν τον ρόλο. Φτάνει να πω πως οπωσδήποτε θα συναντηθώ με τους ομολόγους μου και είναι σημαντικό αυτό. Κύριε Κάλαμ, οι διμερείς σχέσεις ε, των κρατών μελών με τις τρίτες χώρες. Αυτό το οποίο θέλω εγώ να κάνω είναι να οικοδομήσω και να βασιστώ στις σχέσεις των κρατών μελών με τις τρίτες χώρες. Κάποια κράτη-μέλη έχουν ε, διπλωματικές σχέσεις αιώνων ε, που βασίζονται σε ιστορικούς και πολιτισμικούς δεσμούς που αποτελούν για εμάς ε, εφόδιο και όχι πρόβλημα και η υπηρεσία βεβαίως ε, που θα συσταθεί σκοπεύει να προσθέσει αξία, όχι να διαταράξει αυτές τις σχέσεις και υπάρχουν αντιπροσωπείες οποίες έχω ήδη επισκεφτεί και ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είτε στο συντονισμό των κρατών μελών είτε στο να προσφέρει διάφορες υπηρεσίες αναγνωρίζεται και εκτιμάται και θα ήθελα να δω το τι έχουμε αυτή τη στιγμή από πλευράς ε, Συμβουλίου και Κομισιόν, να δω το τι δουλεύει, τι λειτουργεί και να πάρουμε τα καλύτερα στοιχεία. Κάποιοι συνάδελφοι ανέφεραν συγκεκριμένες χώρες, συγκεκριμένα ζητήματα, αναφέρθηκε αρκετές φορές η Γεωργία. Εγώ αυτό το οποίο προσπαθώ να κάνω σήμερα είναι να ακούσω από εσά πού θέλετε να δώσω βάρος και σας ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό γιατί έχω ένα τεράστιο χαρτοφυλάκιο και δουλειά μπροστά μου και πρέπει να δώσω προτεραιότητες κάπου και στο πώς θα χρησιμοποιηθούν οι πόροι και με βοηθήσατε πάρα πολύ. Δεν θα παραστήσω τώρα πως έχω λεπτομερείς απόψεις για τα πάντα γιατί μόλις την προηγούμενη πέμπτη έμαθα πως θα πάρω αυτή τη δουλειά και μια μισή μέρα την έχω και φαντάζεστε πως δεν έχω ακόμα ενημερωθεί οπότε σας ευχαριστώ που μου δίνετε την ευκαιρία να ακούσω από σας το τι έχει σημασία όσον αφορά τώρα το Ιράκ κύριε Μάριο Μάρου και την ε, στρατηγική των διαφόρων χωρών ε, και όχι μόνο τις δικές μου έχει σημασία ο ρόλος των κρατών μελών και η στρατηγική προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πάντα θα διαφέρουν τα κράτη-μέλη, διαφέρουν ιστορικά, πολιτικά λοιπά Και οι πολιτικές διαφορές αντικατοπτρίζονται και σε όλους εσάς. Αυτό το οποίο πρέπει εγώ να κάνω είναι να καταλήξω σε μια στρατηγική κοινή συνισταμένη των σημείων που μας ενώνουν. Δεν σημαίνει αυτό πως συμφωνούμε πάντα. Η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων εδώ πέρα θα παίξει ουσιαστικό ρόλο στο να με κατευθύνει αλλά και να μου δώσει κάποια ευκαιρία να παίξω ένα ηγετικό ρόλο. Αλλά αυτό νομίζω θα παραμείνει δηλαδή πιο τα κράτη-μέλη θεωρούν και θα εξακολουθήσουν να θεωρούν πως είναι κράτη μεμονωμένα εντός μιας ένωσης. Και όπως είπα αυτό δεν είναι αρνητικό. Συγκεκριμένα τώρα για το τι συμβαίνει με τη Ρωσία, ο συνάδελφός μου, κύριος David Miliband, ε, θα εξηγήσει τη θέση του Ηνωμένου Βασιλείου, δεν είναι δική μου δουλειά. Κύριε Κινσάρη, σας ευχαριστώ. Τώρα για τις γυναίκες μπορούμε να μιλάμε όλη μέρα, είναι πολύ σημαντικό Συγγνώμη, αναγνωρίζετε ή όχι το νέο εκλεγμένο πρόεδρο τη Ονδούρα. Σα ρώτησα υπό την ιδιότητά σα, αν είπατε εκπρόσωπο, το νέο εκλεγμένο πρόεδρο τη Ονδούρα. Το αναγνωρίζετε. Από χτε η Ευρωπαϊκή Ένωση, στον αριθμό τηλεφώνου, τον οποίο ανέφερε ο Κίσιγκερ, έχει το δικό σα αριθμό τηλεφώνου Βαρόνι. Um, Δεν το ανέφερα γιατί Μόλι το συζήτησα και σα είπα από Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων θα το δει την ερχόμενη εβδομάδα και θα προκύψει θέση. Ε, συγγνώμη αν δεν με ακούσατε. Νόμιζα πω είχα ήδη απαντήσει. Τώρα για να επανέλθω στον ρόλο των γυναικών υπάρχουν πολλά πράγματα να πούμε. Δεν είναι τώρα η στιγμή. Απλά να πω πως είμαι υπερήφανη που κατέλαβα αυτή τη θέση και είμαι γυναίκα σε αυτή τη θέση. Και αυτό αντικατοπτρίζεται στο ποια είμαι και στο τι θα κάνω. Για την Αρκτική πάλι ενδιαφέρον αυτό το οποίο λέτε γιατί δεν είναι κάτι το οποίο είχα την ευκαιρία να σκεφτώ αν έχω την ευκαιρία θα το κάνω θα γίνει άλλος ένας διάλογος τέλος με ρωτήσατε για την οργάνωση της υπηρεσίας εξωτερικής δράσης πρώτα απ' όλα θα υπάρχει μια ενιαία υπηρεσία Συμβουλίου και Κομισιόν το δε γραφείο μου θα είναι στο κτίριο της Κομισιόν για δύο απλούς λόγους. Πρώτον, ξέρω που είναι η καφετέρια και ξέρω πώς λειτουργεί το κτίριο, οπότε δεν χρειάζεται να σκεφτώ τις λεπτομέρειες κτλ. Επίσης, και κάτι σημαντικότερο, ε, μου δίνει τη μεγαλύτερη ευκαιρία το να μην είμαι στο ε, κτίριο, γιατί θα είναι εκεί πέρα ο αντιπρόεδρος της Κομισιόν, οπότε εγώ θα μπορώ να μην είμαι εκεί, να είμαι στο κτίριο του Συμβουλίου και ως είπατε εκπρόσωπος να ασχολούμαι με ζητήματα εκτός Βρυξελών. Ε, Κύριε Πρόεδρε, με ρωτήσατε και εσείς ένα ερώτημα για γεωγραφικά και θεματικά ζητήματα. Εγώ δεν πήρα απόφαση. Αυτό που θα είναι σημαντικό, όπως προσπάθησα να περιγράψω, είναι να δούμε που υπάρχουν ισχυρές αντιπροσωπείες ήδη, επιτυχείς αντιπροσωπείες. Να δούμε τι τις κάνει επιτυχής δημιουργώντα ένα νέο οργανισμό, είναι να πάρουμε τα καλύτερα από αυτά που λειτουργούν και να προσθέσουμε τα στατικά τα κατάλληλα, τα οποία μα δίνουν μια, ένα νέο οργανισμό που αντικατοπτρίζει τα ευκταία. Τα στοιχεία ποια θα είναι. Να βασιστούμε στην ήδη σαν δουλειά. Να συναθρήσουμε τα διάφορα στοιχεία. Όπως είπε και η κυρία Μοσκαρντίνη, να εξετάσουμε θέματα όπως είναι το εμπόριο, ανάπτυξη και ούτω καθεξής. Και να δούμε ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος να έχουμε αποτελεσματικότερη συνεργασία. Αυτό θα κάνω. Αυτή θα είναι η πρώτη μου προτεραιότητα. Θα τον αλλάγω προσωπικά ίδια. Συνεργαζόμενοι με συναδέλφους, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε και σε διάλογο με το Κοινοβούλιο. Σας ευχαριστώ κύριε Άστον. Έχουμε τον τελικό γύρο, τελευταίο γύρο. Ξεκινάμε 1,5 λεπτό προς τον κύριο Προβέρα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Συγχαρητήρια Βαρώνη. Άστον, καλή δουλειά. Ένα θέμα το οποίο με ενδιαφέρει ως ιδιαίτερος, η πολιτική συνεργασία με τις αναπτυσσόμενες χώρες είναι θεμελιώδους σημασίας για τον έλεγχο των μεταναστευτικών ροών. Η μετανάστευση και η παράνομη μετανάστευση δεν μπορεί να περιοριστεί ή να προγραμματιστεί μόνο με αστυνόμευση ή με σοβαρούς νόμους. Χρειάζεται να δημιουργηθούν οι οικονομικές, κοινωνικές συνθήκες και συνήθειες δημοκρατίας για την ανάπτυξη των φτωχότερων χωρών για τις οποίες χώρες η μετανάστευση θα πρέπει να γίνει μία επιλογή και όχι ε, μια αναγκαία λύση για να ξεφύγουν οι άνθρωποι από την πείνα και τη φτώχεια. Θα πρέπει όμως η συνεργασία στον τομέα να είναι ε, αποτελεσματική με καλή χρηματοδότηση και καλή διακυβέρνηση για να φτάνουν τελικά οι χρηματοδοτήσεις σε εκείνους που έχουν ανάγκη για την ανάπτυξη. Χρειάζεται συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση να υπάρχουν οι σωστές ε, υποδομές για τα διάφορα προγράμματα, λιγότερη γραφειοκρατία, καταπολέμηση της διαφθοράς, μετανα, ε, κατάρτιση των μεταναστευτών, μεταναστών ε, και καταπολέμηση των, ε, της μετανάστευσης. Είναι θέμα διαπραγματεύσεων εξωτερικής πολιτικής. Είναι πολύ σημαντικό θέμα. Ως ύπατη εκπρόσωπος, τι σκοπό έχετε να κάνετε, τι σκοπεύετε να κάνετε όσον αφορά αυτά τα θέματα. Ευχαριστώ κύριε Προβέρα. Ξέχασα να πω ότι πέρα από το ότι είσαστε βουλευτή, είσαστε και πρώτος αντιπρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων. Ο κύριος Αγκουράκης για 1,5 λεπτό έχει το λόγο. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, θα ήθελα να θέσω δύο ερωτήματα στην ε, Βαρονέσα την Άστον. Το πρώτο είναι το εξής ζήτημα. Ε, πώς σκοπεύει να αντιδράσει στο γεγονός ότι όλο και περισσότερο κατά τη γνώμη μου υπάρχει παραβίαση του, διεθνού διεθνούς δικαίου και συχνά βρισκόμαστε στο να εφαρμόζεται μια πολιτική φεακομπλή. ενώ Εννοώ και τον πόλεμο στον Αφγανιστάν, ενώ και τον πόλεμο στο Ιράκ, ενώ και το θέμα του Κωσόβου. Και επειδή το ζήτημα του διεθνούς δικαίου είναι πάρα πολύ σημαντικό και στις σχέσεις με την Τουρκία και στην επίλυση του Κυπριακού, νομίζω ότι πρέπει να έχουμε μια συγκεκριμένη απάντηση στο ζήτημα αυτό. Και ένα δεύτερο ζήτημα που έχει σχέση με το παραπάνω είναι το θέμα τη άρση, τη απαράδεκτης κοινή θέση τη Ευρωπαϊκή Ένωση με την Κούβα, η οποία ισχύει σήμερα παρά το γεγονό ότι στον ΟΗ, όπω άριστα θα γνωρίζει η κυρία Άστον, όλες οι χώρε έχουν καταδικάσει το εμπάργο των ΗΠΑ σε βάρο τη Κούβα, όμω η Ευρωπαϊκή Ένωση με την κοινή θέση ε, τηρεί μια, ένα άτυπο καθεστώ εμπάργο προ τη χώρα αυτή. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ κύριε Αγκουράκη. Για ένα, λεπτό. Κόουαλ. Ενάμιση λεπτό. Κόουαλ. Κύριος Κόουαλ. Ευχαριστώ και συγχαρητήρια. Καλή τύχη σας εύχομαι στη νέα σας αποστολή. Θα σκεφτήκατε ποτέ ε, πώς θα έμοιαζε σήμερα η Ευρώπη αν, είχαν κερδίσει, αν είχε κερδίσει το ειρηνευτικό κίνημα στην οποία, στο οποίο συμμετείχατε όταν ήσταν νεότεροι. Σκεφτήκατε ποτέ πώς ήταν σήμερα η Ευρώπη αν είχε επικρατήσει εκείνο το κίνημα. Επίσης ε, δεν απαντήσατε για τον αγωγό. Το Nord Stream είναι πολύ σημαντικό σχέδιο για ολόκληρη την Ευρώπη. Μπορείτε να μας δώσετε μια ημερομηνία πότε μπορούμε να μιλήσουμε συγκεκριμένα για αυτό το θέμα, πότε θα μας δώσετε συγκεκριμένες απαντήσεις. Επίσης, το σχέδιο Σαρκοζή για το τέλος της διένεξης Ρωσίας-Γεωργίας υλοποιήθηκε τελικά ή όχι. Θα συμμετέχετε στη διάσκεψη κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης Ουκρανίας και πρόκειται να τροποποιηθεί η υπάρχουσα πρακτική με τη συνθήκη της Λισαβόνας και να επιτρέψει σε εκπροσώπους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να συμμετέχουν σε τέτοιες διασκέψεις κορυφής είτε με τη Ρωσία είτε με την Ουκρανία. Θα ήταν μια πολύ καλή χειρονομία εκ μέρους σας. Μπορούμε να περιμένουμε κάτι τέτοιο από εσά. Και αν σε τόσες σημαντικές απαντήσεις δεν δίνετε συγκεκριμένες ερωτήσεις ε, δημιουργείται μια ανησυχία. Γιατί πολλές, πολύ συχνά είπατε ότι ακόμη δεν γνωρίζετε, δεν έχετε ενημερωθεί. Ξέρω ότι είναι η δεύτερη σας μέρα. Αλλά πότε μπορούμε στην Επιτροπή Εξωτερικών να σας έχουμε με μια πολύ πιο συγκεκριμένη θέση και γνωστές τις απόψεις για διάφορα θέματα που ρωτάμε. Σας ευχαριστούμε κύριε Κοβάλ. Μπραντνερ, για 1,5 λεπτό τώρα έχει σειρά. Η κυρία Μπραντνερ. Αξιότιμη κυρία Άστον, αποστολή σας είναι τώρα να οικοδομήσετε την Ευρωπαϊκή Εξωτερική Υπηρεσία. Δεν έχετε εμπειρία κλασικής εθνικής διπλωματίας, αν και απαντήσατε αρκετά διπλωματικά. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει διπλωματική παράδοση. Αυτό μπορεί να θεωρηθεί είτε εμπόδιο είτε ευκαιρία. Εμείς το θεωρούμε ευκαιρία γιατί πρέπει να απομακρυνθούμε από τις εθνικές διπλωματικές παραδόσεις του 19ου αιώνα και να ιδρύσουμε μια ευρωπαϊκή παράδοση του 21ου αιώνα, να μην σκεφτόμαστε σε κουτάκια, να έχουμε ενιαίες ε, αντιμετωπίσεις, να εμπλέξουμε την κοινωνία των πολιτών, να έχουμε σύγχρονη διαχείριση των συγκρούσεων και να έχουμε πρωτοβουλίες οικοδόμησης της ειρήνης. Και σοκαρίστηκα είπατε πολλές φορές πως θα προσθέσει προσθέμενη αξία για τα κράτη-μέλη. Όχι, πρέπει να προσθέσει προσθέμενη αξία για τους πολίτες η νέα υπηρεσία. Θα ήθελα λοιπόν να σας παρακαλέσω να τοποθετηθείτε ξανά για αυτό το ζήτημα. Επίσης το ότι προετοιμάζετε φάκελο για τον Ιανουάριο όπως το έκανε και ο κύριος ε, Μπαρόζο, αναμένουμε κάτι τέτοιο, να καταθέσετε το πρόγραμμά σας δηλαδή και βλέπουμε εδώ πέρα χτες ανακοίνωση πως ε, αναμένεται συνεργασία με Κομισιόν, Συμβούλιο και κράτη-μέλη και ξεχάσετε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Τραγική έκπληξη. Ε, παρόλα αυτά χαιρόμαστε και βεβαίως έχετε μπροστά σας να αντιμετωπίσετε ακόμα πολλά. Σας ευχαριστώ. Λάμστορφ για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε Βαρονιάστον. Οι φιλελεύθεροι σας ε, καλωσορίζουν και όπως είπαμε ταυτόχρονα ήσασταν και μέλος της πρώτης Επιτροπής ε, Μπαρόσο επί συνθήκης ε, Νίκαιας και αυτή τη στιγμή ήσασταν ε, μέχρι χτες μάλλον ήσασταν σε ένα ομιχλώδες νομικό τοπίο αλλά τώρα πρέπει να κινηθούμε στο νέο πλαίσιο κάτι το οποίο βεβαίως δεν προδικάζει καθόλου το τι θα γίνει στις ακροάσεις ε, του Ιανουαρίου, αλλά νομίζω μέχρι στιγμής η πορεία σας υπόσχεται πολλά. Επίσης ε, δεν έχουμε ακόμα συγκεκριμένο οργανόγραμμα της νέας υπηρεσίας. Δεν περιμένουμε και σήμερα τέτοια πράγματα, ούτε προπολογισμό. Αλλά τον Ιανουάριο οπωσδήποτε περιμένουμε συγκεκριμένες απαντήσεις. Μην περιμένετε τον Απρίλιο να μας πείτε πώς θα έχει η δομή της νέας υπηρεσίας. Εδώ πέρα τον Ιανουάριο πρέπει να είστε έτοιμοι συγκεκριμένο ερώτημα για την νομική πτυχή. Κατά την άποψή σας έχετε ένα αξίωμα με δύο διαφορετικές μεθόδους εργασίας ή καταλαμβάνετε δύο διαφορετικά αξιώματα. Θέλω μια σαφή απάντηση. Κατόπιν, τι θεωρείτε για το ότι θέλει ο κύριος Μπαρόσο να προσθέσει στην διεύρυνση και την πολιτική γειτονίας και θέλω να ακούσω την άποψή σας και τέλος τι άποψη έχετε για το να ενωθούν οι έδρες που έχουν τα κράτη-μέλη Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Σας ευχαριστώ. Το λόγο για 1,5 λεπτό ο κ. Βόμποντα. Ευχαριστώ. Πολλές ε, ερωτήσεις ήταν περισσότερο μηνύματα Σωστό είναι αυτό όμω και εγώ έτσι θα συνεχίσω. Για τη Ρωσία, να το επαναλάβω, αναμένουμε πιο ρεαλιστική πολιτική αλλά και αυστηρότητα για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία και επί τη ευκαιρία. Nord Stream είναι έργο προτεραιότητα τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Οπότε μπορείτε να ασκείτε κριτική, αλλά είναι έργο προτεραιότητα. Το έχει αποφασίσει η Ένωση. Δεύτερον, για τι ΗΠΑ χρειαζόμαστε ισχυρή συμμαχία, αλλά από μια ευρωπαϊκή θέση και όσο πιο φίλοι είμαστε τόσο πιο πολύ κριτική μπορούμε να ασκήσουμε κατόπιν για τον πυρηνικό αφοπλισμό. Εμείς χαιρόμαστε και πρέπει να συνεχίσετε έτσι ακόμα και αν πρέπει να είστε τώρα κάπως πιο διπλωματικοί αλλά είναι πολύ σωστό αυτό. Για τα ανθρώπινα δικαιώματα βεβαίως πρέπει να συνδυάσετε και τα ανθρώπινα δικαιώματα με την εξωτερική πολιτική και τώρα για τη συνεργασία με το Κοινοβούλιο αναμένουμε περισσότερη συνεργασία από αυτή η οποία είναι απολύτως απαραίτητη από τη θεσμική πτυχή και τώρα κύριε Βαρόνι βρίσκεστε ενώπιον μας αλλά στο μέλλον πρέπει να αποφασίσετε θα καθίσετε στην πλευρά του Συμβουλίου της Κομισιόν εμείς θέλουμε να καθίσετε στην πλευρά της Κομισιόν χωρίς να ξεχνάτε το Συμβούλιο για εμάς είστε γιατί πρόεδρος της Κομισιόν με ε, ευθύνες έναντι του Κοινοβουλίου. Οπότε, αν μπορείτε να πάτε να καθίσετε εκεί πέρα, θα ήταν πολύ θετικό. Σας ευχαριστώ, κύριε Σβόμποντα. Για 1,5 λεπτό, ο κύριος Μπρόκ έχει το λόγο. Äh, κύριε Πρόεδρε, κυρία Αντιπρόεδρε, έχετε ένα χαρτοφυλάκιο νέο για εσάς και ταυτόχρονα ένα νέο αξίωμα. Μιλάμε για τιτάνια καθήκοντα που έχετε να αντιμετωπίσετε. Τις ε, τελευταίες μέρες χάρηκα όταν άκουσα πως ε, το γραφείο σας θα βρίσκεται στην Κομισιόν. Αλλά τώρα βασικά ακούω πως το κάνετε γιατί ξέρετε που είναι η καφετέρια και ο πρόεδρος και κατά βάση θα δράσετε εκτός. Γνωρίζετε πως μεγάλα τμήματα της δουλειάς σας προέρχονται από την κοινοτική πολιτική που ήταν μέχρι τώρα δουλειά της Κομισιόν. Είναι κατεξοχήν κοινοτική και όχι διακυβερνητική υπόθεση η δουλειά σας ευθύς εξ αρχής. Και γι' αυτό και επιπλέον, πέρα από αυτό, δεν είναι μόνο ε, η συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που απαιτείται, το οποίο ξεχάσατε βεβαίω να ανακοίνωση τύπου, αλλά ήρθατε εδώ πέρα σήμερα, αλλά υπάρχει και η λογοδοσία που είναι υποχρέωσή σας έναντι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ως αντιπρόεδρος ε, της ε, Κομισιόν. Και τέλος αυτό το οποίο είπε η κυρία Μπραντνερ η εξωτερική υπηρεσία είναι προσθέμενη αξία για την κοινότητα και τα θεσμικά όργανα της κοινότητας και όχι για τα κράτη-μέλη. Και αν μιλήσετε με την ε, Κορεπέρ ε, πριν ε, από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο νομίζω πως έχει υπάρξει κάποια παρεξήγηση. Και ελπίζω να μπορέσουμε να τα ξεκαθαρίσουμε όλα αυτά τον Ιανουάριο για να μην έχουμε και παρεξηγήσεις στη συνεργασία μας. Ευχαριστώ. Τηρήσαμε τέλεια το ωράριό μας. Εγώ με γεωνοδορία σας εκχωρώ τα δύο λεπτά μου και σας αφήνω και τα οκτώ λεπτά. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Αντιπρόεδρε, κύριε Αντιπρόεδρε, κάνατε μια άκρως ενδιαφέρουσα ανάλυση σχετικά με τα ζητήματα που δημιουργούν τις περιστάσεις που οδηγούν στην παράνομη μετανάστευση. Και ότι σε πολλά που κάνουμε, όπως αναφέρεται και στην επιχείρηση Αταλάντα, πρέπει να καλύπτουμε αυτή την πτυχή στην εξωτερική πολιτική να προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε όχι μόνο τα συμπτώματα του προβλήματος αλλά και τα αίτια. Είναι ένας πολύ καλός τρόπος αυτός όπως το βλέπω διότι κατά την άποψή μου πρέπει να συναθρήσουμε τις προσπάθειές μας ούτω ώστε να είμαστε αποτελεσματικότεροι στην πρόθεση των αξιών μας, δηλαδή δημοκρατία και ανθρώπινα δικαιώματα. Έτσι θα μπορούν οι άνθρωποι να ζουν ειρηνικά, να αναπτύξουν την οικονομία τους, να στέλνουν τα παιδιά στο σχολείο και να μπορούν να γίνουν αυτό που θέλουν. Αυτό είναι το πλαίσιο που θα διέπει την προσέγγιση μου και μου δίνει τη δυνατότητα αυτή η ανάλυση σας. Να πω αυτά που είπα. Αξιοπρέπεια, ανθρώπινα δικαιώματα, αξίες. Επ' αυτών πρέπει να εδράζονται οι προσπάθειές μας. Αυτό δεν σημαίνει ότι τα πράγματα είναι εύκολα. Ότι αυτά μπορούν να μεταφραστούν εύκολα σε συνιστώσεις των σχέσεών μας, διότι αυτά είναι πάρα πολύ περιπλοκά. Απέφυγα να απαντήσω όχι λόγω ελήψεως απόψεων, αλλά διότι θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό να έχω περιστατωμένη άποψη που θα εκφράζω και όχι να είναι απλώ μια αντίδραση. Μία μέρα μολι είμαι εδώ και μερικε ωρε σε αυτή τη θέση. Και όσο και έξυπνη αν θεωρώ ότι είμαι ε, όταν διαβάζω μία ενημέρωση, είναι ε, πιστεύω ότι πρέπει να μπορώ να σα πω αυτό που σκέφτομαι. Χρειάζομαι τι καλύτερε πληροφορίε. Πρέπει να μιλήσω με του ανθρώπου για να δημορφώσω άποψη. Για να σα δώσω άμεσε, απευθεία απαντήσει και αυτό θα κάνω. παραβίαση του διεθνούς δικαίου. Με ρωτήσατε κάτι, δεν ξέρω αν κατάλαβα καλά, για την Κούβα. Ο Επίτροπος Ντεχούπτ έλεγε πρόσφατα ότι προχωρούν τα πράγματα. Και στην Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να δούμε τι σημαίνει αυτό. Εξού και το δεύτερο σημείο μου. Σπάνια είναι στατικές οι καταστάσεις στον κόσμο. Σπανίως είναι απλές οι απαντήσεις ε, που μπορούν να απαντηθούν με ένα ναι ή ένα όχι. Όταν βλέπουμε όσα συμβαίνουν στον κόσμο, είναι σημαντικό θεσμικά να υπάρχει επαφή με το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Κοινοβούλιο για να γίνεται ο σωστός προβληματισμός επί των αλλαγών. Οι αλλαγέ που είναι συνέπειε των όσων έγιναν στην Ονδούρα, οι δηλώσει του Προέδρου Ομπάμα για το Αφγανιστάν, όλα αυτά τέλο πάντων δημιουργούν μια κατάσταση που πρέπει να εξετάζεται, να τη συζητάμε και να καταλήγουμε σε θέση. Καμιά φορά χρειάζεται να γίνονται γρήγορα αυτά. Αλλά πάντα πρέπει να έχουμε υπόψη μας ποιος είναι ο στόχος. Κύριε Σκοέλιο, με ρώτησε αν θα είμαι σύνοδο κορυφή Ευρωπαϊκή Ενώση Ουκρανία. Δεν θα είμαι εκεί. Η Μπενίτο Φεραίρο η κυρία Μπενίτο Φεραίρο Βάλνερ θα εκπροσωπεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Διότι παράλληλα εκείνη την ημέρα θα έχω τη δυνατότητα να είμαι και στο ΝΑΤΟ και συναντήσω τον Υπουργό Εξωτερικών, τον είπα, ε, την κυρία Κλίντον. Και επειδή είναι τόσο ικανή η κυρία Βάλτνερ, επειδή υπήρχε αλληλεπικάλυψη, μπορούσε να μα εκπροσωπήσει εκείνη στην ε, Σύνοδο Κορυφή και εγώ θα είχα την ευκαιρία έτσι να συναντήσω την Υπουργό Εξωτερικών, την κυρία Κλίντον και το Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ. Θα συνεργαστούμε όμω. Πολλά μπορούν να γίνουν όσον αφορά τι σχέσει με τη Ρωσία, και να δούμε και ποιε είναι οι συνέπειε των όσων πρότεινε ο πρόεδρο Σαρκοζή πέρσι και να δούμε πώ να αναπτύξουμε τη σχέση μα προ Ανατολά με όλε τι χώρε. Δυτικά Βαλκάνια. Τι κάνουμε την Ανατολική ε, σχέση γειτονία. Το έχω υπόψη με αυτό. Όταν ήρθα σήμερα, ήθελα καταρχά να σα ακούσω. Δεν είναι η ακρόαση είμαι αυτή. Στην ακρόασή μου θα έχω πιο εμπεριστατωμένε απόψει για διαμόρφωση πολιτική. Εδώ ήταν η πρώτη δυνατότητα που είχα και χαίρομαι γι' αυτό το όπω τον πρώτο τη Επιτροπή. Ήθελα πράγματι το ταχύτερο δυνατόν, τόσο γρήγορα να έρθω. Όχι γιατί θεωρούσα ότι μπορώ να απαντήσω τα πάντα, διότι είχα, ήθελα να έχω τη δυνατότητα να κάνω δύο πράγματα. Πρώτα απ' όλα να σα ακούσω, να σα δώσω ό,τι απάντηση θα μπορούσα να σα δώσω. Και δεύτερον, να σα γνωστοποιήσω το πόσο σημαντικό θεωρώ το Κοινοβούλιο και πόσο μεγάλη αξία έχει ο διάλογο. Ε, που δεν είναι τελευταία μου παρουσία εδώ. Θα συναντιόμαστε συχνά, όσο πιο συχνά μπορώ. Είναι μία από τι προκλήσει που έχω μπροστά μου. Δηλαδή, πώ να ετοιμάσω το χρονοδιάγραμμά μου για πέντε χρόνια δουλειά. Υπάρχουν πολλά πολλά αντικρουόμενα συμφέροντα. Άρα είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει δυνατότητα επαφή μα. Όσον αφορά τη διπλωματική παράδοση, κυρία Βάντνον και προστιθέμενη αξία τη πολίτε. Έχετε δίκιο, είναι προστιθέμενη αξία τη πολίτε. Εγώ θεωρώ τα κράτη-μέλη σαν χώρες με πολίτες, αλλά καλό είναι να χρησιμοποιώ τις λέξεις πολίτες. Έπρεπε συνέχεια να λέω πολίτες και όχι κράτη-μέλη. Όπως είπατε πρέπει να βρούμε μια νέα παράδοση και είναι νέα πιθανότητα, δυνατότητα που έχουμε η κοινωνία των πολιτών και μάλλον να κάνουμε φρέσκα πράγματα. Αλλά φτάνω σε ένα από τα τελευταία που ήθελα να πω. Αυτό είναι εντελώ καινούριο αυτό που γίνεται. Εγώ δεν έχω γραφείο. Δεν έχω υπαλλήλου του γραφείου μου. Έχω μια ομάδα κληρονόμησα ένα κομμάτι άσπρο χαρτί. Και εκεί έγραψα ένα-δύο πράγματα. Ετοίμασα ένα-δύο συναντήσεις. Δεν λειτουργώ από ένα γραφείο επιτρόπου. Συνεργάζομαι με συναδέλφους που με βοηθούσαν πριν, που εκείνοι προσπαθούν να συνεχίσουν με το πρόγραμμα για το εμπόριο ε, τον ελεύθερο χρόνο τους Και προσπαθώ να γνωρίσω καινούριου ανθρώπους απέναντι στο Συμβούλιο. Ε, μίλησα με τον Γενικό Γραμματέα χθε και με άλλους. Δεν έχω τίποτα. Τον εαυτό μου έχω. Με κάποιες μικρές προσθήκες. Το επεξεργαζόμαστε. Δεν είναι δικαιολογία αυτή. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Προσπαθούμε να βγάλουμε άκρη. Τι σημαίνει συνθήκη. Ε, τι κονδύλι χρειαζόμαστε. Ποιε είναι οι σχέσει με την αναλασσόμενη Προεδρία. Όλα αυτά τα πράγματα είναι ολοκένουργια. Δεν θα σε εκπλήσει το ότι δεν μπορώ να σα δώσω συγκεκριμένη απάντηση. Και ίσως να είναι και πλεονέκτημα αυτό. Επειδή δεν περίμενα ε, εδώ να είναι η μίση, μα θέλετε, εγώ ήρθα εδώ με ένα άσπρο χαρτί και περίμενα τη βοήθειά σας για να σημειώσω κάποια πράγματα. Ο κύριος Λάμστορφ. Ήθελε συγκεκριμένε απαντήσει τον Ιανουάριο, βεβαίω. Άλλη εμπειρία του Ιανουαρίου. σω να μοιάζει κάπω με αυτήν, αλλά τότε θα έχουμε περισσότερε δυνατότητε να διαρευνήσουμε πού έφτασα, πού πήγα και όχι τώρα που είμαι στην αρχή. Θα έρθω να μιλήσω και όπω σα είπα, και εκείνοι που συνεργάστηκαν παλιά μαζί μου οι βουλευτέ θα ξέρουν ότι πάντα προσπαθώ να συνομιλήσω μαζί σα, κύριε Σβόμποντα, Αναφερθήκατε σε κάποιες βασικές σχέσεις με Ρωσία, Ηνωμένα Πολιτείε, πολύ σημαντικές σχέσεις, ρεαλισμό, είναι σημαντικό στοιχείο. Πού θα κάθομαι. Ε, ήρθα και κάθισα εδώ, ε, ήξερα ότι όπου και να καθόμουν θα είχα πρόβλημα. Μακάρι υπήρχε και τρίτη θέση. Προσπάθησα να μετακινηθώ μεταξύ των δύο. Τέλο πάντων, δώστε μου κάποια συμβουλή. Δεν έχει σημασία που θα κάθομαι. Πώ με βλέπετε εσεί, πώ με βλέπετε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, πώ με βλέπει το Συμβούλιο, έχει σημασία. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Και προτίθεμαι να κάνω αυτή την ιστορία τη μεγαλύτερη δυνατή επιτυχία. Ελέγξτε με. Όσο θέλετε. Δικαίωμά σα είναι. Αυτό είναι η δημοκρατία. Είναι μία από τι αξίε τη δημοκρατία. Συνεργαστείτε μαζί μου. Βοηθήστε με να τα κάνω σωστά. Για το επόμενο χρονικό διάστημα είναι μεγάλη δουλειά, δεν αισθάνομαι ότι απειλούμε. Προσπαθώ να δημιουργήσω κάτι για το οποίο θα είμαστε όλοι υπερήφανοι και θα πιστεύουμε ότι έχει εκπληρώσει όλα αυτά που απέρευσαν από έτη συζητήσεων, σύνταγμα, συνθήκη και όλα αυτά. Διάβασα τη συνθήκη επί ώρες. Ε, μάλλον πέρασα ώρες για να περάσω τη συνθήκη από το κοινοβούλιο μου. Αυτά δεν θα είναι εις αν ο ρόλος αυτός είναι επιτυχής. Χρειάζομαι βοήθεια όμως και προσβλέπω σε αυτή τη βοήθειά σας στο μέλλον. Σας ευχαριστώ κυρία Άστον. Όπως είπατε, αυτή είναι η πρώτη συνάντηση. Θα υπάρξουν και άλλες συναντήσεις, κυρίως μια επίσημη συνάντηση τον Ιανουάριο και τότε μπορούμε να συνεχίσουμε και να εξετάσουμε τυχόν κενά που διαπιστώνονται. Πάρα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είστε επανειδήν. Καλή δουλειά. Κλείνει η συνεδρίαση για την ώρα. Σε πέντε λεπτά περίπου θα έχουμε το διευρυμένο Προεδρείο στην ίδια αίθουσα. Συνεδρίαση του διευρυμένου Προεδρείου.